Κυρίσω την επανάληψη των εργασιών της Συνόδου της Ολομέλειας που διεκόπη στις 17 Ιανουαρίου 2019. Πρόεδρε Γκράβλοκ, ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μα. Ε, Εξοχότητε, ε, ε, ξέρετε, προσκεκλημένοι μα, πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνοδρίου, κύριε Πρωθυπουργέ, εκπρόσωποι της Ρουμανικής Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι, σήμερα εορτάζουμε μια μέρα μνήμης την μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος. Οι κοινότητες των Εβραίων, οι οθνοτικές μειονότητες όπως η Ρωμά και η Σύντη, όσοι θεωρούνται ανεπιθύμητοι και θεωρήθηκαν ανεπιθύμητοι από το ναζιστικό καθεστώς. Για πρώτη φορά η μέρα μνήμης ε, λαμβάνει χώρα ως τελετή στην, ε, ε, στο εμικύκλιο, στην αίθουσα του εμικυκλίου του Κοινοβουλίου στη Σύνοδο της Ολομέλειας. Με αυτή τη χειρονομία αποστέλουμε ένα ισχυρό μήνυμα περισσότερο από ποτέ. Εμείς δεν ξεχνούμε, δεν ξεχνούμε και δεν θέλουμε να λησμονήσουμε. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη και να καταπολεμήσουμε αόκνος κάθε μορφή μίσους και διακριτικής μεταχείρισης ή αντισημιτισμού. Θέλουμε να παραμείνει ζωντανή η μνήμη των ανίποτων εγκλημάτων του ολοκαυτώματος. Δεν είναι όμως απλώς μία ε, ε, τελετή αυτό. Είναι μια κίνηση για το συλλογικό μας ασυνείδητο, για τη συλλογική μας, τη συλλογική μας μνήμη. Πρέπει να παραμείνει ένα γεγονός που ποτέ δεν θα ξεχαστεί το όλο καύτωμα. Αυτές τις πράξεις βίας και φιλετικού μίσους δεν πρέπει να τις λησμονήσουμε ποτέ. Βάσει των δεδομένων του τελευταίου Ευρωβαρομέτρου, το 50% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι ο αντισημιτισμός είναι ένα πρόβλημα που αφορά την ίδια του τη χώρα. Αυτό καταδεικνύει ότι ο ιός του αντισημιτισμού δεν έχει ακόμη εκριζωθεί. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε με πυγμή και να αντιμετωπίσουμε ε, να ξεριζώσουμε κάθε σπέρμα μίσους που έχει απομείνει. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη ανεκτικότητας και την βία. Η Ευρώπη έχει ήδη αποδείξει επανειλημμένως ότι μπορεί να το κάνει. Το Ευρωκοινοβούλιο υπήρξε και πάντοτε θα βρίσκεται στο πλευρό όσων είναι θύματα πράξεων μίσου και διακριτική μεταχείρισης. Το 2016 διοργανώσαμε μια σύσκεψη υψηλού επίπεδου για το μέλλον των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το 2017 εγκρίναμε το πρώτο μας ψήφισμα κατά του αντισημιτισμού. Μαζί από κοινού θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προασπιστούμε τις αρχές του ε, ψηφίσματος του ΟΗΕ που όρισε μέρα μνήμης τη σημερινή. Θα πρέπει να προωθήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, να ε, καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε άρνηση του ολοκαυτώματος και να καταδικάσουμε χωρίς ε, αμφιβολία κάθε δείγμα διακριτικής μεταχείρισης λόγω εθνοτικής ή θρησκευτικής διαφοράς. Θα πρέπει ε, να υπάρξει ο σχετικός διάλογος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει χώρος για μίσος και αντισημιτισμό. Δεν θα επιτρέψουμε τα τραγικά σφάλματα του παρελθόντος να επαναληφθούν ποτέ ξανά. Θέλουμε να ακούσουμε την μαρτυρία του Προέδρου Κόρτλοκ... ο οποίος είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Μονάχου. Η Σαρλότ Κόρτπλοκ ήταν μόνο τριών όταν της απαγόρεψαν να παίζει με τα άλλα παιδιά στη γειτονιά της. Ήταν Εβραία και αυτό ήταν το μόνο της αμάρτημα. Επέζησε όμως από τις φρικαλαιότητες του ολοκαυτώματος χάρη σε μια γυναίκα, μια χριστιανή που δούλευε στην οικογένειά της. Η Σαρλότ Γκλόμποκ ε, αφιέρωσε τη ζωή της στην καταπολέμηση του μίσους και του αντισημιτισμού. Σε εκείνην απευθύνουμε όλοι μας την ευγνωμοσύνη. Σας ε, προσκαλώ να έρθετε στο Προεδρείο και να λάβετε το λόγο ενώπιον της Συνόδου Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου. Αξιότιμε Πρόεδρε κύριε Ταγιάννη, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας, τα νευναστικά σας ε, λόγια και τα θαυμαστά σας λόγια. Αξιότιμε Πρόεδρε Γιούνκερ, εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Μισελ, ε, αγαπητοί παρόντες μαθητές, ε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την πρόσκληση την οποία δέχτηνε με μεγάλη ευχαρίστηση. Διότι για μένα μια επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάντα κάτι το ξεχωριστό. Θέλω να σας πω κάτι ως προσκεκλημένοι σε εσά που συνηθίζετε να εργάζεστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πραγματικά ε, ένα ξεχωριστό συνέστημα. Μας δίνει ανάταση ε, το κοινοβούλιο αυτό διαφέρει από όλα τα άλλα. Βέβαια, όλοι σας έχετε εκλεγεί από τη χώρα σας και από το κόμμα σας. Έχετε έρθει εδώ για να κάνετε στη δημοκρατική αρένα πολιτική και να προετοιμάσετε και να διαμορφώσετε ένα καλό μέλλον για τους πολίτες της Ευρώπης. Αλλά δεν σταματούν εδώ όλα αυτά πίσω από το Προεδρείο και τούτο εδώ το βήμα δεν βλέπετε μία σημαία αλλά 28 και στη μέση έχουμε την ευρωπαϊκή σημαία που συμβολίζει την ιδέα της ενότητας της Ευρώπης. Μία ιδέα στην οποία έχετε υποχρεωθεί να είστε προσιλωμένοι εδώ και το Κοινοβούλιο δεν νομοθετεί μόνο αλλά δημιουργεί και μια κοινότητα. Εδώ βασίζεται η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στην ελευθερία, στη δημοκρατία, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο ανοιχτό πνεύμα, στην ανεκτικότητα και ε, την επιθυμία για μια ειρηνική συμβίωση. Αυτά σήμερα είναι αυτονόητα στην Ευρώπη και καθορίζουν την καθημερινότητα, αλλά για μας αυτό δεν ήταν καθόλου προφανές και αυτονόητο και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου εδώ. Όταν ήμουν μικρή έζησα στο πετσί μου πολύ άγρια τη βαρβαρότητα που δεν ήθελε πια να αναγνωρίσει τίποτα ανθρώπινο και χωρίς ενδιασμούς εξολόθρευε και θανάτωνε. Τότε έχασα σχεδόν τα πάντα, πολλούς από τους αγαπημένους μου, το σπίτι μου και την ε, αρχική μου ε, εμπιστοσύνη και πίστη στον κόσμο και στους ανθρώπους. Για πάνω από μία φορά η ζωή μου σώθηκε από τύχη. Ε, πολλές χρόνια ζούσα σε μια κρυψώνα με ένα ψευδόνυμο και μια ψευδή ταυτότητα. Γιατί αν ήμουν ο εαυτό μου αυτό θα σήμαινε σίγουρα τη θανατική μου καταδίκη. Σήμερα μπορώ να βρίσκομαι εδώ ενώπιόν σας γιατί ε, ε, μεταξύ όλων αυτών των πολλών δολοφόνων, συνοδοιπόρων και παρομοίων υπήρχαν και άνθρωποι που ρηψοκινδύνευσαν την ίδια τους τη ζωή για να διατηρήσουν την ανθρωπιά τους. Βρίσκομαι εδώ ενώπιόν σας διότι το φως της ανθρωπιάς δεν έσβησε ποτέ εντελώς, ακόμα και στις πιο σκοτεινές εποχές της ανθρώπινης ιστορίας. Αλλά και εδώ είχα καταλάβει από την αρχή. Με πρώτη ευκαιρία θα έπρεπε να φύγουμε, άνδρας μου και εγώ, από την Ευρώπη. Γιατί ε, θεωρούσαμε εκείνη την Ήπειρο διεφθαρμένη και παντού, οπουδήποτε θα ξεκινούσαμε μια νέα ζωή παρά εδώ στη συνέχεια γεννήθηκαν τα παιδιά μας και συνεχώς αναβάλαμε την αποδημία μας. Και τα παιδιά μας γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε μια χώρα ε, όπου η αβεβαιότητα και η δυσφορία ε, ήταν ε, τα κυρίαρχα συναισθήματα για Κίνα και για όλη την εβραϊκή κοινότητα. Τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο είχαμε μια αβεβαιότητα. Δεν ξέραμε ε, ε, ποιον έπρεπε να συναναστραφούμε που να μην ήταν Εβραίο, γιατί δεν ξέραμε ποιο είχε τα χέρια του αιματοβαμμένα με εβραϊκό αίμα. Και ζούσαμε σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη χώρα ε, να παραμείνουμε στη Γερμανία ε, στο για μας ήταν κάτι το αδιανόητο. Το γεγονός ότι σήμερα βρίσκομαι εδώ ενώπιόν σας είναι ίδια η απόδειξη ότι ευτυχώς κατά τη διάρκεια των δεκαετιών άλλαξαν πολλά και έγιναν πολλά δυνατά τα οποία στο παρελθόν θα θεωρούσαμε αδιανόητα. Ποιο θα είχε άραγε τότε σκεφτεί, υπολογίσει ότι η δημοκρατία μετά τον πόλεμο ε, ε, θα ήταν τόσο ισχυρή. Ποιο θα πίστευε τότε ότι στην Ευρώπη ε, μέσα σε λίγα χρόνια θα μπορούσαν να ξεπεραστούν εχθρότητες αιώνων ολόκληρων. Και ποιος θα το πίστευε ότι μετά από τις φρικαλαιότητες του ολοκαυτώματος τις αδιανόητες και πάλι θα μπορούσε να ζήσει ένας Εβραίος στην Ευρώπη. Όλα αυτά σήμερα φαίνονται προφανή. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, δεν είναι καθόλου προφανή. Και τα επιτεύγματα και οι κατακτήσεις δεν είναι πάντα τόσο σταθερά όπως μπορεί να φαίνονται εκ πρώτης όψεως. Και δυστυχώς αυτές τις μέρες αυτό γίνεται πιο σαφές. Η ελεύθερη και δημοκρατική τάξη στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο σήμερα απειλείται περισσότερο από ποτέ. Και εγώ δεν μιλώ για εξωτερικές απειλές ε, σχετικά με τη δική μας συνοχή. Η ευρωπαϊκή ιδέα, το ευρωπαϊκό δεν θα μπορούσε να τις αντιμετωπίσει αυτές τις εξωτερικές. Αυτό που με ανισχύει περισσότερο είναι η έσωθεν ε, επιθέσεις. Ενωμένη στην πολυμορφία μπορεί να είναι η Ευρώπη και στο μέλλον μόνο ε, εφόσον ξέρει ποιες είναι οι αξίες της και τις θεωρεί σημαντικές για να τις υπερασπίζεται με αυτοπεποίθηση. Αυτό το μέλλον όμως αναγκαστικά συνδέεται με τη γνώση για το παρελθόν. Στις 27 Ιανουαρίου, ε, στην Παγκόσμια ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, θυμηθήκαμε τα 6 εκατομμύρια Εβραίων, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από το 1933 μέχρι το 1945 από την ναζιστική Γερμανία. Η απελευθέρωση του ε, στρατοπέδου συγκέντρωσης Auschwitz στις 27 Ιανουαρίου ε, έγινε πριν από 74 χρόνια όλο και λιγότεροι είναι οι επιζώντες που μπορούν να μιλήσουν από το πρώτο χέρι και να πούν ε, πόσα φρικτά έζησαν εκεί. Γι' αυτό και είναι πιο σημαντικό ε, και περισσότερο σημαντικό το μήνυμα των επικεφαλής των ψηφοδελτίων ε, των χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών για τις επόμενες ευρωεκλογές. Ήταν μαζί ο Μάνφρετ Βέμπερ και ο Φραντ Τίμερμανς στο Auschwitz. Παρ' όλα αυτά παραμένει ένα θλιβερό γεγονός. Όλο και περισσότερο χάνονται αυτές οι φωνές, σβήνουν. Θα έχουμε σε λίγο ένα διάστημα και ένα χρόνο χωρίς αυτόπτες μάρτυρες. και ορισμένοι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται πια να θυμόμαστε ε, αυτά τα πράγματα, το ολοκαύτωμα. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο λανθασμένο. Παντού βλέπουμε στην Ευρώπη πολιτικά κινήματα να κερδίζουν και δύναμη, τα οποία αποφασισμένα ε, αντιστέκονται στη μνήμη ε, και στις Ε, Προπαγανδίζουν ένα παρόν χωρί παρελθόν ω ένα εφαλτήριο σε ένα μέλλον χωρί μνήμη. Ε, έτσι, με τέτοια λύθη της ιστορίας σηκώνει κεφάλι ο αντισημιτισμός και δυστυχώς αυτό δεν είναι απορίας άξιο. Ε, εμείς, τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας, ήδη από σήμερα ζούμε αυτές τις επιπτώσεις και στη Γερμανία και σε πολλά άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να είσαι Εβραίος και να έχεις δημόσια ζωή απαιτεί ε, αστυνομική προστασία και Εβραίοι όλο και περισσότερο αισθάνονται ανασφαλείς. Βέβαια γυρίσανε ε, στο κέντρο των πόλων και συναγωγές χτίζονται και σπίτια ε, και αιστείες κοινοτικέ. Είναι μια νέα μορφή συνύπαρξης. Τα κτίρια αυτά βασίζονται στα θεμέλια της εμπιστοσύνης. Και εγώ μπορώ να σας πω από πρώτο χέρι πόσο χρειάστηκε μέχρι να ε, αισθανθώ ξανά το, μετά το 1945 ε, πόλη μου το Μόναχο που έχω γεννηθεί και είναι η πατρίδα μου. Πραγματικά ε, άδειασα τις βαλίτσες μου με την, τα γένεια της συναγωγής καινούρια στο Νοέμβριο του 2006, οριστικά. Και σήμερα καταλαβαίνω ότι μήπως βιάστηκα να αδειάσω αυτές τις βαλίτσες. Σε ε, πολλές περιπτώσεις αμφιβάλλει ε, ο Εβραίος για το μέλλον του. Ε, οι Εβραίοι πίστευαν ότι ε, ποτέ δεν θα αισθανθούν στη χώρα τους τέτοια πίεση. Είναι πολλές οι επιθέσεις και λεκτικές, αλλά ακόμα περισσότερη η αδιαφορία, η έλλειψη κατανόησης, η έλλειψη ενσυναίσθησης. Γιατί όπου και να γυρίσουμε τη ματιά μας, σηκώνει το άσχημο κεφάλι του ο αντισημιτισμός σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλο το πολιτικό φάσμα. Δεν είναι μόνο οι ακραίοι, είναι και το κέντρο και πολλοί ε, ε μουσουλμάνοι. Η AFD, οι BDS και ακραίοι ε, Ισλαμιστές έχουν κοινά, λίγα κοινά, αλλά στον αντισημιτισμό έχουν κάτι που τους ενώνει όλους αξιότιμοι παρόντες. Βέβαια όλα αυτά είναι η μισή αλήθεια και μόνο. Ευτυχώς παντού στην Ευρώπη υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται για τη μνήμη και τη δημοκρατία και την ε, ανοιχτή σκέψη. Οι φωνές τους είναι πολλές, είναι ηχηρές. Σε πολλά, αν όχι σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, συνιστούν την ευρεία πλειονότητα του πληθυσμού. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε λόγω αυτής της αριθμητικής υπεροχής. Η ε, ιστορία έχει αποδείξει πόσο δύσκολο ε, μπορεί να είναι το έργο της ε, πλειονότητας όταν θέλει να υπερασπιστεί τα ιδανικά της σε μια επίμονη μειοψηφία απέναντι. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα στην ευρωπαϊκή πολιτική, πόσο γρήγορα διαδίδεται ο αντισημιτισμός εάν δεν μπουν κάποια όρια εγκαίρως. Ένα από τα πιο δραστικά παραδείγματα αυτής της εξέλιξης ε, διεξάγεται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Εργατικό Κόμμα που κατά τη μακρά της ιστορία ήταν ένα προπύργιο ε, λογικής, της πολιτικής, με την προεδρία του Τζέρεμι Κόρμπιν τα τελευταία χρόνια ε, έγινε από τα πια κατάφορα προβληματικά κόμματα στην Ευρώπη ε, σε ό,τι αφορά τον πολιτικό αντισημιτισμό. Με τη νέα ηγεσία ε, το εργατικό κόμμα άφησε πίσω του και πολύ μακριά το πολιτικό κέντρο. Είναι προφανές ότι στο ηθικό ημίφος το να μην παίρνει θέση βοηθάει να αναπτυχθούν τα πιο άγρια ζυζάνια της πολιτικής. Πόσο γρήγορα φεύγουμε από την πολιτική της ανοχής και της ανεκτικότητας όταν είναι ευνοϊκά τα σημεία των καιρών. Παράδειγμα λοιπόν είναι το εργατικό κόμμα υπό τον Κόρμπιν και τέτοιες εξελίξεις δεν αφορούν μόνο ε, τον ιδιαίτερο ρόλο του Μεγάλου ε, Ηνωμένου Βασιλείου συγγνώμη, φαίνονται παντού στην Ευρώπη. Κάτι έχει ολιστήσει, κάτι έχει αλλάξει. Ο αντισημιτισμό σε πολλές χώρες της Ευρώπης βρίσκει χώρο και πολιτικό και κοινωνικό ξανά. Ε, αυτό που και πολύ καιρό έρχεται στην επιφάνεια και όπου ο αντισημιτισμός δεν πατάσεται ενεργά και αμέσως ανοίγει δρόμους και το είδαμε πρόσφατα, το είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι παρόντες. Θα ήθελα να είμαι απολύτως ξεκάθαρη. Σε μια Ευρώπη όπου πάνω από το 89% του εβραϊκού πληθυσμού ε, διαμαρτύρεται για την αύξηση του αντισημιτισμού στη χώρα του, ε, είναι προβληματική αυτή η Ευρώπη. Μια Ευρώπη που πάνω από το 1 τρίτο των Εβραίων έχουν σκεφτεί σοβαρά να αποδημήσουν. Έχει πρόβλημα ο αντισημιτισμός δηλητηριάζει γενικά το κλίμα στην κοινωνία. Ελευθερία και ασφάλεια ισχύουν για κάθε πολίτη της Ευρώπης ή για κανέναν. Ο αντισημιτισμός τα περιφρονεί αυτά. Με γεμίζει πόνο και λύπη τόσα πολλά χρόνια μετά το τέλος του ολοκαυτώματος σήμερα να έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο πολύ δεδομένο αντισημιτισμό. Αλλά χρέο όλων μας θα πρέπει να είναι να αντιταχτούμε και να αντισταθούμε σε αυτή την εξέλιξη και να την κάνουμε να υποχωρήσει. Αυτό είναι το δικό μας καθήκον. Διότι η μεγαλύτερη τραγωδία ε, της εβραϊκής ιστορίας έγινε εδώ στην Ευρώπη. Η πόλη που είναι σήμερα το κέντρο της ζωής μας πριν από 80 χρόνια και λιγότερα ήταν τα θέατρα ε, ε, του χειρότερου εγκλήματος στην ιστορία της ανθρωπότητας και τα προκάλεσε η τότε γερμανική κυβέρνηση. Αξιότιμοι παρόντες, αξιότιμοι επίτροποι, αξιότιμοι βουλευτές. Εσείς είστε εκείνοι που ορίζετε τις μοίρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γι' αυτό απευθύνω έκκληση σε εσά και σήμερα και στο μέλλον και μετά τις ε, ερχόμενες ευρωεκλογές να αντισταθείτε ε, στεναρά σε αυτόν τον αντισημιτισμό. Επιθυμώ τούτο το κοινοβούλιο και στο μέλλον να εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στο χρέος που έχει και στην ευθύνη του. Η ελευθερία και η δημοκρατία που απολαμβάνουμε σήμερα είναι πάντα μόνο τόσο ισχυρή όσο ισχυρή είναι η δέσμευση της δημοκρατίας και των δημοκρατών. Και θα πρέπει η πλειονότητα να αντισταθεί στη μειονότητα δεν μπορούμε να αφήσουμε να κερδίσει αυτό το μίσος. Όχι πια, όχι ξανά. Από το, όχι, το ποτέ πια δεν επιτρέπεται να γίνει και τώρα ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε για για την τόσο πολύτιμη κατάθεσή σας που για μας έχει ανεκτιμητή αξία. Τώρα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην μνήμη όλων των θυμάτων του ολοκαυτώματος και έχουμε κατά το ότι ένα λεπτό για κάθε θύμα θα σήμαινε ότι θα πρέπει να κάτσουμε για πέραν από 11 έτη στην ε, σιωπή. Κατόπιν. Κατά, αυτή, κατά αυτό το λεπτό θα έχουμε προβολή κάποιων σχεδίων ε, παιδικών. Ήταν 15.000 και σώθηκαν 150 και μας ε, άφησαν αυτές τις ε, εντυπώσεις, αυτά τα παιδιά που χάθηκαν με τις εντυπώσεις τους, επομένως και πρόκειται, αυτά έχουν έρθει από την συναγωγή της ε, Πράγας. Εκεί αποτυπώνονται τα συναισθήματά τους ενώπιον αυτών των φρικαλαιοτήτων που κανένα παιδί δεν θα πρέπει πια να υποστεί. Ποτέ πια.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 seduta è e sospesa Διακόπτεται η συνοδός για 5 λεπτά. Presidente. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσω να μιλώ για κάτι το οποίο μα θλίβει πάρα πολύ. Πρόκειται για τη Βενεζουέλα, όπω γνωρίζετε την περασμένη εβδομάδα, με την ευκαιρία αυτών των μαζικών συλλαλητηρίων κατά του καθεστώτο, ο πρόεδρο τη Εθνοσυνέλευση, Χουάν Γουάιντο, ανακηρύχθηκε πρόεδρο προσωρινό ε, δυνάμει του συνταγματο τη χώρας. Στη συνέχεια, ένα μεγάλο τμήμα τη διεθνούς Κοινότητα και κυρίως οι χώρε της Λατινικής Αμερικής τον ανεγνώρισαν ως πρόεδρο τη χώρας. Και έχουμε πάνω από 40 νεκρούς και περίπου 900 ε, τραυματίε. είχαμε κατόπιν αυτών των ε, διαδηλώσεων και τώρα έχει κατέβει στο πεζοδρόμιο ο λαός και ζητάει δημοκρατία, ελευθερία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο κατά αυτή την θητεία ήδη 8 φορές έχει αποφανθεί για την κατάσταση στη χώρα και ουδεμία άλλη χώρα δεν έτυχε τόσης προσοχή. Δυστυχώς η κατάσταση επιδεινώνεται και φτάνει στο σημείο μη επιστροφής. Το καθεστώς Μαδούρο ε, οδήγησε στο να εγκαταλείψουν τη χώρα 3.000 Πρόκειται για μια ροή μεταναστευτική που είναι η πιο μεγάλη στην ιστορία τη Λατινική Αμερική. αν δεν αλλάξουν τα πράγματα σύντομα στη χώρα, τότε θα γίνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και οι συνέπειε θα είναι καταστροφικέ για όλη την ε, περιοχή. Ενώπιον αυτών των γεγονότων τη προηγουμένη ε, εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι δυνατόν να μένει άπρακτο να σιωπεί και ήδη ήρθα σε τηλεφωνική επαφή με τον πρόεδρο Γκουαϊδό που είναι ο μοναδικό μα συνομιλητή, ούτω ώστε να τον ε, διαβεβαιώσω για την υποστήριξή μα και είπαμε ότι έχουμε ήδη το 17 που είναι το ε, βραβείο Ζαχάροφ στην ε, αντιπολίτευση μας ήταν η πρώτη που καταγγείλαμε την ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είπαμε να υπάρχουν κυρώσει κατά τη κυβέρνηση και να υπάρξει κάτι στην περιοχή, κάποια μέτρα για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες. Κάποιες ε, χώρες ενδιαφέρονται για το πετρέλαιο, εμάς μας ενδιαφέρει το πόσο υποφέρει ο λαός. Repito, risus abundat in ores stultorum. Pides la traducción desde el latín en... Al Και οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει κάποια ειρηνική λύση και πώς θα υπάρχει δημοκρατικός μετασχηματισμός ή Άλλο ε, υπάρχει κίνδυνο για την ενότητα της χώρας για να επανέλθει ο, ο λαός στην φυσιολογικότητα να βρούμε φάρμακα, ε, τροφή, να υπάρξουν επενδύσεις στη χώρα. Εμείς είμαστε στο πλάι του λαού της Βενεζουέλας και ενώπιον αυτών των ιστορικών γεγονότων τίθεται εν κινδύνο η δημοκρατία. Οπότε είναι ξεκαθαρό ότι θα πρέπει εμεί να υποστηρίξουμε την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι την καταστολή. Voglio Πρέπει να απευθύνουμε έναν χαιρετισμό και στην οικογένεια του κυρίου Άνταμιτς που στις 13 Ιανουαρίου ε, δολοφονήθηκε. Πρόκειται για το, την σύζυγο του Φανόντος και για τα τρία παιδιά του. Τα πρακτικά της 17ης Ιανουαρίου έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Ωραία. Τα πρακτικά έχουν εγκριθεί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ και 12 ημέρες η Ιταλική κυβέρνηση κρατά ομήρου 47 ε, ε, πρόσφυγε που διασώθηκαν στη Μεσόγειο με τη συνενοχή άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων οι οποίες ήθελημένα ε, στην τύχη των μεταναστών βασίζουν την πονίδιστη προκλογική του εκστρατεία. Αυτά που συμβαίνουν στη Σιρακούζα είναι όνειδο για ολόκληρη την Ευρώπη. Η διαστάσει του μεταναστευτικού φαινομένου πρέπει να μπουν στο κέντρο τη κοινοβουλευτική μα συζήτηση και πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα εργαλεία που διαθέτουμε προκειμένου να σεβαστούμε πλήρω το άρθρο 80 που απαιτεί αλληλεγγύη και σωστή κατανομή των ευθυνών. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ζητώ στην έναρξη τη συνόδου αυτή να γίνει συζήτηση για την περίπτωση του Sea-Watch, ώστε να αποφύγουμε και άλλε τέτοιε παρόμοιε περιπτώσει ούτε στην Ευρώπη ούτε άλλο στον κόσμο. Και θέλω να απευθύνω και μια προσωπική έκκληση, Πρόεδρε. Ε, τις μέρες αυτές που επισκέφτηκα τη Σιρακούζα, ε, είδα ότι η ευρωπαϊκή αντίδραση ε, και απόκριση αμφισβητείται πάρα πολύ. Ο στόχος μας είναι να προασπιστούμε όμως και το αξίωμα του Ευρωβουλευτού διότι πρέπει να μπορούν να γίνουν και συγκεκριμένε ερευνητικέ επισκέψει εφόσον χρειαστεί. Δεν πρέπει να επιτρέπονται αυτά ούτε στην Ιταλία ούτε αλλού. Κάθε Ευρωβουλευτή θα πρέπει να είναι ελεύθερο να εξασκήσει τα καθήκοντά του και τι αρμοδιότητέ του σε οποιοδήποτε τόπο. Δεν μπορεί να ε, μην μπορεί να επισκεφθεί ανθρώπου που του έχει αποστερηθεί η ελευθερία του. Ευχαριστώ. Εάν τα κράτη-μέλη είχαν εγκρίνει τη μεταρρύθμιση του συστήματο του Δουβλίνου, όπω και προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, αυτή η υπόθεση δεν θα είχε καν ε, έρθει στο φω τη επικαιρότητα και δεν θα είχε υπάρξει. Ούτε άλλε παρόμοιε. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να ανασκομποθούν, να βιαστούν και να εγκρίνουν την μεταρρύθμιση του συστήματο του Δουβλίνου. Μισό λεπτό. Ηρεμία. Κυρία Μορβάη, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αντίστοιχα με την Κυριακή έγκαι θα ήθελα και εγώ να προτείνω ε, να γίνει επίγουσα συζήτηση εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας με τα θύματα ε, των αστυνομικών επιθέσεων και της βιαιότητας αστυνομίας του Εμμανουέλ Μακρόν. Όπως γνωρίζετε, 15 άνθρωποι έχουν χάσει το μάτι τους, 80 έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και προτείνω η συζήτηση για την Ουγγαρία να διαγραφεί από την ημερήσια διάταξη, γιατί αυτή η παραβίαση ή παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων στη Γαλλία είναι πολύ σοβαρότερες από εκείνες που συμβαίνουν στην Ουγγαρία. Ευχαριστώ. Sono οι πολιτικέ ομάδε με την ανάλογη αριθμητική συνάθρηση ευρωβουλευτών μπορούν να ζητήσουν την πρόβλεψη θέματο ε, συζήτηση ε, για την μέσα διάταξη. Εάν λοιπόν η ομάδα σα ή ένας ανάλογος αριθμό ευρωβουλευτών το προτείνει, εγώ θα ζητήσω από την Ολομέλεια να ψηφίσει, αν το δέχεται, και η Ολομέλεια θα λάβει την τελική απόφαση. Ε, και για τη δική σα πρόταση και για αυτή τη κυρία Κέγκε. Η κυρία Γκόμες, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτή την τελετή την οποία οργανώσατε, στην οποία όλοι εκφράσαμε το συνέστημα που μας κυριεύει με αφορμή το ολοκαύτωμα. Δυστυχώς όμως είχαμε μία επίθεση κατά του εργατικού κόμματος ε, λόγω αντισημιτισμού και νομίζω ότι αυτό αδικεί όλους, όλους τους ε, Βρετανούς, ε, όλους τους ε, Εβραίους οι οποίοι πολέμησαν τον ναζισμό και πέθαναν γι' αυτό. Δεν ακούστηκε ούτε μία κουβέντα για τους Ρωμά, για τους ΛΟΑΔ που και αυτοί ήταν θύματα του ολοκαυτώματος. Ονορεύολε Γκόμες, Κυρία Γκόμες, σας υπενθυμίζω. Λέγω, υπενθυμίζω ότι τα θύματα του ολοκαυτώματος αλλά και οι survivors, αυτοί που ε, ε, επεβίωσαν, το, το θυμούνται. Και στην, ε, στην ομιλία μου σας υπενθυμίζω αν μου αφήσετε θα σας απαντήσω. Λέω, δεν γίνεται. Έλεγα ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου υπενθύμησα ότι τα θύματα του ολοκαυτώματος δεν ήταν μόνο ε, Ευρωπαίοι πολίτες προέλευσης ελληνική Ήταν και ε, Ρωμά και ομοφιλόφιλοι. Ονορεύολε Άντερσον. Άντερσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να μιλήσω για τη διάταξη 115 του οικονομισμού εκεί που λέει ότι οι δραστηριότητες μας θα πρέπει να γίνονται με άκρα διαφάνεια. Μου προξενεί μεγάλη έβλεξη να μάθω ότι το έλεγχο του κυρίου Βέμπερ έκανε κάτι χωρίς προηγούμενο. Επέβαλε να υπάρξει μυστική ψηφοφορία αύριο τις ψηφοφορίες που θα γίνουν. Δεν νομίζω ότι νομοθετεί κανένα εν, κρυπτό. Ο πολίτη έχει δικαίωμα να ξέρει πω οι εντολοδόκοι του οι εκπρόσωποι του ψηφίζουν και αναγκάζει έτσι όλο το κοινοβούλιο να ψηφίσει με μυστική ψηφορία για ένα θέμα πολιτικό. Αυτό δεν είναι μόνο γελίο. Αυτό υπονομεύει επίση την εμπιστοσύνη του κόσμου στο κοινοβούλιο. Γιατί το Λαϊκό Κόμμα φοβάται να μάθει ο κόσμο τι ψηφίζουμε. Οπότε παρακαλώ κύριε Βέμπερ, κάντε αυτό που πρέπει και μην αφήσετε να παρακάμψει έτσι τις ε, διαδικασίες μας πολιτικές σας ομάδα. Κάντε το σωστό. Ιδάλλως, ντροπή σας. Bene. Un appello, non c'è nessun richiamo all'ordine del... Vi prego di quando ci sono... Όταν μιλάμε για την ημερήσια τη διά, διάταξη, καλό θα είναι να αναφερόμαστε σε σημεία τη ημερήσια διάταξη. Πολιτική συζήτηση θα πρέπει να γίνεται όταν προβλέπεται πολιτική συζήτηση. Θέλω να σα ενημερώσω λοιπόν ότι στι 11 Ιανουαρίου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο απόφαση για τη σύναψη συμφωνία τη αποχώρηση του ΕΒ Βασιλείου, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Βορειοϊρλανδία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομική Ενέργεια. Κατά συνέπεια, το Κοινοβούλιο έχει λάβει έτοιμα από το Συμβούλιο για να δώσει σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο απόφαση αυτή. Το σχέδιο απόφαση μαζί με τη συμφωνία ε, της αποχώρησης έχει αναπευθεί στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων βάσει του παρατήματος 5 του Ιστορικού ε, Κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου κ. Γκονζάλες Πόνς. Για την ημερήσια διάταξη. Ναι, παρακαλώ, λέει ο πρόεδρος. Μετά την εκλογή του κυρίου Κριστιανού Κάριν ε, ω Πρωθυπουργού τη Λετωνία, το Κοινοβούλιο βάσει του στρογγονισμού καταγράφει τη χειρία τη θέση του από τι 23 Ιανουαρίου 2019. Οι αρμόδιε αρχέ τη Λετωνία είναι πάντα μάλλον ευχάριστο να έχουμε έναν Ευρωβουλευτή που γίνεται Πρωθυπουργό. Οι αρμόδιε αρχέ τη Λετωνία ε, με ενημέρωσαν ότι ο ε, Ευρωβουλευτή στη θέση του θα γίνει ο κ. Αλεξέη Λοσκούτοφ Αντικαθιστά τον κύριο Κάριν από τι 24 Ιανουαρίου 2019. Καλώ ορίζω τον νέο συνάδελφο και θυμίζω ότι μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του πλήρω βάσει των προποθέσεων προβλέποντα από τον ιστορικό Κανονισμό. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έλεγξε την κοινοβουλευτική εντολή των κυρίων Μπόγκοσλαβ Αντρέη Σόνικ, Ραλφ Πάκετ και Κάρλι Αντούρσκη και πρότεινε την έγκριση των κοινοβουλευτικών εντολών από Τη 20, 22, 28 Νοεμβρίου 2018 αντιστοίχω. Υπάρχουν παρατηρήσει. Ωραία. Ε, έτσι εγκρίνονται οι κοινοβουλευτικέ εντολέ. Οι αρμόδιε, αρχέ, μάλλον ε, από το ΕΛΚ ζητήσαμε ε, και από την EFTD ζητήσαμε τι εξή αλλαγέ στι επιτροπέ και αντιπροσωπείε του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Λοσκουτόφ στην Επιτροπή ε, και τάξ ε, και στην αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ο κύριος Νάταν Τζίλ στη θέση του κύριου Πάτρικο Φλίν στην Επιτροπή Αλίας. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Οι διορισμοί αυτοί εγκρίθηκαν. Διάφορε επιτροπέ αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διαθεσμικέ διαπραγματεύσει βάσει του άρθρου 69 C, παράγραφο 1 του ιστορικού κανονισμού οι εκθέσεις που αναφέρονται οι εντολές αυτές για τις διαπραγματεύσεις διατίθενται στον ιστότοπο της Ολομέλειας και τίτλους θα δημοσιευθούν στα επόμενα πρακτικά της Συνόδου Ολομέλειας. Βάσει το αρθρο 69 69C, παράγραφος 2, ε, ε, εάν οι ε, ευρωβουλευτές ή πολιτικές ομάδες που φτάνουν την απαρτία που απαιτείται από τον ιστορικό κανονισμό μέχρι αύριο 31 Ιανουαρίου τα μεσάνυχτα ε, δεν προβάλλουν αντίρρηση, τότε ξεκινούν οι διεθνισμικέ διαπραγματεύσει. Ε, αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο ε, και δεν χρειαστεί να ψηφιστεί το θέμα στην Ολομέλεια. Οι επιτροπή θα ξεκινήσουν τι τριμερεί διαλόγου. Επίση, να σα ενημερώσω ότι την Τετάρτη ε, μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου θα συνυπογράψουμε μαζί βάσει τη τακτική νομοθετική διαδικασία, βάσει του άρθρου 78 των Ιστορικών Κανόνων του Κοινοβουλίου, τι σχετικέ πράξει και αυτά θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά. Περνάμε τώρα και στο τελευταίο, το τελικό σχέδιο μερικής διάταξης που εγκρίθηκε από την Διευθυντή των Προέδρων στις 17 Ιανουαρίου, το οποίο σας έχει μοιραστεί. Κύριε Γκονζάλες Πόντς, θέλετε να ζητήσετε αλλαγή στην ημερική διάταξη. Μάλιστα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα ε, να πω το εξής. Ε, είναι εδώ ο Φρανθίσκο Σούκρε στο θεωρείο, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας. Δηλαδή είναι το νούμερο 2 της νόμιμης κυβέρνησης της χώρας αυτής. Επίσης είναι εδώ και ο Αντώνιο Λετέσμα που είναι ο δήμαρχος του Καράκας. Αφού σας άκουσα προηγουμένως κύριε Πρόεδρε, ως εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το μόνο που μας απομένει είναι να κάνουμε σήμερα συζήτηση για την πολιτική κατάσταση στη Βενεζουέλα και να ψηφίσουμε αντίστοιχο ψήφισμα στη συνέχεια. Κύριε Γκονσάλες Πόνς. Ο κύριος Γκονσάλες Πόνς ζητεί σήμερα συζήτηση και ψηφοφορία αύριο. Διαφωνούν βουλευτές. Κανείς δεν διαφωνεί. Το ψηφίζουμε υπέρ της πρότασης του κυρίου Γκοσάλες Πόνς και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Κατά. Ο καθένας μπορεί να ψηφίζει όπως ε, φρονεί. Απόχες. Ε, ωραία. Η συζήτηση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα, λοιπόν, προστίθεται στις ε, συζητήσει τη σημερινή ημέρα και αύριο θα υπάρξει και ψηφοφορία επί του ψηφίσματος. Παρακαλούμε, κύριε Λάγκερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ω Πρόεδρος τη Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, θα ήθελα να ζητήσω αναβολή της συζήτηση για τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν από λίγες μέρες ο ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε ε, εντολή και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε αυτό. Η Επιτροπή μας φρονεί ότι θα πρέπει να έχουμε ε, βαθιά συζήτηση με ψήφισμα στην Ολομέλεια για να έχουμε τη θέση του Κοινοβουλίου για τη Μπάφα. Προετοιμάζουμε ψήφισμα και γι' αυτό το λόγο θα παρακαλούσαμε να αναβληθεί η συζήτηση ε, με την δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου και να συνοδευτεί τότε η δήλωση με ψήφισμα. Η κυρία Κέλλερ θέλει το λόγο. Κατά. Βεβαίως, έχετε το λόγο. Με ευχαριστώ. Κοιτάξτε πώς έχουν τα πράγματα. Το Συμβούλιο και ε, έδωσε την εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα. Αν θέλει το Κοινοβούλιο να έχει τον παραμικρό λόγο στις διαπραγματεύσεις, τότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας τώρα και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Αργότερα δεν θα παίξουμε κανένα ρόλο, δεν θα έχουμε κανένα λόγο και πάλι θα είμαστε τελείως εκτός νυμφώνος και εκπλήσωμαι πάρα πολύ γιατί μέχρι τώρα οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες πάντα αγωνίζονται για ε, επίσημη και τυπική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με εκπλήσει πάρα πολύ αυτή η πρόταση και παρακαλώ να απορρίψουμε την αναβολή. Να δούμε ποια είναι η θέση μας, τα αιτήματά μας για την εντολή και τις διαπραγματεύσεις και να βεβαιωθούμε ότι η φωνή του Κοινοβουλίου θα ακουστεί στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ Οπότε ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση του κυρίου Λάγκια εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για αναβολή σε επόμενη συνοδολομέλεια για την έναρξη των εμπορικών συμφωνιών Ένωση και ΗΠΑ. Άρχεται την ψηφοφορία. Il Η πρόταση απορρίπτεται. Βάσει των ετοιμάτων των πολιτικών ομάδων, μας ενημέρωσαν οι πολιτικές ομάδες. Τι? Έκτο σημείο μετά τη δήλωση του ΣΥΠΑ της προ για τις σχέσεις Κίνας-Ταϊβάν προβλέπετε το θέμα αυτό για επόμενη φορά, όπως και το θέμα ΝΑΙΑΔΕΣ 2, η στήριξη της εσωτερικής μας Οπότε εγκρίνεται και αυτή η αλλαγή. Σε σχέση τώρα με αλλαγέ την Πέμπτη, για αυτό που θέλουμε για τον κύριο Κόρμπετ, ωραία. Ε, η ομάδα EFTD ζήτησε να ψηφίσουμε ε, σε επόμενη φάση την έκθεση Κόρμπετ. Επίσης, η Πράσινη και η Ελεύθερο Συνασπισμός για την Ευρώπη ζήτησε η έκθεση αυτή που ψηφίστηκε απευθείας να αναβληθεί μέχρι την ε, συνόδο του Φεβρουαρίου για να γίνεται ελεγχή συζήτηση έχοντας ακούσει τις παρεμβάσεις υπέρ και κατά, θα ψηφίσουμε για την έκθεση αναβολής της ε, εξέταση της έκθεσης Κόρμπε. Το να έχουμε μια λεπτομερέστατη συζήτηση για το θέμα αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε και στην επόμενη διάσκεψη των Προέδρων και για το πότε θα οργανωθεί. Ο κύριος Καστάλντο τώρα για να παρουσιάσει την, ε, το έτοιμο της ομάδας του. Ευχαριστώ, πρόεδρε συνάδελφοι. Το 107 προβλέπει ότι αλλαγέ στην ε, διαδικασία θα πρέπει να εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή, Επιτροπή Συνεργματικών Υποθέσεων. Αυτό είναι διάταξη του κανονισμού, αλλά επίση πρόκειται και για κάποια βασική αρχή τη δημοκρατία. Αύριο θα ψηφίσουμε τρει τροπολογίε για την έκθεση ε, Κόρμπετ όσον αφορά ε, τον κανονισμό μα, πολύ σημαντικέ, αλλά ποτέ δεν υπευλήθησαν ούτε συζητήθηκαν σε μια σειρά συναντήσεων τη ομάδα εργασία, αλλά και τη επιτροπή το, το, το, το S&D, ο κύριος Σέφλιν και ο κύριος Γκέρντς επίσης είπαν ότι όλα αυτά θα πρέπει να αποφασιστούν από την απόλυτη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ε, που θα ψηφίσουν βάσει κάποιες πολιτικής ε, συγγένειας. Τι κριτήριο, τι κριτήριο καθόρισε αυτή την ε, πρόταση. Όχι, είναι η πολιτική συγγένεια κύριε Σέφλιν και της ομάδας σας αφού διασπαστήκατε για την ε, έκθεση Αρχεντίνη σε σχέση με την ενεργοποίηση του άρθρου 7 κατά της ε, Ουγγαρίας ε, και όλα αυτά πρωτοβουλία της δικής σας ομάδας και επίσης μετά ψήφισαν συναδελφοί σας υπέρ της χώρας μπας και πρέπει να πάτε στους μη εντεταγμένους Ρητορική ερώτηση. Επίσης είχαμε πολιτική συγγένεια όσον αφορά την ερμηνεία των δημοκρατών αρχών για το Φίντες, για το Φίντες το οποίο τόσο πολύ επικρίνεται σε άλλες περιπτώσεις εδώ στην Ολομέλεια για να μην πούμε επίσης για την Άλτε που επανειλημμένα ε, σε μια σειρά ψηφοριών ο κύριος Γκέρεντς πρόσφατα ε, καθόταν ε, δίπλα σε συναδέλφους του και μάζεψε υπογραφέ για την έξοδο της Φιλανδίας από το ευρώ παρά την γενικότερη ρητορική του. Οπότε βλέπουμε ότι η δημοκρατία σημαίνει κατοχήρωση της αντιπολίτευσης και όχι τυραννία της ε, πλειοψηφίας. Ε, Από η ευθυντή ε, ζητώ να αναβληθεί δυνάμει του 149α ψηφορία επί της εκθέσεως Κόρμπετ και σας ευχαριστώ. Κύριε Κόρμπετ, εσείς έχετε το λόγο για να μιλήσετε κατά της πρότασης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά όχι 100% σχετικά με το διαδικαστικό ζήτημα το οποίο είχε προταθεί ε, όσον αφορά την ε, ε, ψηφοφορία σε κάποια ε, ολομέλεια. Και εδώ και καιρό την έχουμε μελετήσει αυτή την πρόταση, αυτή την έκθεση και σας υπενθυμίζω ότι συνετάγει από μια ομάδα εργασίας της Επιτροπής Συνεμωτικών Υποθέσεων, ομάδα εργασίας, όπου όλες οι πολιτικές ομάδες ε, εξεπροσωπήθηκαν. Και επίσης στη συνέχεια το σύνολο της ε, Συνεμωτικής Επιτροπής το εξήτασε, τώρα υποβλεβάλλεται στην Ολομέλεια ε, κατά τα συνήθεια, ακριβώς όπως προβλέπετε, γιατί οι περισσότερες εκθέσεις μας έχουν κάποιες τροπολογίες, έχουμε επίση κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και όλα αυτά κατεβαίνουν στην Ολομέλεια. Ήδη από Δεκέμβρη και πάει στην 1η του Ιανουαρίου ως ε, αναβολή. Μετά από την 1η του Ιανουαρίου πήγε στη δεύτερη σύνοδο του Ιανουαρίου, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, σαν την ε, κυρία Μέη από εκεί, το αντιγράψατε αυτά στο, στο να αναβάλει και να ξαναναβάλει. Μπα και αυτό θέλει το EFTD. Τέλο πάντων, εγώ σα προτείνω να μην εγκρίνετε την σχετική πρόταση. Η ε, κυρία Κέλλερ, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Εμεί τι προτείνουμε, να γίνει κανονική συζήτηση για την έκθεση Κόρμπετ για μας το θέμα δεν είναι πότε θα γίνει τώρα ή το Φλεβάρι. Δεν θέλουμε να αναβληθεί, αλλά να συζητηθεί. Γιατί το Κοινοβούλιο αξίζει να κάνει μια κανονική συζήτηση για τον κανονισμό και το πώς συστήνονται εδώ πολιτικές ομάδες. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Θα πρέπει να γίνει κανονική συζήτηση στην Ολομέλεια, να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Και όχι να το διεκπαιρεώσουμε σε λίγα λεπτάκια. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα για το πώ συστήνεται μια πολιτική ομάδα, για το τι λόμπι κυκλοφορούν και τι κάνουν, τι μάθαμε από το κίνημα Me Too. Αφορά πολλά πράγματα. Πρέπει να γίνει συζήτηση κανονική. Αυτό λέμε εμεί και αυτό θέλουμε. Και μπορεί να γίνει και τώρα, δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε το Φλεβάρι. Μπορεί να γίνει και το Φλεβάρι τώρα, αλλά συζήτηση θα γίνει. Αυτό ζητούν οι πράσινοι. Να ψηφίσουμε πρώτα για την πρόταση της ομάδας EFTD με ονομαστική ψηφοφορία. Εάν η πρόταση εγκριθεί, θα αναλάβει η διάσκεψη των Προέδρων. Εάν όχι και θέλετε, θα ψηφίσουμε τη δική σας την πρόταση, δηλαδή να γίνει συζήτηση εκτός ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε λοιπόν με ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση Καστάλη του ονόματο του τη EFTD. Άρχεται η ψηφοφορία. Avete votato tutti? Εψήφισαν άπαντες. Ωραία. Πέρα στις προφορίες. Η πρόταση απορρίπτεται. Κυρία Κέλλερ, θέλετε να παραλάβετε το έτοιμά σας, την πρότασή σας, μιας και θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Θέλω να ζητήσω να γίνει μια πλήρη συζήτηση για την έκθεση Κόρμπετ σε αυτήν τη φήμη Πολομέλειας. Ωραία. Άρα σήμερα ψηφίζουμε την πρόταση των πρασίνων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι κατά. Αλλά αν θέλετε να ελέγξουμε... Με συγχωρείτε, αλλά ηρεμήστε. Τι έλεγχο θα κάνουμε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Σιγά. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας. Η πλειοψηφία είναι υπέρ. Οπότε προβλέπεται η συζήτηση. Πριν την ψηφοφορία. Βάσει των ε, διαβουλεύσεων με τις πολιτικές ομάδες ήθελα να υποβάλω στην Ολομέλεια τις σχετικές προτάσεις ε, για αλλαγές στην ημερήσια διαταξη. Και έγκαια, καθίστε, σας είδα. Ε, αφήστε με να μιλήσω πρώτα. Μετά λοιπόν τι διαβουλεύσει με τι ε, πολιτικέ ομάδε, θα ήθελα να ψηφίσει η Ολομέλεια για τι εξή αλλαγέ στην ημερήσια διάταξη. Τετάρτη συζήτηση για τι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσθεση, προσθήκη ω πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης ένα γύρο των πολιτικών ομάδων, κοινή συζήτηση για την ισορροπία των φύλων, πρώτο σημείο αύριο ε, το πρωί ε, ισορρόπη εκπροσώπηση των φίλων σε θέση με εκτελεστικών διοικητικών στελεχών εταιριών. Και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση με τον ε, Πρωθυπουργό τη Φιλανδία, Γιούχα Σιπίλα, σχετικά με το μέλλον τη Ευρώπη. Οι ψηφοφορίε θα αρχίσουν στι 12. Επιπλέον, ε, προστίθεται στι ψηφοφορίε η εκθέση Σικέρσκι για τι άμεσε πληρωμέ και την υποστήριξη τη ανάπτυξη τη υπαίθρου για το 2019-2020. Η αντίρρηση για το άρθρο 106 για του γενικώ τροποποιημένου οργανισμού. Η για το άρθρο 106 για το γενικώ τροποποιημένο και ένα συγκεκριμένο είδος καλλιέργειας και βάσει του άρθρου 106 για το βάμβακα που είναι γενετικό τραποποιημένος ε, βάσει του άρθρου 114. Κυρία Κιέγγε, Πρόεδρε, αλλαγή για την ημερήσια διάταξη, γιατί σήκωσα και γι' αυτό το χέρι μου. Έκανα πολύ συγκεκριμένο αίτημα εκ μέρου τη ομάδα μου. Ε, στην Ολομέλη αυτή θέλουμε να γίνει συζήτηση για την υπόθεση Sea-Watch. Ε, η υπόθεση αυτή πρέπει να συζητηθεί στην Σύνοδο της Ολομελίας. Είναι ένα θέμα και ευρωπαϊκό και πρόκειται για παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, έχω κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα. Θέλω να ψηφιστεί. Κυρία μου, όπω προβλέπει όμω ο κανονισμό, από την ομάδα σα δεν ήρθε κανένα αίτημα για αλλαγέ στην μέση διάταξη. Έπρεπε να έχει έρθει εγκαίρω. Ε, γιατί από τι υπόλοιπε ομάδε τα λάβαμε στην ώρα του. Εγώ δεν έλαβα κάτι εξ ονόματο τη ομάδα σα. Γι' αυτό και δεν ψηφίσαμε, διότι ο κανονισμό προβλέπει ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη τη Ολομέλεια η υποβολή του αιτήματο. Δεν είναι δική μου ευθύνη δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν έχει, γίνει, δεν έχει υποβληθεί έτοιμα από την ομάδα σα. Η ημερήσια διάταξη λοιπόν όπω άλλαξε εγκρίνεται. Προβλέπετε τώρα δήλωση του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω στου βουλευτέ ότι για τη συζήτηση αυτή δεν προβλέπεται διαδικασία κατσδιάη, ούτε θα γίνουν δεκτέ ερωτήσει βάσει τη γαλάζια κάρτα και του συστήματό τη. Πρώτη παρέμβαση. η κυρία Τσιότ, εκ μέρους του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, honorable members. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, πριν από δύο εβδομάδε. είδαμε τι διαβήματα ήδη έχει κάνει το Συμβουλίο κατόπιν τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη συμφωνία τη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κατόπιν τη εγκρίσεω τη πολιτική δήλωση. Εκεί όπου ξεκαθαρίζεται το πλαίσιο για τις μέλουσες σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου του Νοεμβρίου. Αυτό έγινε αμέσω μετά αυτή τη τόσο σημαντική ψηφοφορία στο Westminster. Και πρόκειται για μια ψηφοφορία που ήταν ατυχή, που μα λυπεί. Και ελπίζαμε ότι τουλάχιστον αυτό θα είναι ένα ξυπνητήρι, θα είναι σήμα κινδύνου, τόσο ώστε η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο, το Ηνωμένο Βασιλείο, να συνέλθουν και να ξαναβρούν τη σωστή ρότα. Από ό,τι καταλάβαμε από τη χτεσινή ψηφορία όμως και τέτοιο δεν ισχύει. Και τώρα μάλλον η αβεβαιότητα έχει ενταθεί. Τι ρυθμίσεις εναλλακτικέ θα μπορούσαν να υπάρξουν όσον αφορά τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τη χώρα. Πώς είναι δυνατόν αυτά να τα συγκεράσουμε. Ε, μια τέτοια ρύθμιση με μια ξεκάθαρη θέση δική μας ότι η συμφωνία της αποχώρησης είναι καλύτερος δυνατός συμβασμός. Αυτό το κείμενο το οποίο προέγυψε από τις διαπραγματεύσεις. Δεν θέλω τώρα να προβώ σε κάποιο είδου ε, ε, μαντεψιά για το τι θα γίνει σχετικά με αυτές τις προτάσεις, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έτσι όπως είναι τα ε, πράγματα, η άτακτη έξοδος γίνεται πιο πιθανή και οι συνεπιές της θα καταστούν ακόμα χειρότερες για μας και ακόμα χειρότερες για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ε, οικονομική κύκλοι όλο ένα και περισσότερο επισημαίνουν ε, αυτή την κατάσταση αβεβαιότητος και σε σχέση με την τροχιά πήραν τα πράγματα και σε σχέση με το τι γίνεται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητε στη Βρετανία και για τις θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν. Οπότε τώρα οδηγούμεθα σε περισσότερες ε, εντάσεις, συγκρούσεις και Όλα αυτά μας δοκιμάζουν όσον αφορά την ενότητά μας, την αποφασιστικότητά μας, γιατί θέλουμε να αντισταθούμε στον πειρασμό κάποιων διμερών ε, ρυθμίσεων. Για την άλλη μεριά υπάρχει ένας κοινό ε, στόχος όταν ε, τα αναγκαία κατεπιβάντα μέτρα εγκριθούν η ευθύνη και η αρμοδιότητα είναι της κυβέρνησης της χώρας. Εμείς πάντως θέλουμε να βοηθήσουμε, θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της κύρωσης. Οπότε σε σχέση με αυτό, μέσα στα όρια και στο πνεύμα των αρχών μας και των θέσεών μας, όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών και όσον αφορά το backstop, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε επαφές, σε διευκρινήσεις, εάν αυτό βοηθάει τα πράγματα της διαδικασίας κύρωσης και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας δεν προβλέπεται. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση μόλις το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκαθαρίσει ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία θα κάνει και στο μεταξύ εμείς συνεχίζουμε την διαδικασία της ε, κύρωσης σε μας που ε, προχωράει παράλληλα με την διαδικασία που ακολουθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από πλευρά χρονικών ε, πλαισίων, πλευρά περιεχομένων θα πρέπει να εισηγήσουμε την προπαρασκευή για κάθε δυνατό σενάριο, ακόμα και αν έχουμε έξοδο χωρίς συμφωνία. Το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο, επομένως, έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους, ε, τις προπαρασκευαστικές για καταστάσεις ε, έκτακτες ε, ούτως ώστε να υπάρχει ένα στεγανό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ε, νέα νομοθεσία σε αυτή την ύστερη φάση από πλευρά νομοθετικών ερχών, αλλά πιστεύουμε ότι με την συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Και με ενθαρρύνει η συμφωνία που ήδη έχει κλείσει όσον αφορά τις προτάσεις σχετικές με το Brexit. Η Προεδρία σε συνεργασία με εσά θα διευκολύνει το να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για κάτι πήγουσα ανάγκη εγκαίρως και σας ευχαριστώ πρόεδρος εμείς ευχαριστούμε κύριε Ρία επόμενος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής ο κύριος Ζων Κλόντ έχετε το λόγο Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε λιγότερο από 60 ημέρες το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια κακή απόφαση. Ακούστε, ακούστε. Ακόμα και ενώ η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπερασπιζόταν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντα αυτό γινόταν με σεβασμό. Η συμφωνία αποχώρησης και η πολιτική ε, δήλωση που συμφώνησαν 27 και η κυβέρνηση του Ρωμαίου Βασιλείου είναι το αποτέλεσμα. Η συμφωνία αποχώρησης παραμένει η μόνη και καλύτερη δυνατή συμφωνία. Αυτό το είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο, το είπε και το Δεκέμβριο, το είπε και τον Ιανουάριο, μετά από την πρώτη σημαντική ε, ψηφοφορία στη Βολή των Κοινοτήτων. Η συζήτηση και η ψηφοφορία εχθέ στη Βολή των Κοινοτήτων δεν αλλάζουν το γεγονό αυτό. Η συμφωνία αποχώρηση δεν πρόκειται να τύχει επαναδιαπραγμάτευση και οι δύο πλευρές έχουν διατρανώσει ότι δεν μπορεί να επανέλθει σκληρό σύνορο ε, στην ε, Ιρλανδία. Δεν πρόκειται να αλλησθήσουμε στους σκοτεινούς καιρούς του παρελθόντος. Πιστεύω την Πρωθυπουργό. Επίσης πιστεύω ότι χρειάζεται και ένα δίχτυ ασφαλείας που θα πρέπει να μας εξασφαλίζει απέναντι σε αυτό το κίνδυνο. Δεν έχουμε ούτε επιθυμία, ούτε ε, έναυσμα για να χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο ασφαλείας. Αλλά κανένα δίκτυο ασφαλείας δεν θα είναι ασφαλές αν μπορεί να αφαιρείται ανα πάσα στιγμή. Καμιά φορά έχω την αίσθηση από καιρό σε καιρό ότι ορισμένοι ελπίζουν 26 ε, άλλες χώρες να εγκαταλείψουν το backstop και να αφήσουν μόνοι τους την Ιρλανδία την τελευταία στιγμή. Αλλά αυτό δεν είναι παιχνίδι, ούτε είναι διμερός απλώς το θέμα. Αγγίζει την ίδια την καρδιά το τι σημαίνει να είσαι μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σύνορα της Ιρλανδίας είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων μας. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε από τη χθεσινή συζήτηση ότι η βολή των κοινοτήτων είναι κατά πολλών πραγμάτων είναι κατά του Brexit χωρίς συμφωνία, είναι κατά του Brexit έτσι κι αλλιώς, αλλά παρόλα αυτά δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ακριβώς επιθυμεί η Βουλή των Κοινοτήτων. Υπέρ είναι. Η αρχή, ε, η έννοια των εναλλακτικών ρυθμίσεων δεν είναι καινούρια. Συζητήθηκε και στις διαπραγματεύσεις και αναφέρεται και στην πολιτική δήλωση και στην επιστολή μας προς την Πρωθυπουργό Μέη, ο πρόεδρος Τούσκ και ο υποφαινόμενος ε, δεσμευτήκαμε να το διερευνήσουμε περαιτέρω κατά προτεραιότητα. Αλλά η έννοια δεν είναι σχέδιο, δεν είναι επιχειρησιακή λύση. Πολλοί στη Βουλή των Κοινοτήτων και μεταξύ εκείνων που υπερψήφισαν και μεταξύ εκείνων που καταψήφισαν την τροπολογία ε, έχουν επίγνωση αυτού του γεγονότος. Εγώ θα εξακολουθήσω να είμαι σε στενή επικοινωνία και επαφή με την Πρωθυπουργό Μέη, την οποία σέβομαι και τιμώ απολύτως και θα ακούσω τις ιδέες της, αλλά θα είμαι και απολύτως ξεκάθαρος σχετικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία σήμερα παρουσίασα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας πω ρητά ότι η χθεσινή ψηφοφορία ύφξησε τον κίνδυνο μιας άτακτης υποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια ε, συμπεριλαμβανομένου και του χειρότερου δυνατού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε την προετοιμασία της το Δεκέμβριο του 2017 και τις τελευταίες εβδομάδες σε στενή συνεργασία με το Κοινοβουλίο σας κύριε Πρόεδρε επιταχύναμε τις προετοιμασίες μας. Έχω στείλει μια ομάδα σε κάθε πρωτεύουσα για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστήριξε την προσπάθεια αυτή από την αρχή ήδη. Αυτή τη στιγμή Μέχρι στιγμής έχουμε κοινοποιήσει και δημοσιεύσει 88 κοινοποιήσεις για να δείξουμε τις ε, συνέπειες του Brexit σε διάφορα θέματα και 18 προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι τρεις τελευταίες αφορούν το πρόγραμμα Εράσμου, την κοινωνική ασφάλιση και τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα εγκρίθηκαν και παρουσιάστηκαν. Θα ήθελα ήδη από τώρα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενέχονται ε, έτσι ώστε να φτάσουμε σε σύντομα σε λύση για όλα τα επίγοντα θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, περισσότερο από ποτέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την ψυχραιμία της, την ενότητά της, την αποφασιστικότητά της, ε, όπως ε, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Στην υπόθεση αυτή υπάρχει ο εξής χρυσός κανόνας. δεν θα πρέπει να ε, υποτιμούμε ε, την ε, συμφωνία και την πολιτική δήλωση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ είμαι εκφύσιος αισιόδοξο και παραμένω και πιστεύω στους δημοκρατικούς θεσμούς. Έτσι είμαι πεπισμένος και από πεποίθηση. πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία και θα υπάρξει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζού, μαζί συγγνώμη, μου με τη νέα μας εταιρική σχέση. Νυχθημερών εργαζόμαστε για να ε, είμαστε έτοιμοι. Ό,τι και να γίνει, πάντα θα εξασφαλίσουμε ότι θα είστε οι πρώτοι ε, που θα μάθετε τι σημαίνει και οι τελευταίοι που θα αποφασίζετε. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον ε, επικεφαλής διαπραγματευτή κύριο Μισελ Μπαρνιέ, Θέλω να τονίσω και προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον επικεφαλής διαπραγματευτή για το Ευρωκοινοβούλιο, ποια και αν είναι η λύση του προβλήματος του Brexit. Για μας η προάσπιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών 350.000 ε, που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι προτεραιότητα. Το ίδιο και για του Βρετανού πολίτε που κατοικούν σε εμά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ε, αυτή τη στιγμή λοιπόν μας ενδιαφέρουν το ίδιο οι Βρετανοί πολίτες όσο και οι δικοί μας που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριε Μπαρνιέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, κυρία Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε ξανά εδώ στη Σύνοδο Λομέλειας να παρουσιάσω εδώ τις θέσεις μου. Μέρα με τη μέρα, μαζί με τον Πρόεδρο Γιούνκερ, Προσπαθούμε να χτίσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνη, διαφάνεια στο διάλογο και την όλη συζήτηση που από κοινού οικοδομήσαμε. Μαζί σα, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, μαζί με τον κύριο Φερχόφστατ, μαζί με όλους τους συνεργάτες σε κάθε γύρο συζήτηση που έχουμε. Για πρώτη φορά η Πρωθυπουργό Τερέζα Μέη ζήτησε να ξανανοίξει η εξέταση της συμφωνίας αποχώρησης. Και εφόσον θα υπάρχει ψηφοφορία απόψε το βράδυ, υπάρχει και μια απόσταση πλέον σε σχέση με μια συμφωνία που ίδια είχε διαπραγματευτεί και επί της οποίας είχαμε καταλήξει σε συμφωνία. Η Βρετανική κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την ανοιχτή της υποστήριξη στην τροπολογία του κυρίου Γκράμ Μπράντι, ο οποίος ζητά την αντικατάσταση του συστήματος backstop που είχαμε προβλέψει στο πρωτόκολλο για την Ιρλανδία με εναλλακτικές διευθετήσεις. Διευθετήσεις που σε καμία περίπτωση δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη. Ταυτόχρονα η Βουλή των Κοινοτήτων απέρριψε το σενάριο της έλλειψης της απουσίας συμφωνία χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να διευκρινιστούν οι τρόποι με του οποίου θα αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο. Να, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα το απόγευμα. Στη διάρκεια αυτή τη μακροσκελούς και ε, πέραν του συνηθισμένου ε, Και κύριε Πρόεδρε, όπω βρισκόμουν στι πρώτε γραμμέ του αγώνα αυτού ε, στο πλευρό του Προέδρου Γιούνκερ, Τούσκ και εσάς του ιδίου. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πω ότι τα πράγματα ήταν και σοβαρά και δύσκολα. Χθε το βράδυ με τον κύριο Γιούνκερ ε, θυμήσαμε ότι συμμεριζόμαστε τη βούληση του Βρετανικού Κοινοβουλίου να αποφύγουμε την απουσία, την έλλειψη συμφωνίας και με την κυρία Μέη, ε, καλώς καταψηφίστηκε ε, το σενάριο του no deal. Αυτό όμως δεν το απαλήθηκε πλήρως το σενάριο αυτό. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι για μας η συμφωνία της αποχώρησης παραμένει και είναι το καλύτερο μέσο για να ε, προβλέψουμε μια τακτική αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και με τρόπο έφτακτο να μπορέσει η να γίνει σεβαστή η τοποθέτηση τη πλειοψηφία των Βρετανών πολιτών να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί το σεβόμαστε. Πιστεύω ότι παρά τι σημερινέ δυσκολίε μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο υπό την προπόθεση ότι θα είμαστε ταυτόχρονα και ρεαλιστέ και διαυγεί στη σκέψη μα. Θα είμαστε πλήρη σεβασμού και θα αναλάβουμε τι ευθύνε μα. Και η μεν και η δε. Μάλιστα, η μεν μαζί με του δε. Ε, η ο μηχανισμό του backstop για τον οποίο μίλησε ο κύριο Γιούκερ είναι μέρο τη συμφωνία αποχώρηση. Και η συμφωνία αυτή δεν μπορεί να ξαναγίνει αντικείμενο διαπραγμάτευση. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, που ε, συμπίπτουν πλήρω με τι δηλώσει και τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου για το θέμα, δεν αφήνουν να ε, υπάρξουν εδώ αμφιβολίε. Θέλω να πω δύο κουβέντε για το μηχανισμό backstop ώστε όλοι να αντιληφθούν πλήρω περί τίνο πρόκειται. Ο μηχανισμό backstop δεν είναι δογματική απόφαση. Είναι μια λύση, μια ρεαλιστική λύση που προσφέρεται. Επιζητήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και υπό τον πλήρη ελεγχό σα να εξεύρουμε λύσει σε προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όλο ιδιαιτέρω, αλλά όχι μόνον, στη Βόρεια Ιρλανδία με την προοπτική του Brexit ο μηχανισμός backstop, όπω προβλέπεται στη Συμφωνία Αποχώρησης, είναι το αποτέλεσμα, το πόρισμα αυτών των ε, εντατικότατων διετών ε, διπλωματεύσεων που έχουμε ε, ε, διενεργήσει μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και ποτέ κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι μια ρεαλιστική απόκριση για το τι θα γίνει με την ίσο της Ιρλανδίας εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε ε, με την πλήρη του εθνική κυριαρχία να αποχωρήσει όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την Ενιαία Αγορά και την Τελωνιακή Ένωση χρειάστηκαν δύο χρόνια για να βρούμε αυτή τη λύση. Λύση που επιτρέπει να συγκεντρωθούν και να ικανοποιηθούν πολλές προϋποθέσεις ταυτόχρονα. Πρώτη, να αποφύγουμε την, ε, ε, το νέο σκληρό σύνορο μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλαδή να σεβαστούμε τις συνθήκες ειρήνης, διαλόγου και συμφιλίωσης που επικρατούν εδώ και 20 χρόνια στην ίσο της Ιρλανδίας. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής στο Μπέλφαστ. Θυμίζω ότι το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο με την ε, ψήφο της Πρωθυπουργού του επανειλημμένος επανέλαβε την δέσμευσή του να παραμείνει συνεγγυητής της ε, πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας αυτής της Μεγάλης Παρασκευής και με το πρόγραμμα PIS, με το ευρωπαϊκό δίκαιο, με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό εδώ και χρόνια φροντίζουμε να είναι ομαλή η συνεργασία και η συνύπαρξη των διαφορετικών κοινοτήτων στην Ιρλανδία. Πρώτη προϋπόθεση αυτή. Δεύτερη, η βούληση, το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου, της κυβέρνησης του, να παραμείνει η Ιρλανδία, ε, η Βόρειος Ιρλανδία, ένα ξεχωριστό, ε, μια ξεχωριστή επικράτεια του κράτους. Τρίτη προπόθεση, κάτι που ε, για το οποίο είμαστε όλοι συλλογικά υπεύθυνοι. Η διασφάλιση και η προφύλαξη της ε, ενιαίας αγοράς. Αυτό για μας κυρίε και κύριοι είναι καθοριστική σημασία. Τα ευρωπαϊκά σύνορα, επειδή το θέλησε το Ηνωμένο Βασίλειο, θα γίνουν σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί θα σταματούν τα σύνορα τη εσωτερική αγορά. Θα είναι τα νέα μα εξωτερικά σύνορα. Άρα, αυτό που διακυβεύεται είναι η προστασία όλων των καταναλωτών και όλων των επιχειρήσεων της Ένωσης. Για να το πω πολύ πιο σταράτα, η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να φύγει από, το από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ένωση της Εσωτερικής Αγοράς έχει και πρακτικές συνέπειες. Το κάθε εμπόρευμα, το κάθε αγαθό, το κάθε ε, ζωντανό ζώο, το κάθε προϊόν ζωικής ή προέλευσης που έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι απλώς περνάει στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ιρλανδία, αλλά μπαίνει στην εσωτερική αγορά στην εσωτερική αγορά των δικών σας των χωρών. Η φύση, η ποιότητα, η ασφάλεια και η νομιμότητα των προϊόντων αυτών. Η ασφάλεια για την ε, προστασία των ζώων και το λέω γιατί αφορά τους Υπουργούς Γεωργίας και Κτηνοτροφίας των χωρών μας. Όλα αυτά απαιτούν ελέγχους. Ελέγχους που κάνουμε σε κάθε σημείο των εξωτερικών μας συνόρων παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελέγχους τελωνιακούς, υγειονομικούς, οικονομικούς, κτηνιατρικούς και νομικού. Αυτήν την προστασία την οφείλουμε σε όλου μα του καταναλωτέ. Τα 507 εκατομμύρια μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, τα 20 εκατομμύρια επιχειρήσει μα. Το οφείλουμε σε όσου ζουν και εργάζονται στην εσωτερική αγορά. Ιδού. Και μεταξύ όσων σήμερα ζητούν την ε, αναστολή, την απάλληψη του μηχανισμού backstop, υπάρχουν και Βρετανοί βουλευτέ. Μίλησα σήμερα, σήμερα το πρωί με έναν από αυτού είναι σημαντικό να διαπραγματευτούν μαζί μα. Ε, γνωρίζουν ότι ο μηχανισμό backstop όμω είναι η λύση που καταφέραμε με δυσκολία να βρούμε, γιατί όπω είπε και ο πρόεδρο Γιονκέρ, είναι η, ε, ε, η προστασία τη καρδιά τη Ευρώπη. Βρίσκεται στην καρδιά των υποχρεώσεων και των αρχών μα, δηλαδή την προστασία τη εσωτερική αγορά σε όλε τι τις διαστάσει και τι προεκτάσει. Δίκαιο για τι εταιρείε και δικαιώματα των καταναλωτών, για τι επιχειρήσει, για το περιβάλλον. Όλα αυτά είναι στην καρδιά των προτεραιοτήτων μα. Για να είμαι ειλικρινή, όταν ακούω κάποιους που συμμετείχαν και όλα στι διαπραγματεύσει να εκφράζονται όπω τοποθετήθηκαν, ε, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να δεχτώ αυτό το εγκεφαλικό παιχνίδι και τη χειραγώγηση που προσπαθούν να παίξουν. Το παιχνίδι κατηγοριών που προσπαθούν να παίξουν. Και εδώ δεν είναι τόσο απλό ε, να πούμε ότι θα αφήσουμε στην τύχη του το, την εσωτερική αγορά. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να κινδυνεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε και εναλλακτικέ διαθετήσεις όπως αυτοί, αυτές που αναφέρθηκαν χθε από την Βουλή των Κοινοτήτων. Ακούσαμε και το Βουλή τη Ιρλανδία και τι πολιτικέ δηλώσει. Και τα είπε και ο πρόεδρο Γιούγκερ. Θα είναι προτεραιότητα στι μελλοντικέ διαπραγματεύσει. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε εντατικά αμέσω μετά την υπογραφή τη Συμφωνία Αποχώρηση. Σήμερα όμω, κανεί ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη δεν είναι σε θέση να προβλέψει ε, ξεκάθαρα και κατά ποια θα είναι η φύση αυτών των εναλλακτικών διευθετήσεων, εάν θα μπορούν να λειτουργήσουν, εάν θα ε, πλέον ε, ε, απόλυτα του ίδιου στόχου με το μηχανισμό backstop. Αυτά θέλω να σας πω. πλήρη διαυγεία και ε, ηρεμία. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αυτό είναι το σχέδιο συμφωνία που σα προτείνουμε να κυρώσετε και χρειαζόμαστε το μηχανισμό backstop ω έχει. Εάν απορριφθεί στη σημερινή του μορφή, ουσιαστικά απορρίπτεται η λύση που έχουμε εξεύρει μαζί με τους Βρετανούς. Και το πρόβλημα θα παραμένει όπως το περιέγραψα. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα και πέραν των εναλλακτικών διευθετήσεων που επίσης υπενήθηκα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπως και το Ευρωκοινοβούλιο ήδη επανειλημμένος και σαφώς απέριψαν την ιδέα να υπάρξει χρονική, ε, χρονικό όριο ή μονομερής απάλληψη του μηχανισμού backstop διότι σε αυτή την περίπτωση θα αλλοιωνόταν απευθείας η ίδια η φύση του backstop. Δεν θέλουμε εμείς να το χρησιμοποιήσουμε ε, είναι ένα μηχανισμό ασφαλεία που υπάρχει γιατί πρέπει να υπάρξει. Όπω και εσεί έχετε ασφάλεια για τα σπίτια σα, τα διαμερίσματά σα, είναι κάτι που χρησιμοποιείτε εφόσον χρειαστεί. Η συμφωνία λοιπόν αποχώρηση, την οποία συζητούμε και την οποία πολύ καλά γνωρίζετε, πάει πολύ μακρύτερα από το θέμα τη Ιρλανδία. Η συμφωνία αυτή διασφαλίζει τα δικαιώματα 4,5 εκατομμυρίων πολιτών. Κύριε Ταγιάννη, αναφέρατε την προτεραιότητα του Κοινοβουλίου. Είναι και δική μας από την αρχή των διαπραγματεύσεων. Και ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν γίνει η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ε, συμπολιτών μα, των συμπατριωτών μα, 3,5 εκατομμυρίων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τι διαφορετικέ μα χώρε είναι ε, προτεραιότητα. Το ίδιο και για το 1,5 εκατομμύριο Βρετανών που ζουν στι χώρε μα. Παραμένει προτεραιότητα η διασφάλιση των δικαιωμάτων του. Επίση, προστατεύουμε το σύνολο των δικαιούχων του ευρωπαϊκού προπολογισμού και στι 28 χώρε μέλη. Οι δεσμεύσει που αναλάβαμε όταν ήμασταν 28 θα πρέπει να γίνουν σεβαστέ και μετά. Ε, το ίδιο και για τη μετάβαση του, ε, της 21 μηνών για τι επιχειρήσει και τι ε, διοικητικές Ώστε και από τι δύο πλευρέ να ε, είμαστε προετοιμασμένοι και οι μελλοντικέ σχέσει να μπορούν να εξομαλυνθούν. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να διαπραγματευτούμε και αυτέ τι μελλοντικέ σχέσει. Πρέπει να περάσουμε από νέε φάσει, νέα κύματα διαπραγματεύσεων. Αυτή η συμφωνία λοιπόν είναι μια προπόθεση για να δημιουργηθεί και να οικοδομηθεί το κλίμα εμπιστοσύνη μεταξύ ΜΟΝ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια χώρα που θα παραμείνει φίλη, σύμμαχο, εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πραγματική εταιρική σχέση, ε, ακλόνητη και σταθερή. Για τις μελλοντικέ αυτές σχέσεις, οι Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι και θα παραμείνουν πρόθυμοι τι ερχόμενε ημέρε να δείξουν ακόμη μεγαλύτερη φιλοδοξία, να εργαστούν επί της ποιότητας και της, εντατικό, της έντασης που θα έχουν οι μελλοντικέ μας ιδίω οικονομικές σχέσεις. Και το γνωρίζετε κυρίες και κύριοι βουλευτές. Υπάρχουν πολλά μοντέλα συνεργασίας που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Μοντέλα οικονομικής συνεργασίας με άλλες χώρες, τρίτες χώρες. Το καθένα από αυτά τα μοντέλα πρότυπα έχει διαφορετική εξισορρόπηση δικαιωμάτων υποχρεώσεων, αλλά υπάρχουν πολλά. Και απλώς να πω ότι αν τα βρετανικά αιτήματα εξελιχθούν και ξεπεράσουν το θέμα της, ε, την περίπτωση της απλής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, είμαστε και θα είμαστε προθυμότατοι να συζητήσουμε το οποιοδήποτε από αυτά τα μοντέλα για να δούμε τι νέε φιλοδοξίε μπορεί να εκφράσει η βρετανική πλευρά που θα ανταποκρίνεται και στι δικέ μα τι φιλοδοξίε. Όπω είπατε κι εσεί και όπω έχουμε πει και εμεί και θα πει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι με πλήρη διάβια και ρεαλισμό, κυρίε και κύριοι, όπω κάνατε κι εσεί, κυρία Υπουργέ, βρισκόμαστε λιγότερο από 60 μέρε από την τελική προθεσμία, τη λήξη τη προθεσμία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, μέχρι τώρα ήταν η στάση τη Βουλή των Κοινοτήτων θετική για την λύση που ε, είχε προταθεί και ήταν παραδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπε και ο πρόεδρο Γιούγκερ λοιπόν, είναι ε, επίγον και αναγκαίο να προετοιμαστούμε για όλα τα δυνατά σενάρια και να προβλέψουμε όλα τα έκτακτα μέτρα, τα contingency μέτρα που μπορεί να χρειαστούν για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπω διαμορφώνεται μέσα από την δική μα την εργασία, την εργασία των Πρόεδρων, των συνεργατών σα και όλου του ε, συνεργάτε μα στα κράτη-μέλη. Σα ευχαριστώ και για την εμπιστοσύνη σα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαρνιέ. Ε, μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτο, ο κύριο Μπροκ, εκ μέρου του ΕΛΚ. Herr Präsident, Ευχαριστώ πρόεδρε. κύριε Πρόεδρε, κύρια Προεδρεύουσα, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητέ Μισελ Μπανιέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχά τον Ζαν Κλωτ Ιούνκερ και τον Μισελ Μπαρνιέ για την καλή συνεργασία, την πραγματική διαφάνεια, την ενημέρωση που είχαμε, αλλά και το γεγονό ότι μα άκουγαν. Καλό παράδειγμα αγαστή συνεργασία. Και εδώ ερχόμαστε να το συνειδητοποιήσουμε πάρα πολύ καλά ότι στηρίζουμε αυτή τη διαπραγματευτική στρατηγική. Εχθές ζήσαμε μια ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων όπου απέρριψαν κάθε ε, λογική λύση για το νέο δημοψήφισμα, για την Τελωνιακή Ένωση. Το μόνο που συμφωνούν είναι να στείλουν ε, στις Βρυξέλλες για τρίτη-τέταρτη φορά την κυρία Μέη να μιλήσει για το backstop, ουδέν νεότερον. Είναι πολύ σημαντικό τώρα, πριν έρθει εδώ η κυρία Μέη, επιτέλους, να μιλήσουν μεταξύ τους. Είναι σκάνδαλο να μην μιλάει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης με την Πρωθυπουργού τρία χρόνια και παραπάνω. Όταν θες να βγεις πρέπει να ξέρεις ε, τι σε περιμένει πριν επιβαρύνεις τους άλλους. Ελάτε με μία ενιαία θέση, μιλήστε μεταξύ σας, φέρτε μια επικοδομητική ιδέα και λύση στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς είμαστε ενωμένοι, εσείς δεν είστε ενωμένοι. Κυβέρνηση, τόριδες, Λέιμπορ είναι διχασμένοι. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ. Έχουμε αρνητική πλειοψηφία που απαρτίζεται από διάφορες ομάδες. Από τους σκληροπυρηνικούς του Brexit μέχρι εκείνους που είναι υπέρ της παραμονής και αυτοί μπορούμε να προτείνουμε οτιδήποτε. Δεν θα ψηφίσουν αυτοί που θέλουν το Brexit και το σκληρό και εκείνοι που ελπίζουν να παραμείνουν. Οι ε, ορισμένοι θα απορρίπτουν τα πάντα όσο δεν είναι δημοψήφισμα. Αυτούς τους καταλαβαίνει η καρδιά μου, αλλά το μυαλό μου όχι. Και η κυρία Μέι να διαπραγματευτεί ένα οποιοδήποτε backstop, το ίδιο θα το απορρίψουν για τους ε, γνωστούς λόγους. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η Ιρλανδία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε μεγάλη συμμετοχή στη συμφωνία ε, της Μεγάλης Παρασκευής. Θυμάμαι το φίλο μας και παλιό συνάδελφο, τον Τζον Χιούμ, που από εδώ από το Κοινοβούλιο κατέβαλε κάθε προσπάθεια να το κάνει. Και εμείς θα το υπερασπιστούμε και το πρόγραμμα για την ειρήνη. Δεν θέλουμε σκληρά σύνορα εκεί. Αλλά Όπω είπε και η Βρετανική κυβέρνηση, υποτίθεται δεν θέλει και αυτή η σκληρά σύνορα και επανειλημμένα υπέγραψε ότι θέλει backstop το Δεκέμβρη του 2017 για πρώτη φορά. Αυτά πρέπει να τα λέμε ξεκάθαρα. Εμείς θα υπερασπιστούμε την Ιρλανδία και θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα μαλακό σύνορο. Αλλά θα πρέπει να έχεις και την προθυμία του άλλου. Και το σημερινό backstop με αυτή την τελωνιακή ένωση είναι μια βρετανική εφεύρεση, βρετανική πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάνει άλλες προτάσεις. Δηλαδή θέλουν να διαπραγματευτούν κάτι το οποίο πρότειναν οι ίδιοι. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί. Μιλήστε μεταξύ σας. Στο Λονδίνο. Και λύστε το μεταξύ σας. Και αν έχουμε την ε, συμφωνία αποχώρησης, υπάρχει και μεταφατική ρύθμιση, όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε πάρα πολλά πράγματα που εκκρεμούν. Νορβηγία, Ελβετία, ό,τι θέλετε συζητάμε για τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά γι' αυτό δεν χρειάζεται backstop. Κατά 99% στη μεταβατική περίοδο ε, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί το backstop. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τίποτα στην ουσία. Αυτοί δεν θέλουν συμφωνία για τους διάφορους λόγους δικούς τους που σας ανέφερα. Λοιπόν, θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Βεβαίω, ε, τώρα είμαστε προετοιμασμένοι με την νομοθεσία και είναι σημαντικό ότι είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε αν έρθει πρόταση για να βρεθεί λύση. Τα καλωσορίζω όλα αυτά. Αυτό που επιβολεί των κοινοτήτων, το ότι δεν θέλουν σκληρό Brexit, ούτε εμεί το θέλουμε. Καλά, εγώ δεν θέλω να φύγουν έτσι κι αλλιώ, έτσι για να ξεκαθαρίσω τα χαρτιά μου και να τα ανοίξω. Αλλά είναι βρετανική απόφαση. Τι να κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε και να περιορίσουμε όσο γίνεται τις ζημίες εκατέρωθεν. Αλλά για μένα είναι ξεκάθαρο, θα πρέπει να το γνωρίζει και ο λαός της Βρετανίας. Η ζημιά για το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πάντα μεγαλύτερη. Η ευρωπαϊκή ε, αγορά είναι 16 φορές μεγαλύτερη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και όσοι παράγουν για την ευρωπαϊκή αγορά θα σηκωθούν να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο και θα είναι μια πικρή ώρα αυτή που θα ζήσει η Βρετανία. Ελάτε να τα βρούμε, ελάτε να συμφωνήσουμε, αλλά θα πρέπει η Βρετανική πλευρά να έχει μία θέση και επικοδομητική. Ευχαριστώ πολύ. Excellent German from the British bench there. Thank you. Εξαιρετικά τα γερμανικά της, της ε, βρετανικής πλευράς εκεί. Επόμενος ομιλητής εδώ, κύριος Γκουαλτιέρη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητέ Μισελ, είναι δύσκολο να πει κανεί ότι δεν βρίσκεστε με μια περίπλοκη δύσκολη καταστάσεω και ότι δεν έχει αυξηθεί ο κίνδυνος του No Η Βουλή των ε, Κοινοτήτων ε, ψήφισε. Δεν θέλει το ένα No Αυτό είναι καλό. Ταυτόχρονα όμω, ζήτησε το backstop να αντικατασταθεί με εναλλακτικέ ρυθμίσεις το οποίο δεν προβλέπεται και είδαμε επίση η ίδια από την που είπαν από λίγες εβδομάδες μας είπε ότι το καλύτερο backstop ήταν ένα απόστασμο τμήμα της ε, καλύτερης δυνατή συμφωνίας τώρα, τώρα ζητεί την αντικατάσταση αυτού αυτό ε, έχει φέρει ε, συμπαράταξη και απέφυγε το διχασμό στο κόμμα της αλλά έχει μπλοκάρει την κατάσταση. Θα πρέπει να σε εκείνη γιατί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στην εντολή τους προς το διπραγματευτή ξεκαθάρισαν ότι ένα λειτουργικό και δεσμευτικό backstop είναι το τμήμα της συμφωνίας. Οπότε δεν θα δώσουμε το πράσινο φω σε κανένα deal χωρίς ε, τον backstop να μπορέσουμε να μην έχουμε κλειστά σύνορα στην Ιρλανδία, να συνεχιστεί η ειρήνευση εκεί, η ειρήνη εκεί να διασωθεί. Αυτό δεν είναι μικροπολιτική και οπότε αυτό είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο. Και το backstop αποτελεί μια εγγύηση, αποτελεί μια επιλογή, μια τελευταία λύση και είναι αναγκαίο για να εξασφαλίσουμε ότι αν έχουμε μια συμφωνία και της μέλους και στον Οικονομικό Βασιλείο δεν υπάρξει μέχρι το τέλος της περίοδου τότε τα ελάχιστα διασφαλιστικά μέτρα θα πρέπει να ισχύσουν για να μείνουν ανοιχτά τα σύνορα και έτσι να διασωθεί η νέα αγορά. Και δεν χρειάζεται να σας επαναλάβω ότι έχει αλλάξει τον το απαιτήσει των Βρετανών και αυτό δεν ήταν μια εύκολη παραχώρηση από πλευρά μα. Το κάναμε όμω για να επιτρέψουμε στην Βόρεια Ιρλανδία να μείνει τμήμα τις ίδιες τελειωνικής υπηρέτες όπως το υπόλοιπο βασίλειο και έτσι να μην έχουμε ποσοστώσεις, ε, ελέγχους, δασμούς και αυτό το, το, το, το συμφωνήσαμε παρά το ότι είχαμε την αρχική πρόταση η οποία ήταν δίκαιη, απλή και δεν, δεν επέβαλε κάποιο είδους ε, περιορισμούς ε, στο εμπόριο της θάλασσα της Ιρλανδίας. Γι' αυτό και δεν θέλουμε να υπάρχει ένα τέτοιο νοντήλ. Φυσικά το νοντήλ είναι κακό για όλες τις πλευρές, αυτό θα ήταν ένα ναυάγιο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ορθώς οι ευρωβουλευτές ξεκαθάρισαν, συγγνώμη οι βουλευτέ είπαν ε, ότι αυτό δεν το δέχονται και επαναλαμβάνουμε σήμερα για άλλη μια φορά ότι θέλουμε να υπάρξει όσο γίνεται πιο στενή σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και τη ε, Ευρωπαϊκής ε, πρόκειται για κόκκινη γραμμή του Βασιλείου που μέχρι τώρα μας ε, εμπόδιζε. Αυτό για μας σημαίνει ότι η μόνη εναλλακτική στο backstop είναι μια στενότερη σχέση με την χώρα. Οπότε αν θέλετε να εξασφαλίσουμε το να μην επικαλυστεί κανείς το backstop, τότε φτιάξτε μια θετική πλειοψηφία για μια πιο φιλόδοξη σχέση για την Ελληνική Ένωση και κάποιο είδου καλύτερη ευθυγράμμιση με την ενιαία αγορά. Λιγότεροι από δύο μήνε απομένουν ε, μέχρι την αποχώρηση. Κατεπηγόντω θα πρέπει να δούμε μια επικοδομητική πρόταση από ε, το Ηνωμένο Βασίλειο για να σταματήσει η εμπλοκή. Αλλιώ θα πρέπει να ξαναρωτηθεί ο Βρετανικό λαό αν χρειαζόνται περισσότερο χρόνο και σε αυτό είμαστε νυχτοί. Αλλά χρειάζεται ένα ξεκάθαρο πλάνο, μια ξεκάθαρη πρόταση για το πώς αυτό θα βοηθήσει. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε μια παράταση για ψεύτικες υποσχέσεις ε, και τα λοιπά. Εμείς είμαστε ε, συνασπισμένοι, είμαστε συσπηρωμένοι. Ε, μπροστά έχουμε τον διαπραγματευτή μας ξεκάθαρη εντολή και θα ακούσουμε τι θα πει και ό,τι έχει πει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενότητα. Ανησυχούμε αλλά και είμαστε αισιόδοξοι ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Σας ευχαριστώ, Fox, για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστάς. Παρακαλώ να σέβεστε τους ομιλητές, κύριε Κόμπερν. Thank you. Mr. Fox, I hope he shows you respect. Κύριε Fox, ελπίζω και να σας δείξουν τον ίδιο σεβασμό. Κυρία Πρόεδρε, άκουσα πέντε ομιλίε τώρα σήμερα το απόγευμα που περιγράφουν τι προσπάθειε διαπραγμάτευση για τη Συμφωνία Αποχώρηση και πόσο καλή είναι. Όμω είμαι βέβαιο ότι θα έχετε προσέξει όλοι ότι αυτή η ίδια Συμφωνία Αποχώρηση απερίφθη πριν από δύο εβδομάδε στη Βουλή των Κοινοτήτων με συντριπτική πλειοψηφία. Γι' αυτό τώρα δεν είναι στιγμή να ευχαριστούμε του αυτούς μα με, με ρητορικά σχήματα, αλλά πρέπει να συλλογιστούμε σοβαρά. Ήταν δύσκολο να απεμπλακεί το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμω τώρα ο δρόμο που ανοίγεται μπροστά μα είναι ξεκάθαρο, εφόσον επιλέξουμε να τον ακολουθήσουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν εδώ κάποιοι, όπως ο κύριος Μπροκ, που ελπίζει, ε, ακόμα ελπίζουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζουν θέσει που εκφράζουν αυτή την ελπίδα. Όμω αυτό δεν είναι γραφτό να συμβεί. Είναι απλώ, ε, θα ήταν μάλλον απλώ ε, ε, εξωφρενικό και παράλογο να αγνοήσουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο. Και δεν υπάρχει πλειοψηφία στην Βουλή των Κοινοτήτων υπέρ μια τέτοια επιλογή. Η πρόταση για να διοργανωθεί δεύτερο δημοψήφισμα απεσύρθη διότι ε, τύχανε τόσο λίγη υποστήριξη. Η Βρετανική κυβέρνηση και η Βουλή των Κοινοτήτων θέλουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο έφτακτον και με συμφωνία. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε τα του πρωτοκόλου τη ε, Βορείου Ιρλανδία. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να υποστηρίξουμε τη Συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή. Όμω είναι παράδοξο το γεγονό ότι ο μηχανισμό του backstop που σκοπό έχει να αποφύγει το σκληρό σύνορο, ίσω μέσα σε 58 μέρε να γίνει το αίτιο δημιουργία ενό τέτοιου σκληρού σύνορου στην ίσο τη Ιρλανδία. Να επαναλάβω, ο μηχανισμός backstop στην τωρινή του μορφή δεν θα αποφύγει τη δημιουργία σκληρού συνόρου. Ίσα ίσα θα το δημιουργήσει Γι' αυτό λοιπόν ας σταθούμε όλοι δύο λεπτά και ας συλλογιστούμε. Ίσως να είναι εύκολο να καθόμαστε σήμερα και να προασπιζόμαστε χειροκροτώντας την άκαμπτη προάσπιση μιας ήδη καταγεγραμμένης θέσης. Η ιστορία όμως δεν θα είναι τόσο ευγενική μαζί μας, διότι όπως έχουν τα πράγματα συμφωνία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συμφωνία εκτός και οι δύο πλευρές την έχουν εγκρίνει βάσει του νόμου τους. Οπότε δεν αρκεί να επαναλαμβάνουμε μέχρι αηδία ότι η συμφωνία δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Αυτό θα οδηγήσει σε συμφωνία μηδέν. Και όπω επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα οδηγήσει και σε σκληρό σύνορο μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδία. Οπότε ελπίζω ότι ακόμα και σε αυτή την τελευταία στιγμή προσθήκες και αλλαγές μπορούν να γίνουν ώστε να πάρουμε επιτέλους μια καλή συμφωνία και να την πάμε στην Βρετανία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, όπως είπε και ο κ. Μπαρνιέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει έναν εναλλακτικό τρόπο για να διεξαγάγει ελέγχους και εποπτεία χωρίς να υπάρχει νέο σύνορο. Να το δούμε τώρα λοιπόν αυτή την αυτή την, τον εναλλακτικό τρόπο. Ας σκεφτούμε τι μηχανισμούς και τι χρονικά όρια μπορούμε να βρούμε ως λύση. Ας προχωρήσουμε με καλή προαίρεση. Έχουμε δείξει διαλλακτικότητα και γενναιοδορία. Α μην υποχωρήσουμε και φανούμε αδύναμοι, αλλά α φανούμε δυνατοί. Αυτό που αυτή τη στιγμή διακυβεύεται δεν είναι απλώ το σχέδιο συμφωνία, είναι η μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου Α βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια μελλοντική σχέση που θα επιτρέπει να καλλιεργούμε τι κοινέ μα αξίε, τα κοινά μα συμφέροντα και αυτό σε ένα κόσμο βεβαιότητα. Α βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε μαζί Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα για τους ε, φιλελεύθερους και δημοκράτες ο κ. Φερχόφστατ. Μετά τη χθεσινή ψηφοφορία η κυρία Μέη ανακοίνωσε ότι θα έρθει στις Βρυξέλλες και να σας πω ειλικρινά την ε, δική μου την ε, θέση είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Ας έρθει και στο Ευρωκοινοβούλιο επιτέλους. Το έχουμε ζητήσει επανειλημμένως πριν από περισσότερο από ένα χρόνο. Το ερώτημα όμω είναι γιατί έρχεται, τι σκοπό έχει, τι θα κάνει. Θέλει να αλλάξει τις κόκκινες γραμμές, τις απαγορευτικές γραμμές της Βρετανικής κυβέρνησης, τις οποίες έχει παραμείνει η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα. Θα αλλάξει η έκβαση της διαπραγματεύσης της όλης διαδικασίας και η δεύτερη ερώτησή μου, η δεύτερη παρατηρήσή μου είναι τι εντολή θα έχει. Διότι προ στιγμή πρέπει να σα πω, κύριε Φόξ, ότι έχω ή τουλάχιστον μέχρι χθε δεν είχα δει το κοινοβούλιο σα να δίνει μια σαφή εντολή στην Τερέζα Μέη. Ψηφίσανε κατά ε, μια σειρά πραγμάτων κατά της συμφωνίας, κατά της μηδενικής συμφωνίας κατά του backstop, όμως ως σήμερα έχουν περάσει δύο χρόνια και η Βουλή των Κοινοτήτων δεν έχει ψηφίσει ούτε μία πρόταση υπέρ κάποιου πράγματος, υπέρ του ενο ή του άλλου, υπέρ μιας σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ. του τελευταίους δύο μήνες πρέπει να σας πω ότι πραγματικά εξαντληθήκαμε. Εξαντληθήκαμε όχι μόνο από την άλλη πλευρά και εδώ ατελείωτε συζητήσει, μακροσκελέστατη κατάλογη τροπολογιών, τροπολογίε που πήγαιναν δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, που τι επέλεγε ο πρόεδρο. Και χαθήκαμε για μια ελάχιστη διαφορά στην πλειοψηφία. Να σας να φέρω κατάλογο. 4 Δεκεμβρίου τροπολογία Γκριφ, η οποία ήταν υπέρ του Remain. 22 η τροπολογία Κούγκλ, οποία πέρασε στις 8 Ιανουαρίου. Χάθηκε για 7 ψήφους. Μετά μια άλλη ε, τροπολογία, με 23 ψήφους χάθηκε. Η τροπολογία Brady, ε, η τροπολογία υπέρ Μία προς 16 χθε ε, και μια πάλι μια τροπολογία Remain, η Spellman, η οποία ήταν να μην υπάρξει καμία συμφωνία επιτάπητος. Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα, έτσι θα λυθεί το πρόβλημα αυτών των διαστάσεων, με αυτή τη συμπεριφορά, με αυτή τη διαδικασία. Κάθε μέρα μεταβάλλετε τη στάση σας και τις απόψεις σας και δημιουργείτε ένα κλίμα αβεβαιότητας, ανασφάλειας, αντί να οδηγείται σε, κάποιο, ε, σε κάποια τελική έκβαση η μελλοντική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Πραγματικά βλέπω τι συμβαίνει και δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω κάτι που ξεκίνησε σαν ένας τσακωμός και μαλλιοτράβηγμα στο κόμμα των συντηρητικών έχει γίνει υπαρξιακό πρόβλημα για όλη τη Βρετανία. Η τροπολογία Σπέλμαν χθε καταψηφίστηκε με 8 ψήφου, που έλεγε, μάλλον πέρασε η τροπολογία Σπέλμαν που έλεγε ότι είναι, αποκλείεται να μην υπάρξει καμία συμφωνία. Και αποσύρει την πρόταση αυτή και ήρθε πέντε λεπτά μετά η Πρωθυπουργό και είπε ότι όχι, αυτό δεν αποκλείεται. Είναι ένα σενάριο που μπορεί να συμβεί το μηδενική, η μηδενική συμφωνία. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Υπάρχει απουσία βεβαιότητα, απουσία διάβγεια. Και αυτή τη στιγμή, καθώ μιλάμε, λαμβάνει η χώρα μια συνάντηση μεταξύ του κ. Κόρμπιν, του επικεφαλή αντιπολίτευση και του Πρωθυπουργού κ. Μέη. Ελπίζω κάτι να αποφασίσουν κάτι να συζητήσουν που να έχει περιεχόμενο. Όχι μόνο να τρώνε μπισκέ, μπισκότα βουτώντα τα στο τσάι του το απόγευμα. Διότι θα θέλαμε μια λύση στο πρόβλημα. Θα ήταν λύση αν άρχιζαν να συνεργάζονται για μια διακομματική προσέγγιση. Μπα και μάθουμε κι εμεί ποια είναι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στο μέλλον. Δεν την γνωρίζουμε ακόμα. Κύριε Φόξ, θα πρέπει πρώτα να μπει η χώρα σας και μετά τα κόμματα. Πρέπει να μας πείτε ως χώρα πώς βλέπετε τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασίλειου. Όχι να χρησιμοποιείτε και να κάνετε κατάχρηση της ύπαρξης του Brexit για να προχωράτε σε διελκυστήμβες δύναμης μεταξύ εσάς των ιδίων. Και η Πρωθυπουργός Νέη ας έρθει, να έρθει στις Βρυξέλλες ε, να μας πει ποια είναι η πλειοψηφία του κόμματό της και τι θέλει για τη μελλοντική μας σχέση αυτό η πλειοψηφία. Να που έγκυται η λύση για τον backstop. Διότι εάν υπήρχε στενή σχέση, βαθιά όπως αυτή που περιέγραψε ο κύριος Μπαρνιέ, τότε το backstop θα υπάρχει. Αλλά δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί. Θα είναι θεωρητική διασφάλιση δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιείται καθημερινά. Οπότε και πάλι είμαστε έτοιμοι να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το είπε και ο κύριος Μπαρνιέτα και ο κύριος Γιούγκερ. Είναι στιγμή η πολιτική τάξη της Βρετανίας επιτέλους να πάει και σε αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα εξπρές, διότι εσείς θα πληρώσετε το τίμημα εάν δεν υπάρχει σαφήνεια. next Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Σκοτ Κέιτο για τους ε, πρασίνους. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Westminster καταραίει. Έχουμε εσωτερικές αντιφάσεις λόγω του Brexit που ε, αναδύθηκαν χτες. Τελικά ήταν ένα σύνολο συνθημάτων. Ποτέ δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι σαν την θέση προς διαπραγμάτευση. Ε, τώρα τελειώνει αυτή η ιστορία, ξεγυμνώνεται η υπόθεση και βλέπουμε όλες αυτές τις φάνταστες ε, ιδέες, αποτυχία και αυτό το χάος του Westminster σημαίνει ότι οι περισσότεροι Βρετανοί γνωρίζουν ότι το μέλλον της χώρας είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εδώ μπορούμε να συνεχίσουμε να, να, προς αυτό το όραμα που είναι το πιο πτωσμό για την ειρήνη, να αντιμετωπίσουμε όλα τα υπερεθνικά ζητήματα όπως είναι του κλίματος πρόκειται για την πλειοψηφία και οι νέοι ψηφοφόροι θέλουν να μας ψηφίσουν να βελτιώσουν την Ευρώπη μέσα σε κλίμα φιλίας όλο ένα και περισσότεροι και τώρα έχουμε τους φουλευτές απέριψαν τον Οντήλ άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις πώς αυτό θα γίνει remain, πώς θα μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να αποφασίσει ο λαός και η εχθρότητα αυτών που θέλουν τον Brexit τους βλέπουμε εδώ απέναντί μας ε, η εχθρότητά του εναντί αυτών των δημοκρατικών αρχών σημαίνει ότι φοβούνται γιατί ξέρουν όπω ξέρουμε και εμείς ότι η θέληση του λαού άλλαξε, ε, άλλαξε το ρεύμα, όχι στο χάος του Brexit. Συνάδελφοι, αν μπορούσα, που δεν μπορώ, θα απαγόρευμα τη, τη λέξη βλακή, σκουπίδια και δεν συμφωνώ μαζί σας που την είπατε κύριε. Λέει στον κύριο Φάρατζη, πρόεδρος. Τσίμερ. Σας παρακαλώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα. Το, το, το, ελάχιστο μπορούμε να κάνουμε είναι να σεβαστούμε τον εκάστοτε μιλήτη. Έχουμε ένα σωρό ομιλητέ. Να και εδώ βλέπω προ τα δεξιά μου πάρα πολλοί, πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι παρεμβαίνουν. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι δυνατόν να το καταντήσουμε θέατρο εδώ στο Κοινοβούλιο. Ούτε είναι εδώ η Βουλή των Κοινοτήτων. Εδώ είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φυσικά και σήμερα στην πολιτική μας ομάδα το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Τι θα κάνουμε σε σχέση με τη χτεσινή ψηφοφορία και την κατάσταση που έχει προκύψει και για μας ως πολιτική ομάδα τα πράγματα είναι σαφή. Εμείς στηρούμε, μένουμε στη συμφωνία για την αποχώρηση που ήταν η μόνη εφικτή λύση. Δεν είναι το καλύτερο δυνατό που θα επιθυμούσαμε για να οικοδομήσουμε τις μελλοντικέ μας σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά από ό,τι φαίνεται είναι αυτό που με μεγάλη ενέργεια, κόπο, απώλεια νεύρων πετύχαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο να εκπονήσουμε και κάποια στιγμή πιστεύω θα πρέπει κάποιος να αποφασίζει ε, αν αυτό που μπορεί να επιτύχει από κοινού με κάποιον άλλον, αν το τιμάει ή αν ο καθένας προσπαθεί από την πλευρά του να κερδίσει κάτι παραπάνω, να βγάλει κάτι και τελικά να ανατρέψει και να απειλήσει μαζικά τα συμπεφωνημένα. Και θέλω να θυμίσω εδώ και ε, το λέω και εν ώψη των συναδέλφων ε, και υπόψη των συναδέλφων στο Ηνωμένο Βασίλειο, Συμβουλή των Κοινοτήτων. Πριν από δύο χρόνια περίπου, τι καταφέραμε, να έχουμε επιρροή στην εντολή που έλαβε ο κύριος Μπαρνιέ. Και στη συζήτηση αυτή μεταξύ άλλων καταφέραμε να καταδείξουμε πόσο σημαντικό είναι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και των Βρετανών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός για αφετέρου να υπάρχει ε, πλήρως το θέμα ε, της ε, σταθεροποίησης της νευτικής διαδικασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά ήταν οι κόκκινε γραμμέ. Δεν ήταν τα δικά μα συμφέροντα. Αλλά η σταθερότητα και η ειρήνη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αρχέ Γενάρη, στην πρώτη ψηφοφορία, είδα πολύ προσεκτικά τη συζήτηση και τη χθεσινή στη Βουλή των Κοινοτήτων. Και έχω την αίσθηση ότι δεν μας παίρνουν σοβαρά οι Βρετανοί μας συνάδελφοι και ορισμένοι δεν κατανοούν κάποιες διαδικασίες και συζητούν, λες και είναι οι μόνοι που θα ψηφίζουν για τις αλλαγές. Αγαπητοί μου συνάδελφοι στο Λονδίνο, θα πρέπει να συζητήσετε και μαζί μας ε, για αυτά τα θέματα και να λάβετε υπόψη τη δική μας θέση. Δεν μπορεί να υποδίεστε ότι ισχύει η, Βρετανική Αυτοκρατορία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε τη δική μας δημοκρατία. Μέχρι τώρα ήσασταν τμήμα τη και πάντα πάντα φρόντιζα πάρα πολύ και εκτιμούσα πάρα πολύ ε, να ακούω αυτά που ήξερα από την Βρετανική διπλωματία και πραγματικά έχω φρίξει από αυτό το θέατρο που μας παίζουν. Είναι πολύ σημαντικό να επανέλθουμε, να επανέλθουμε στα βασικά και στα αυτά που θέλουμε τελικά να πετύχουμε και να μην περιχαρακωνόμαστε και κλεινόμαστε. Και η μόνη ελπίδα που έχω, το λέω, είναι στη συνεννόηση Κόρμπιν Μέι να υπάρξει κάποια μετακίνηση υπέρ των διαπραγματεύσεων με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μπορεί να λένε συχνά ότι είμαστε πρόθυμοι να έχουμε ε, συνεργασία. Αλλά αυτό που δεν θα κάνουμε, τουλάχιστον η δική μου πολιτική ομάδα, και χαίρομαι που οι περισσότερε από τι άλλε ομάδε το βλέπουν αντίστοιχα και παρόμοια. Εμεί δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν να θυγούν τα εργασιακά δικαιώματα, τα περιβαλλοντικά πρότυπα, η προστασία των ε, καταναλωτών, ούτε πιθαμή, πιθαμή. Δεν θα επιτρέψουμε η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής να μην γίνει σεβαστή ε, σε όλα τις τα τμήματα. Ούτε θα αφήσουμε κλειστά σύνορα στην Ιρλανδία. Ούτε να θεωρούνται πολίτες τρίτων κρατών ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και να υφίστανται διακρίσεις και να τους αφαιρούνται όλα τα δικαιώματα. Αυτό θέλω να το πω συνολικά στους συναδέλφους στη Βουλή των Κοινοτήτων. Τελειώνω. Χάρηκα όταν οι Βρετανοί συνάδελφοι πάλεψαν και απέκτησαν φωνή στη διαδικασία. Αλλά θα πρέπει να την εκφράσουν και τη φωνή τους και δυνατά να μας πούν επιτέλους τι θέλουν. Κύριε Φαράζ, έχετε το λόγο. Ε, όλοι αυτοί, όλες αυτές οι ψηφοφορίες επηρεάστηκαν από το θύμο του κόσμου και είδαμε ότι δεν υπάρχει θέμα δεύτερη δημοσίευση. Τώρα έχουμε το άρθρο 50, δεν είναι πια ω επιλογή και ακούσαμε όλου του ομιλητέ να λένε ότι ανησυχούν και ότι έχει αυξηθεί το ρίσκο του no deal, έχετε δίκιο, μεγαλύτερο ρίσκο. Όχι όμω λόγω του, ότι έγινε χτες το βράδυ, αλλά κύριοι λόγω του των όσων εσείς είπατε τώρα απόψε ακόμα και όταν η Πρωθυπουργό συσπήρωσε μια πλειοψηφία εντάξει δέχομαι ότι έκανε ένα τερατώδες λάθος με τον να προσυμπόραψε για το backstop και τέσσερα τα ξημερώματα έφυγε την Downing Street πήγε ε, να, να σας βρει γιατί βάλετε το τελεσίγραφο και υπέγραψε κάτι που είναι ένα ναυάγιο. Υπέγραψε κάτι που καμία χώρα, εάν δεν έχει χάσει ένα πόλεμο, δεν θα υπέγραφε ποτέ. Ε, τώρα συνειδητοποιούμε το λάθος και η Βουλή των Κοινοτήτων και όλη η χώρα τώρα αναζητούν μια συμφωνία. Ξέρετε όμως κάτι, πριν το δημοψήφισμα ουδής ήξερε ποια είναι, τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, τίποτα άγνωστη. Και τι είδαμε, ότι τώρα στην Βρετανία βλέπουν και εκτιμούν το ότι οι γρυφικότητες των ε, Βρυξελών ε, πείσανε, παρέπισαν, ε, ταπείνωσαν την Πρωθυπουργό και το λαό. δεν μας αρέσει αυτό. Και κάθε φορά που έρχεται και κάθεται για προς προσπαθεί την είναι λογική και εσείς δεν υποχωρείτε ούτε ένα εκατοστό. να, Τώρα το Brexit είναι πιο κοντά. Και γιατί, λόγω της δικής σας γλώσσας, της στάσης σας, όχι μόνο της Κομισιόν, αλλά και ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι ε, του λαού, έναντι της χώρας μας. Και οπότε υπάρχει μεγάλος τιμός τώρα ε, έναντι των Βρυξελών. Και τι, τι, θα έλεγε κάποιο. πρόκειται για φανατικούς που δεν προτίθενται να δείξουν λογική. Κανένα συμβασμό δεν θέλουν. Και βεβαίω η Τερεζα συμβιβάστηκε ξανά και ξανά και ξανά. Ένα σωρό συμβασμοί παρασυμβιβάστηκε. Οπότε αρχίζουμε να λέμε το ότι ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει ότι το no deal είναι καλύτερο από το backstop. Να το μεγάλο πρόβλημα για σας που θέλετε να επανεκλεγείτε σε λίγες εβδομάδες. Γιατί το no deal σημαίνει δεν θα υπάρχουν τα 39 δις. Πού θα βρείτε τα λεφτά. Αυτό σημαίνει ότι 100 εκατομμύρια προσέκο που κάθε μέρα από την Ιταλία θα ακριβίνουν και επίσης και όλα αυτά τα 750.000 γερμανικά αυτοκίνητα που αγοράζουμε άρα τι σενάριο ε, ετοιμάζουμε, γιατί ετοιμαζόμαστε να επικαλεστείτε το 24 ούτως ώστε όταν εμείς ε, φύγουμε τέλος του Μαρτίου να έχουμε δύο χρόνια χωρίς δασμούς, χωρίς ποσοστώσεις και περιορισμούς κανένας ε, είδους. να έχουμε προβλήματα ή δυσκολίες με την Ιρλανδία να έχουμε ξεμπλέψει με το Brexit και εσείς θα προστατευτείτε για δύο χρόνια Α, οι ψηφοφόροι σας. Να, να ποιο είναι το επικοδομητικό βήμα που πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια ήταν μια μακρά και κοπιαστικότατη διαδικασία δυσκολιών, επανειλημμένων δυσκολιών που μας εμποδίζουν να εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως υπόθηκε και με το τρίκ, το βασικό αυτό τρίκ του backstop. Γι' αυτό απορρίφθη η συμφωνία και γι' αυτό επέστρεψε η κυρία Μέη να διαπραγματευτεί και πάλι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που όμω μα είπε δεν θέλει να διαπραγματευτεί. Υπάρχει ψηφοφορία από τη Βουλή των Κοινοτήτων για παράταση του άρθρου 50, όμω ξέρουμε ότι δεν γίνεται να συμβεί αυτό χωρί να συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα ζούμε όλοι για την 29η Μαρτίου. Θα τα καταφέρει το Βρετανικό πολιτικό ε, σύστημα να αποφύγει το δημοψήφισμα για δεύτερη φορά. Εάν δεν έχουμε συμφωνία στις 29 Μαρτίου και φύγουμε χωρίς πράξη αποχώρησης και εκτός κανονικού το άρθρο 50 δεν θα ισχύει πλέον ούτε οι συνθήκες. Εάν η Βρετανική Βουλή δεν το αφήσει αυτό να συμβεί, είναι σαν να εξεγείρεται κατά του Βρετανικού λαού. Θα έχει βαθίε συνέπειε για οποιαδήποτε πίστη στη δημοκρατία που έχει απομείνει στον Ηνωμένο Βασίλειο κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε ο κύριος Γούλφ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τον Brexit. Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Βρετανική Δημοκρατία. Διότι τα τελευταία δυόμιση χρόνια η κυβέρνησή μα έχει χάσει τον μπούσουλα. Αντί να διαπραγματεύεται αποτελεσματικά, ε, συμβιβάζεται και υποχωρεί ε, δείχνοντα αδυναμία. Θέλετε να μα παγιδεύσετε σε ένα μηχανισμό backstop που θα πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Όχι, δεν μπορείτε να μονοπολείτε το πολιτικό προσκήνιο του κόσμου. Θα πρέπει να δούμε τους συνεργάτες αυτού του σώματος και του Westminster που δεν μπορεί να αφήσει τους ε, υποστηρικτές του Ρημένα του Ίσλινγκτον να πίνουν σαμπάνια στην υγεία της απουσίας συμφωνίας. Πέραν όλων αυτών και των αδυναμιών του νόμου, ο Βρετανικός λαός δεν θα σκύψει το κεφάλι. Δεν αισθανόμαστε φόβο, δεν ε, φοβόμαστε μια συμφωνία του ΠΟΕ, δεν φοβόμαστε ένα μέλλον ανεξαρτησία. Η Βρετανική κυβέρνηση επιτέλους κατάλαβε τι θέλει ο κόσμο και επιτέλους θα φροντίσει να απελευθερώσει το εμποριό μα. Καταλαβαίνει ότι η μάχη για αυτοδιάθεση, η ανεξαρτησία και η ελευθερία μα είναι τα βαθύτερα θεμέλια του έθνου μα. Θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε για να μπορέσουν αυτές οι πίστες μας να εκφραστούν ξανά ελεύθερα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το Brexit θα κάνουμε και θα ξαναγίνουμε ανεξάρτητη χώρα και πάλι. Ευχαριστούμε και τώρα για να ολοκληρωθεί η συζήτηση ο λόγο στην κυρία Τσιότ από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, κυρίε και κύριοι σε περίπτωση που η κοινοβουλευτική διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο οδηγήσει σε κύρωση της συμφωνίας ε, ε, αποχώρησης, ελπίζουμε εντός προθεσμίας, θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα και θα αρχίσει η εφαρμογή της. Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να ε, παρακολουθείτε στενά έτσι ώστε να αποδώσει αποτελέσματα προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων και να συνεισφέρει στην εμπιστοσύνη που χρειάζεται για τις διαπραγματεύσεις των μελλοντικών μας σχέσεων οι οποίες ε, ε, μάλλον δύσκολες θα είναι. Ε, γι' αυτό προσβλέπουμε στη συνεργασία σας καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών αυτών τα επόμενα έτη. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Κλείνει εδώ αυτή η συζήτηση αγαπητοί συνάδελφοι. Ο Πρόεδρος, καλησπέρα σα κύριε και κύριοι. Το επόμενο θέμα στην τη διαταξή μα είναι οι δηλώσει τη Επιτροπή όσον αφορά την καταπολέμηση του μίσου και τη ε, βία εναντίον δημοκρατικά εκλεγμένων στην συζήτηση αυτή δεν προβλέπονται μπλε κάρτες. Και τώρα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τζούλιαν Κίνγκ, ο Επίτροπος. Ε, chair, uh, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ. Ε, βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Στην ε, δημοκρατία, ο πολιτικό διάλογο πολλέ φορέ μπορεί να λάβει άγριο ή πολύ άγριο χαρακτήρα. Αλλά το να καταφύγει κανεί στην βία ή να υποδαβλήσει το μίσο είναι απαράδεκτο. Ε, και σωματική βία είναι κάτι το οποίο σοκράτη, είναι κάτι το οποίο ε, αντιβαίνει στις αξίες μας ε, ήδη ε, σήμερα στη σημερινή σύνοδο μιλήσαμε ε, για τον ε, πρόεδρο του Γκντάνσκ. 20 χρόνια υπεραμήθηκε των ε, ελευθεριών των αξιών που είπαμε. Αφιέρωσε τη ζωή του στην πόλη του και στην κοινωνία. Όσο περισσότερο μιλάμε γι' αυτό, τόσο περισσότερο θυμόμαστε τον θάνατο μιας βουλευτήνας της Κόξ του Τζο Κόξ που υπεραμείνθηκε των δικαιωμάτων όλων, όλων στην κοινωνία και αυτών που έφταναν από το εξωτερικό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι πολλές φορές ε, οι άνθρωποι παρασύρονται στην ε, βία, ριζοσπαστικοποιούνται από πολλωμένες συζητήσεις, από συνωμοτικέ θεωρίε, από κρίση τη λογή. Μα δεν είναι δυνατόν να έχουμε ελεύθερε εκλογέ. Οπουδήποτε στην Ευρώπη, αν υπάρχει κλίμα μίσου, απειλέ άσκηση βία κατά των υποψηφίων που έχουν δημοκρατική εντολή. Και αυτό το διαπιστώσαμε ακόμα και κατά ε, μελών αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ούτε αυτή είναι στο απειρόβλητο. Άρα αυτό θα πρέπει όλα να τα καταδικάσουμε. Πάντως ε, κάποια στιγμή η κυρία Γιούροβα φέτος μίλησε για το δίκτυο συνεργασίας για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο διάβημα. Είναι θετικό για να δούμε το, το, το σύνολο των μέτρων που ξεκίνησαν να θεσπίζονται από το φθινόπωρο. Στενότερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, και έτσι όλοι μαζί να επισημάνουν και να αντιμετωπίσουν ε, τις απειλές κατά των δημοκρατικών λειτουργιών και να προστατευτούν οι εκλογές. Έγινε μια σειρά ανταλλαγής απόψεων πέρσι όσον αφορά τις σχετικές απειλές και αυτό περιλαμβάνει και τα γεγονότα του Απριλίου, δημοκρατική συμμετοχή όσον αφορά τα των εκλογών, μια διάσκεψη τον Οκτώβριο για τις εκλογές την εποχή των ψηφιακών, το Νοέμβριο ένα συμπόσιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα, οπότε με όλε αυτέ τι ενταλλαγές απόψεων προκύπτει ένα, το εξή. ότι μπορεί να έχουμε μίσο με την παραπληροφόρηση, με τι ε, εκστρατείε αμάύρωση που πολλέ φορέ γίνονται με τα κοινωνικά μέσα δικτύωση ή που τέλο πάντων αυτά τα δίκτυα είναι ε, κάτι που το επιταχύνει. Ε, ε, κάτι το οποίο γίνεται πολλές φορές από τρίτες χώρες φέρνουν αυτόν τον καταλήτη. Πολλές φορές ε, υπάρχουν διάφορα συμφέροντα μέσα στις χώρες μας ε, που δεν ενδιαφέρονται για το συμφέρον των πολιτών και της δημοκρατίας. Οπότε το να καταπολύσουν αυτά τα φαινόμενα, αυτό είναι μια πρόκληση. Οι απειλέ είναι κάτι που γνωρίζει σύνορα. Θα πρέπει να φροντίσουμε τι θα γίνει με τις εκλογές, τι θα γίνει με τις πολιτικές αγορεύσεις θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ψευδείς πληροφορίες ε, και να αντιμετωπίσουμε τις ε, απειλές. Επίσης, έχουμε και ε, πολλές φορές το τι γίνεται με τη χρηματοδότηση, την προεκλογική, και επίση το ίντερνετ που χρησιμοποιείται για να παρακάμψει το, το εκλογικό δίκαιο. Ε, αυτά κάνουν το πρόβλημα ακόμα πιο αγανθώδες. Ε, γι' αυτό και θα πρέπει να συνεργαστούμε και έτσι να εξασφαλίσουμε το ότι μπορούμε να συγκεράσουμε τους πόρους που χρειάζονται, τις γνώσεις που χρειάζονται για να είμαστε σε μεγαλύτερη ετοιμότητα για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα και στα πλαίσια τη δικτύου συνεργασίας για τις εκλογές συζητήσαμε το τι μπορεί να γίνει ε, να φέρουμε κοντά τους, ε, πελά, τους ε, πολίτες να αποκτήσουν ξανά την εμπιστοσύνη να δούμε τι έγινε στη Σουηδία ε, στις τελευταίες αυτό το πράγμα προς μίμηση και έτσι να εμπλακούν περισσότεροι πολίτες να γίνουν στεγανές οι δημοκρατικές διαδικασίες αυτό το απέδειξε ότι γίνεται η Λετωνία γιατί Εκλήθησαν οι πολίτες να καταγγείλουν το τι παράνομο έχει χρησιμοποιηθεί στην ε, ε, προεκλογική εκστρατεία και να το κατήγουν στις αρμόδιες αρχές. Επίσης χρειάζεται προστασία όσον αφορά τους οικονομικούς ελέγχους, να μην έχουμε παραθυράκια, ε, γιατί έχουμε τις νέες τεχνολογίες που οδηγούν σε καταστρατήγηση του νόμου σχετικά με τις εκλογές. Εκεί θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ε, θα πρέπει έτσι να συμπληρωθούν οι κρατικές προσπάθειες και έτσι να εξασφαλίσουμε ότι οι ιντερνετικές πλατφόρμες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να είναι στο ύψος των περιστάσεων να κάνουν όλα αυτά που έχουν υποσχεθεί σε σχέση με κώδικες διαντολογίας, όχι στη, στο, στο, στο στην παραπληροφόρηση, ε, στη ρητορική του μίσους και έχουμε αυτές τις αιτήσεις εκθέσεις όσον αφορά ε, το πόσο προοδεύουν οι Ιντερνετικές πλατφόρμες για την παραπληροφόρηση. Χθες αυτά τα συμφωνήσαμε τώρα όσον αφορά τη ρητορική του μίσους θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι δεν πρόκειται εδώ περί της ελευθερίας του λόγου είναι καθήκον, καθήκον όλων των ερετών να το καταδικάσουν ε, να μην το υποδαβλίζουν οπότε έχουμε και το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων που προβλέπει ότι τα κράτη μπορούν να καταπιέζουν οτιδήποτε έκφραση που προάγει, βοηθά, δικαιολογεί ε, το μίσος και ε, τη μειονεκτικότητα. Οπότε βλέπουμε ότι πρόκειται ουσιαστικά για απειλή προς την κοινωνία. Στρέφεται κατά ε, του, του, του κόσμου, έχει θύματα άμεσα αλλά επίση ε, σκοτώνει και την ελευθερία της έκφρασης και όχι μόνο τα αρνητικά, αλλά παντού στην κοινωνία. Οπότε ο στόχος βασικός θα πρέπει να είναι ότι ε, αυτοί που χρησιμοποιούν την ε, ρητορική του μίσου προσάγονται στην δικαιοσύνη και θα πρέπει να ισχύσει η απόφαση πλαίσιο για ρατσισμό και ξενοφοβία. Οπότε το πρόβλημα που το έχουμε να για τις εκλογές είναι περίπλοκο, δεν είναι δυνατόν να λυθεί από μόνο μία αρχή, από ένα κράτος ή οποιαδήποτε εταιρεία ιδιωτική. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να αφαιθεί μόνος του να τα αντιμετωπίσει ή να αφήσουμε έναν μόνο να έχει όλα τα του στα χέρια του, να κρίνει μόνο ένας. Όχι, χρειάζεται σφαιρική προσέγγιση για ασφάλεια σε εκλογές, για νομιμότητα, για δημοκρατικό διάλογο, για ισότητα ενός εκλογές και για ασφάλεια όσων εμπλέκονται στις δημοκρατικές διαδικασίες. Ποτέ να μην ξεχνούμε ότι όλες μας οι προσπάθειες πρέπει να κατατείνουν στο πώς θα υπάρχει κράτος δικαίου, σεβασμός δικαιωμάτων, ελευθερία της έκφρασης συγκεκριμένα και ελευθερία του συνέρχεστε, γιατί αυτό είναι καθήκον μας για τις εκλογές και τη λειτουργία της δημοκρατίας. Μπράβο, ευχαριστώ που το έχετε στη διάταξη και περιμένω πώς και πώς να ακούσω την συζήτηση και στη συνέχεια μέχρι τις εκλογές να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ακολουθεί η συζήτηση. Θα ακούσουμε πρώτα τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και μετά τους ε, ε, μη εγγεγραμμένους και τους ε, λοιπούς. Ο κύριος Λεβαντόφσκι από πλευράς ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα εδώ στην καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Μιλούμε για το πώς θα προστατεύουμε τη δημοκρατία από τη ρητορική του μίσους που καταστρέφει την κοινωνία, προάγει τη βία και ε, τα εγκληματικά καθεστώτα. Σήμερα ε, τιμήσαμε τη μνήμη του ολοκαυτώματος. και αυτό δεν αφορά μόνο τη δολοφονία του φίλου μου, Παύλ ε, Ανταμόβιτς, του Δημάρχου του Γκτάνσκ, αλλά και γενικότερα. Ο άνθρωπος αυτός δεν ένιωθε μίσος, ούτε τους εχθρούς του δεν μισούσε, κανέναν. Και ξέρουμε την πόλη του Γκτάνσκ, ε, ποια ιστορία είχε. Ο ίδιος ήταν πάρα πολύ φιλάνθρωπος, έκανε πάρα πολλά πράγματα για την πόλη, για τους συνανθρώπους του, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα παρευρίσκεται η οικογένειά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το θέμα είναι να στραφούμε στο μέλλον, γιατί το πρόβλημα δεν είναι πολωνικό, αλλά ευρωπαϊκό. Ο κύριος Ανταμόβιτς ε, είναι από την Πολωνία, αλλά είχαμε και την κυρία Κόξ ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ε, Σουηδία και από τη δολοφονία του Ούλοφ Πάλμε ε, και μετά αργότερα της Υπουργού Εξωτερικών και ακόμα και στη Μάλτα και στη Σλοβακία δημοσιογράφοι. Θα πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά. Δεν είναι του περασμένου αιώνος. Έχουν γίνει πάρα πολλά φρικτά στον 20ο αιώνα, αλλά θα πρέπει ε, να τα αντιμετωπίσουμε στον 21ο αιώνα. Η τρομοκρατία τρέφεται από το μίσος και ο κάθε ολοκληρωτισμός, ε, ο μολυσεβικισμός, ε, ο, ναζισμός που στιγματίζουν κάποιους ανθρώπους ως εχθρούς της πατρίδας. Δυστυχώς σηκώνει κεφάλι αυτό στο διαδίκτυο. Ανοίγουν παλιές πληγές. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, είχαμε και στα δημόσια μέσα ενημέρωσης διασπορά μίσους ε, και ε, ουσιαστικά ε, λιντσάρανε τον δήμαρχο Ανταμόβιτς και αυτό το ανεχόντουσαν. Στο Κατοβίτσε το είχαν κάνει και εικονική κρεμάλα και τον είχαν κρεμάσει στην Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ οδυνηρό ε, για τις κοινωνίες μας. Έχουμε τελείως διαφορετικές αρχές και αξίες. Σεβόμαστε τον άνθρωπο, ε, την ποικιλομορφία, την πολυμορφία, την ειλικρή. Ο θάνατος του Δημάρχου Ανταμόβιτς θα πρέπει να είναι ένα καμπανάκι που να μας ταρακουνήσει. δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα πράγματα με εθελοντικούς ε, κώδικες και συμφωνίες. Ε, πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί στην αντιμετώπιση και στο διαδίκτυο, γιατί εκεί είναι τα πράγματα χειρότερα, διότι είναι και ανώνυμα. Για παράδειγμα, ε, και ο Χάικο Μας έχει πει κάποια πράγματα και ε, συστάσεις ο Πολωνός συνήγορος του πολίτη έχει απευθυνεί 20 συστάσεις και στο διαδίκτυο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να νικήσουμε αυτά τα δεινά και να τα καθυποτάξουμε. Αυτό ζητάει και η οικογένεια του Αμόβης για να μην πάει χαμένος, ο άδικο χαμένος Αδαμόβης. Ευχαριστούμε. Και τώρα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες η κυρία Φαγιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι εκπρόσωποι της Λίγκα του Βορρά αποκάλεσαν την συνάδελφό μας Κιέγκε ουρακοτάγκο. Είπαν ότι θα ήταν καλό να την ε, ε, κακοποιήσουν, να τη στείλουν πίσω τη χώρα της εκλουβή και ούτω καθεξής. Η κυρία Φορέντζα κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω τραυματισμών. Άλλοι συνάδελφοι δέχτηκαν γροθοκοπήματα ε, από την Φίντες. Η Σλοβενία ε, επίσης είχε προβλήματα με το κόμμα SDS και με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Κάποιοι αποκλήθηκαν μισθοφόροι με τα χέρια τους βαμμένα με αίμα ε, φωνιάδες ε, ζητήθηκαν ποινικέ ευθύνες και αυτοί που δυσφημούσαν είπαν ότι ε, όχι δεν χρειάζεται γιατί έχω ήδη πάρει εκδίκηση. Σε κάθε περίπτωση, κυρίε και κύριοι, δεν ισχύει αυτό. Θα θέλαμε η πολιτική και η κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην κινδυνεύουν. Πριν από τρει μήνε, οργάνωσα διάσκεψη για τι εκφράσει μίσου στη Λιουμπλιάνα. Στην εκδήλωση αυτή, τονίσαμε και παρουσιάσαμε μια σειρά από φαινόμενα που θα έπρεπε να συζητηθούν εντελεχώ, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ποιο είναι ο ρόλο των μέσων μαζική ενημέρωση, που θα έπρεπε να είναι αντικειμενικά αλλά κατά κατα... κατηγοριοποιούν του ε, υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων ω ρατσιστέ. Δεν θα έπρεπε να απαγορεύεται το μίσο και η έλλειψη ανεκτικότητα στην δημόσια σφαίρα. Και εμεί πάντοτε ε, σεβόμαστε τι αρχέ μα και έχουμε δείξει ανοχή έναντι όσων είναι μη ανεκτικοί. Έχουμε προσπαθήσει με ορθολογικά επιχείρημα γιατί να τους για να του εξηγήσουμε γιατί οι ομοφοβικέ εκρήξει είναι ε, εκτό δημόσια σφαίρα. Και τώρα θέλουμε να ε, φορέσουμε την ελευθερία της έκφρασης όπως μας την έχουν σχεδιάσει εκείνοι. Να τους αφήνουμε ατιμωρητοί να εκφράζονται όπως θέλουμε, όπως θέλουν. Ή να μένουν ατιμόρυτοι οι αντίπαλοι όπως ε, συμβαίνει στην Ουγγαρία. Θα πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να πάψει η καλλιέργεια του φόβου στι καρδιέ των ανθρώπων, γιατί αυτό προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί ε, για να ε, σφετεριστούν την εξουσία. το κόμμα SDS στη Σλοβενία έχει χρηματοδοτηθεί εξωτερικώ από την Ουγγαρία για τη διαφημιστική τη εκστρατεία. Με εθνιστική ιδεολογία, με εκφράσει ε, πρωτογονικέ και βάρβαρες. Αυτοί μάλιστα που είναι τα μεγαλύτερα θύματα είναι κοινωνικά μειονεκτούντε. Δεν θέλουμε λοιπόν ε, άνθρωποι όπω ο Ορμπάν, ο Γιάντσεν και άλλοι να εκμεταλλεύονται αυτές τις εκφράσεις. Οι εκφράσεις πριν μίσου πολύ συχνά κρύβουνταν και ε, καλλιεργούνταν μόνον ε, κρυφά. Τώρα γίνονται και ανοιχτά οι τοποθετήσει αυτέ. Συνάδελφοι, οι εκφράσει μίσου, η βία, σωματική και ψυχολογική, η λεκτική, δεν μπορεί να είναι ένα κανονικό φαινόμενο. Οποιαδήποτε μορφή μίσου θα έπρεπε να απαγορεύεται για του πολιτικού, του δημόσιου λειτουργού, για του πολίτε. Είναι κάτι το καταστροφικό και το αντιπαραγωγικό. Δεν το αξίζουμε ω Ευρωπαίοι, δεν το αξίζει η Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να προειδοποιήσω ποιον προσπαθεί να κερδίσει από αυτόν ότι οι προσπάθειέ σα δεν θα ευδοκιμήσουν. Από την πλευρά των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, καλό όλου να χρησιμοποιήσουν την ορθή του λογική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φαγιόν. Και τώρα εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμισών, ο κύριος Λεγκούτκο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε ομόλογο ότι θα ήμουν πιο προσεκτικός στην νομοθετική ρύθμιση του προβλήματος αυτού της ρητορική του μίσους ή του πολιτικού κλίματος. Είναι πολύ ασαφή και συγκεχημένα αυτά ως έννοιες και χρησιμοποιούνται συχνά από πολιτικούς κατά των πολιτικών τους αντιπάλων. Πάντα εκείνοι είναι που έχουν ρητορική μίσους. Πάντα οι αντίπαλοι μας είναι αυτοί. Έχετε ένα πολύ καλό ε, παράδειγμα. Ακούσαμε δύο παρεμβάσεις πριν από τη δική μου και σε κάθε μία από τις παρεμβάσεις αυτές είμαστε εμείς και, και αυτοί. Εμείς ποτέ δεν είμαστε. Πάντα αυτοί είναι. Και εδώ στο κοινοβούλιο αυτό ε, είναι, που είναι πολύ ε, πολιτικό θεσμικό όργανο. Δεν ακούμε αυτή την επίθεση. Την ακούμε όταν μιλάει κάποιος από αυτό το τμήμα ε, του ημικυκλίου ε, που θεωρείται προσβλητικό τον τιμωρούν και υφίσταται πρόστιμα. Όταν πει κάποιος κάτι φρικτό και τρομακτικό από την άλλη πλευρά του ημικυκλίου, ε, τι να κάνουμε, είναι ελευθερία του λόγου και ποιος ορίζει τους κανόνες και ποιος εκτελεί αυτούς τους κανόνες. Ε, σκέφτομαι τις δύο προηγούμενες παρεμβάσεις και λέω στον εαυτό μου ότι αν αυτή είναι η γλώσσα της αγάπης και της ε, διαλλακτικότητας, τι να το κάνουμε το μίσος και την αδιαλαξία. Πια. Περιτεύουν να σας πω μερικά γεγονότα. Πριν από λίγα χρόνια, μάλλον πριν από λίγες μέρες, δολοφονήθηκε ο δήμαρχος του Γκτάνσκ από κάποιον που ήταν καταδικασμένος εγκληματίας με μεγάλο ψυχιατρικό ιστορικό. Και αμέσως μετά τη δολοφονία, η πολιτική αντιπολίτευση στην Πολωνία κατηγόρησε την πολωνική κυβέρνηση, τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, κάνοντας κάτι ε, ε, που ήταν τελείως μη πολιτικό, ένα ιδεχθές έγκλημα, μια δολοφονία που δεν είχε καμία σχέση απολύτως με την πολιτική, το έκαναν πολιτικό ζήτημα και στράφηκαν εναντίον μας. Ποιο είναι το πιο αήθες, αήθες αν, ανήθικο ε, και οι δεχτές παράδειγμα πολιτικού κινησμού δεν υπάρχει μεγαλύτερο από το συγκεκριμένο τα ακούσατε εδώ μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούσατε ότι ε, λίντσαραν τα μέσα ενημέρωσης τον τα δήμαρχο. Αυτή είναι η γλώσσα της αγάπης, ε, κύριε Επίτροπε. Θα τον τιμωρήσουμε το συνάδελφο του ΕΛΚ ή θα την γλιτώσει. Αν πω ότι με λιντσάρουν εμένα, τι θα γίνει. Κάτι θα πάθω. Ε, οι αρχές ε, θα μου επιβάλλουν κάτι. Εν πάση περιπτώσει. Ποιο είναι το πρόβλημα, ότι ακόμα και ένας τραγικός θάνατος δεν σας αποτρέπει μερικούς από εσά να τον χρησιμοποιήσετε και να τον εκμεταλλευτείτε για τις πολιτικές σας σκοπιμότητες και επιδιώξεις. Αυτός είναι πολιτικός κινησμός. Δεν έχετε κανένα ηθικό φραγμό, δεν τρέπεστε καθόλου τσίπα, δεν έχετε πάνω σας. Όταν πριν από λίγα χρόνια ο κύριος Σόιμπλε δέχτη επίθεση από έναν τρελό, δεν είπαμε για πολιτικό κλίμα. Και ήταν καλή απόφαση. Όταν πριν από λίγα χρόνια κάποιος από το κόμμα μου δολοφονήθηκε από έναν άνθρωπο ηχέφρονα που ήθελε να σκοτώσει ε, τον ε, Κανσίσκη, τον πρόεδρο του κόμματός μας. Εδώ είπαμε ότι ήταν ένα ανθρώπινο σφάλμα και δεν μιλήσαμε ποτέ για μίσος και ρητορική μίσος. Θυμάμαι ε, και μια προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ήσασταν τότε εσείς, και τι έπαθαν, αφασία ε, τότε. Ε, δεν μίλησαν καθόλου. Και έχω ζήσει πολλά στη ζωή μου γιατί είμαι αρκετά μεγάλος, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις αναλογίζομαι και λέω «Μα μου, είναι δυνατόν οι άνθρωποι που θεωρούμε πολιτισμένους να λένε τέτοια πράγματα. Και τόσο χαμηλά πια πέφτουν. Πόσο χαμηλά ακόμα θα πέσουν. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, εξ ονόματος των Πρασίνων, η κυρία Άννα Μιράντα, παρακαλώ. Ε, τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο καιρό οι εξτρεμιστές ε, επιτίθενται στη δημοκρατία. Ε, είναι μια προφασιστική και μια εποχή πριν το φασισμό που πάει από την Ισπανία, την Ιταλία, και τη Γαλλία και δεν έχει πολιτικά σύνορα, ούτε διεθνή σύνορα. Η Ελενάρα Φορέντσα, η Τζούντι Χεντίνη και άλλοι συνάδελφοι ε, καταδικάζουμε ε, τις δολοφονίες γυναικών. Είμαστε υπέρ πολιτικών ε, διαφορετικών εναλλακτικών και μας επιτίθενται μέρα με τη μέρα στο δρόμο, στο δημόσιο λόγο μας, στην άσκηση των καθηκόντων μας. Και εδώ στο Κοινοβούλιο, στην περασμένη σύνοδο, ακούσαμε το εξής. Το αριστερό τμήμα, εμείς δηλαδή, του Κοινοβουλίου, μας είπε κάποιος το ΑΕΛΚ ότι είμαστε ε, απολυτικοί, ότι είμαστε ε, φασιστές, ρατσιστές, ε, αδιάλακτοι. Θα περιμένουμε να τα ακούμε αυτά με σταυρωμένα τα χέρια. Θα πρέπει να απαιτήσουμε να είναι ελεύθερες οι ιδέες μας και να εκφράζονται. Και εδώ στο Κοινοβούλιο είναι μεγάλη ευθύνη μας. Δεν φτάνουν πια τα κούφια λόγια, χρειάζονται έργα. Άλλο είναι η ελευθερία της έκφρασης, όπως είπε ο και άλλο είναι να επιτρέπουμε εδώ να ακούμε ε, ρητορική του μίσους, όπως πολύ συχνά από την άλλη πλευρά της Ολομέλειας. Και το αποτέλεσμα θα το δείτε στις επόμενες ευρωεκλογές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ από την Ενωτική Αριστερά. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Κούνεβα. Παρακαλώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του παύελ Αντάμοβιτς, τον Δήμαρχο του Γκδάνσκ, υπερασπιστή των ανοιχτών συνόρων για τους πρόσφυγες που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής συναυλίας. Εχθροί της δημοκρατίας δεν υπάρχουν μόνο στην Πολωνία. Παρακολουθήσατε τις συνθήκες στις οποίες ψηφίστηκε στην Ελλάδα η Συμφωνία των Πρεσπών γνωρίζετε ότι ενώ αυτή τη συμφωνία χαιρέτησαν όλες οι πολιτικές ομάδες στην ευρώπη οι βουλευτές που την υποστήριξαν κατηγορήθηκαν από κάποιους ως προδότες. κολλήθηκαν αφήσει με τα πρόσωπά τους. Επιτέσεις από κουκολοφόρους με πέτρες και μολότοφ στα σπίτια τους και μέσα τα παιδιά τους αυτοί που οργάνωσαν την επίθεση ενάντια στους εκλεγμένους βουλευτές ήταν ακροδεξιοί και ακραίοι εθνικιστές. Η πολιτική του μίσους και της τρομοκρατίας είναι, είναι πολιτική αυτών που μισούν την δημοκρατία. Η απάντηση είναι μία. Παιδεία και δημοκρατία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Από την ομάδα EFTT, ο κύριος Γιώργ Μόιτεν, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, ε, χαίρομαι που ε, εγγράφει στην ημερήσια διάταξη αυτή η συζήτηση που ζήτησα εγώ. Δείχνει πάρα πολύ ε, ότι χρειάζεται. Ε, το κλίμα στην κοινωνία είναι όλο και πιο οξυμένο. Πολύ συχνά καταλήγει σε σωματική βία κατά εκλεγμένων και σκέφτομαι τον ε, δήμαρχο Ανταμόβιτς του Γκτάνσκ που έπεσε θύμα της ιδεχθούς δολοφονικής επίθεσης. Τα είπε όλα ο συνάδελφος Λεβαντόφσκι. Πραγματικά το πένθος έχει σκεπάσει και άλλες χώρες, όχι μόνο την Πολωνία. Το λέω ξεκάθαρα θα πρέπει όλοι να καταδικάζουμε συστηματικά οποιαδήποτε μορφή πολιτικής βίας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πω ότι η ακροδεξιά βία πραγματικά καταδικάζεται, αλλά η ακροαριστερή βία δεν σπουδαιολογείται πολύ συχνά. Οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες ε, το έχουν κάνει και ιδεολογία. Ο αντιπρόεδρο του S5 Στέγνερ λέει ότι η βία δεν είναι αριστερή. Ο σύντροφό του Μάρτιν Σούλτ, πολύ γνωστό εδώ και μη εξαιρεταίο, λέει ότι η αριστερά και η χρήση βία αλληλοαποκλείονται. Αρκεί να ρίξουν μια ματιά στα βιβλία τη ιστορία. Τα μαύρα κατάστοιχα του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού γεμίζουν χιλιάδε σελίδε και αριστερή εξτρεμιστική ακραία βία είναι ένα πρόβλημα του σήμερα. Κοιτάξτε τι κάνουν οι αντιφασιστικές αριστερές οργανώσεις. Ε, καλούν ε, σε ε, θανατικές επιθέσεις κατά το μελών του κόμματό μου. Εγώ ευτυχώς όχι ακόμα. Ε, θα πρέπει αυτά να τα καταδικάζουμε. Το αντίθετο όμως, εδώ στο Κοινοβούλιο υπάρχουν βουλευτές, Γερμανοί πράσινοι που στην Ολομέλεια ε, ποζάρουν με την σημαία την αντιφασιστική. Ε, ε, ε, οι αριστεροί εξτρεμιστές τους βρίσκουν σύμφωνους. Η κυρία Κέλλερ κατάφερε να γίνει και ευρωβουλευτής. Μα καλά δεν τρέπεστε. Εάν επιστρέψει ο φασισμός, δεν θα σας πει είμαι ο φασισμός, θα πει όχι εγώ είμαι ο αντιφασισμός. Αυτό το είχε προφητεύσει ο Ιγνάτσιο Σιλόνε ε, και αυτό κάνουν οι υποτιθέμενοι αντιφασίστες και οι αριστεροί δεν παίρνουν αποστάσεις αλλά εκφράζουν αλληλεγγύη με αυτούς τους τραμπούκους και με την άδειά σα αυτά είναι ικτρά πράγματα όποιος ε, θεωρεί την αριστερή βία κάτι το θεμητό ε, δεν θα πρέπει να εκπλήσεται ότι δεχόμαστε επιθέσεις με βόμβες εμείς όμως πάντα θα αγωνιζόμασταν οι αριστεροί να έχουν το δικαίωμα να λένε ό,τι μπαρούφα θέλουν ενώ οι αριστεροί θέλουν να μας φημώσουν και τους υποσχόμε ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρουν. Ευχαριστούμε. Και τώρα για την Ευρώπη τη Ελευθερία και τη Άμεση Δημοκρατία, συγγνώμη για την, των Εθνών και τη Ελευθερία, ο κύριο Μπέ. Ευχαριστώ. Ε, η συζήτησή μα έχει θέμα να καταπολεμήσουμε το κλίμα μίσου και σωματική βία κατά των ε, δημοκρατικών εκλεγμένων των λαδόχων. Είναι ένα θέμα που γνωρίζω καλά γιατί οι εκλεγμένοι του κομματό μου, του Ρασαμβλωμό Νασιονάλ και ακόμα και υποψήφοι και οι στρατευμένοι μα πολίτε, συναισθηματικά έχουν τύχει λιντσαρίσματο από τα μέσα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και παρενόχληση σωματική και ηθική δέχονται καθημερινά από τις ακροαριστερές ε, ομάδες. Είναι σαφέ ότι στη Γαλλία και τι περισσότερε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Δυτική Ευρώπη, οι περισσότεροι ουσιαστικά ε, χωρί να αμφισβητούνται ε, στηρίζουν τις κυβερνήσεις και ξερνάνε το μίσο τους ε, ονομάζοντάς τους λέκιστες, ε, προσπαθούν να εκφραστούν εμποδίζοντα κάθε δημοκρατική συζήτηση. Αυτό συνέβη και στην Γερμανία. Δεν άκουσα κανένα διαμαρτυρία ότι είναι συνάδελφο Φων Στόρχ. Ε, είδε το αυτοκίνητο τη να φλέγεται τον Οκτώβριο του 2015, όπω επίση και όταν ε, από την Ομοσπονδιακή Βουλή ο Φρανκ Μάγνιτ δέχτηκε δύο επίθεση. Και στη Βρέμιο ο κύριο Μάγνιτ ξυλοκοπήθηκε αγρίω και τον άφησαν σχεδόν νεκρό μια ομάδα από αριστερίζοντε και παραστατική ομάδα στην ουσία τη προαριστερά. Η ε, Βρετανική, η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει τα μέτρα της για να προστατεύσει και τα μέλη της ε, ΑΕΦΔ. Ε, θα πρέπει λοιπόν στο κύκλο αυτό να ε, σταματήσουμε να ακούμε όσους με συγχωρείτε αλλά ξεπεράσετε το χρόνο σας κύριε Μπέι. Οπότε τώρα θα περάσουμε στον επόμενο, τον κύριο Συναδεινό. Η ελευθερία του λόγου είναι επιβεβλημένη. Το μονοπόλιο στην άσκηση βίας θεσμικά το κατέχει αποκλειστικά η πολιτεία ω εντολοδόχοι οι κυβερνώντε οφείλουν να αντιληφθούν ότι τα λόγια και οι πράξει του μπορεί να οδηγήσουν του πολίτε σε ακραίε εκδηλώσει όταν προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. η εξουσία δεν ασκείται δίχω όρια ή έλεγχο. όσοι καλλιεργούν κλίμα μίσου βία και διχόνοια μεταξύ των πολιτών μοιραία θα δεχτούν αντίστοιχη συμπεριφορά ω ίσα μέλη τη κοινωνία. όπω τώρα στην ελλάδα που μια προδοτική μειοδοτική κυβέρνηση απαγορεύει τη χρήση του όρου μακεδονία η ιστορία παραχαράσεται, δημοτικά τραγούδια και ύμνοι λογοκρίνονται εκδηλώσει απαγορεύονται παιδαγωγοί διώκονται το δικαίωμα τη ελευθερία του λόγου και ο επί προσδιορισμό προσδιορισμός μας ως έλληνες μακεδόνες καταστέλλεται βιαίω. ό,τι σπέρνουν θερίζουν και θα ειδούν στο μέλλον χειρότερα. οι απλοί Έλληνε πατριώτε που ο τσίπρας διασύρισε ξένου ηγέτε ω λαϊκιστές και φασίστε δεν πρόκειται να συμβιβαστούν με την αντισυνταγματική αντιδημοκρατική και παράνομη συμφωνία των πρεσπών επομένως μην περιμένετε έστω και ένας έλληνας να τρέφει συμπάθεια σε πολιτικούς προδότες. τώρα δρέπουν την αντίδραση των πολιτών. η μακεδονία είναι γη ελλήνων και είναι ελληνική. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και ε, κανονικά ε, ε, δεν υπάρχει εδώ κατσιά. Ζητούν κάποιοι συνάδελφοι ε, δεν έχουμε ούτε μπλε κάρτε ούτε τίποτα. Ένας από κάθε πολιτική ομάδα και ένας μη Ε, σας ευχαριστώ κύριε ε, Επίτροπε για τη συζήτηση. Ολοκληρώνεται η συζήτηση και ε, προχωρούμε στο επόμενο θέμα και θέλω να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Φρανς Τίμερμανς, καθώς επίσης και την κυρία Υπουργό. Ε, δήλωση ε, Επιτροπής και Συμβουλίου για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία. Εξελίξεις από το Σεπτέμβριο του 2018 και μετά. Θα λάβει πρώτα το λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου η, η κυρία Μελάνια Τσότ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Κυρία Τσότ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ, κύριε Επίτροπε, οι κοινέ αξίε όπω η ανθρωπινή αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτο δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η η λύθη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα θεσμικά οργάνα αλλά και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σεβαστούν, να τι προστατεύσουν και να τι πρόθουν η Ρουμανική Προεδρία και όλοι μας συμφωνήσαμε ότι η προστασία του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ε, δικαιωμάτων είναι κάτι το θεμελιώδες για την Ένωση. Της 18 Ενάτου του 18 το Συμβούλιο έλαβε ε, την τεκμηριωμένη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγράφος 1 ε, καλούσε το Συμβούλιο να καθορίσει και να διερνήσει κατά πόσον υπάρχει παραβίαση ή κίνδυνο παραβίαση των θεμελιωδών αξιών από πλευρά τη Ουγγαρία και αυτό υποβλήθηκε τον Οκτώβριο, ε, Νοέμβριο και Δεκέμβριο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Στι 12 Ινδεκάτου το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων έλαβε από την ε, Ουγγαρία μια έγγραφη απάντηση στην αιτιολογημένη πρόταση του Κοινοβουλίου και επίσης μια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την εκκρεμούσα διαδικασία επί παραδιάση κατά της Ουγγαρίας. Τον Δεκέμβριο οι Υπουργοί για πρώτη φορά αντίλαξαν απόψεις όσον αφορά τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τη διαδικασία, εμείς θα συνεχίσουμε την μελέτη και εξέταση αυτή τη αιτιολογημένη προτάσεω του Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε, δεν μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα όσον αφορά την κατάληξη της διαδικασία. Θα σα ενημερώνουμε όσον αφορά τις ε, εξελίξεις μια που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο προβληματισμός των ε, βουλευτών του Κοινοβουλίου και είναι κατακλείδη έχω να σας πω ότι τα θέματα τα οποία θέσατε κατά αυτήν την συζήτηση είναι κάτι κομβικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη δική μας προσφύλωση σε αυτές τις οπότε θεωρούμε ότι όλες οι πλευρές θα αντιδράσουν υπεύθυνα τόσο ώστε να υπάρξει μια κατάληξη αυτή τη διαδρομής σύμφωνη με τις ε, βασικές μας αξίες και σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κυρία... Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που μας παρουσιάσετε τη θέση του Συμβουλίου και τώρα ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Τίμερμαν. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που προέβλεψε την κατάσταση της Ουγγαρίας σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Η τελευταία φορά που συζητήσαμε την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία ήταν στις 11 Σεπτεμβρίου πέρσι. Την επόμενη μέρα το Κοινοβούλιο ανέκρινε το ψήφισμά του που ενεργοποιήσε το άρθρο 7.1 της συνθήκης και της σχετικής διαδικασίας κατά της Ουγγαρίας. Όπως έχω εξηγήσει και τότε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου όπως εκφράζονται στην ε, πρόταση που έχουμε μπροστά μας, ιδίως για τα θεμελούδη δικαιώματα, ε, την προστασία του, τη μεταχείριση των Ρωμά και την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου. Ναι. Σήμερα θα ήθελα να σα ενημερώσω για τι πρόσφατε εξελίξει που έχουν λάβει χώρα από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μεταξύ των οποίων των αποφάσεων του Συμβουλίου. Πρώτον, όπω έχω πει και το Σεπτέμβριο, σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει τη συνθήκη, έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραβάση και στην περίπτωση τη Ουγγαρία έχει ξεκινήσει πολλέ διαδικασίε παραβάσει που έχουν σχέση με θέματα τη αξία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο την διαδικασία αυτή. Την περασμένη εβδομάδα στείλαμε μία επιστολή ε, σε σχέση με την νομοθεσία στο Ψόρο, η οποία επιβάλλει κυρώσει για διαδικασίε και αναστέλει αιτήσει ασύλου και αιτήσει διεθνού προστασία από οποιοδήποτε είναι ύποπτη. Οι εγκρικέ αρχέ έχουν τώρα δύο μήνε να απαντήσουν στι τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Επιτροπή. Επιπλέον, τον περασμένο Δεκέμβριο, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νέο νόμο που ε, αναθεωρεί το εργατικό δίκαιο. Όπω ξέρετε, ο νέο αυτό νόμο έχει προκαλέσει έντονε διαδηλώσει στου δρόμου τη χώρα τι τελευταίε εβδομάδε. Αναλύσαμε την ε, συμβατότητα του νέου αυτού νόμου με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ιδίω την ε, οδηγία για το χρόνο εργασία και αποστήλαμε σχετική επιστολή στι Ουγγρικέ Αρχέ. Βάσει τη απάντηση που θα λάβουμε, θα αποφασίσουμε για τα ενδεχόμενα μελλοντικά βήματα. Επίσης το Δεκέμβριο ακούσαμε ότι το Πανεπιστήμιο αν τη Κεντρική Ευρώπη αναγκάστηκε να μετακινήσει την έδρα του από την ε, Ουγγαρία στην Βιέννη. Το να έχουμε ένα πανεπιστήμιο που εξαναγκάζεται να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω κυβερνητικών μέτρων και συστηματική πίεση είναι άνευ προηγουμένου στην ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι θλιβερό και πολύ ανησυχητικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά την διαδικασία που παραβάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι σαφεί προειδοποιήσει από πολλού ενδιαφερομένου και εταίρου. Ε, μια τελευταία εξέλιξη του Δεκεμβρίου είναι η συγχώνευση 400 σταθμών μέσων μαζική ενημέρωση ε, που ελέγχονται από, από το κόμμα που είναι φιλεπροσκευμένο στην κυβέρνηση. Αυτό σχετίζεται και με την κυβερνητική απόφαση να εξαιρέσει την συγχώνευση αυτή από από, την, από τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής για τον ανταγωνισμό της χώρας και τον νόμο για τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμενού εξετάσαμε και τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος στην Ουγγαρία, όπως την πρόθεση για τον τηρισμό των δικαστών, το πώς είναι οργανωμένη η εισαγγελία, και ε, το αν θα δημιουργηθούν νέα ε, δικαστήρια διοικητικού χαρακτήρα. Πέρσι τον ε, Δεκέμβριο το Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο νόμους για την δημιουργία, την ίδρυση διοικητικών δικαστηρίων που θα αρχίσουν να λειτουργούν από το 2020. Είναι θλιβερό. Περιμένουμε τον Μάρτιο φέτος την έκθεση της Επιτροπής της Βενετίας για να δούμε τη συμβατότητα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας θα τροφοδοτήσει την τελική μας αξιολόγηση. Επιπλέον από τη διαδικασία υπεραβάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί και άλλα μέσα, ελέγχους, έρευνες που έχουν να κάνουν με τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της ε, τήσιας διαδικασίας ε, δημοσιονομικών. Ε, εκτιμούμε επίσης και τις συστάσεις προς την Ουγγαρία για να δούμε κατά πόσο καταπολεμείται η διαφθορά. Οι προσπάθειες για τη διαφάνεια, για τον ανταγωνισμό, για τις δημόσιες συμβάσεις. Όσον αφορά τη διαδικασία του άρθρου 7 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυστυχώ δεν έχει δώσει την ευκαιρία προς το παρόν ε, να περάσουν οι προτάσεις του στο Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι όποια και αν είναι η θέση τελικά του Συμβουλίου θα πρέπει να υπάρχει επεξεργασία της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πλήρως. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος και πρέπει να σέβονται αυτή τη διαδικασία όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θέλω να σα πληροφορήσω ότι τον Νοέμβριο, μετά από αίτημα τη Αυστριακή Προεδρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στο Συμβούλιο μία επισκόπηση γεγονότων και δράσεων που έχει αναλάβει σε σχέση με την διαδικασία επιπαραβάση. Άσυλο, ε, βοήθεια προς τους ετούντες άσυλο, ανώτατη εκπαίδευση διακρίσεις σε βάρος στο Ρώμα. Οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις εκκρεμούν ακόμα στο δικαστήριο. Όπως γνωρίζετε, η εγκρική κυβέρνηση ήδη απάντησε στην αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο τώρα έχει όλα τα στοιχεία στη διάθεσή του προκειμένου να αρχίσει τη δικιά του αξιολόγηση των θεμάτων αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριο Τόμας Ντόιτς, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Γιατί η φιλελεύθερη πλειοψηφία για άλλη μια φορά βάζει το θέμα της Ουγγαρίας στην ημερήσια διάταξη έτσι για να ακουστούν κάποιες ομιλίες ή γιατί με απελπισία προσπαθούν να τα βάλουν με την Ουγγαρία. Στην πραγματικότητα ο λόγος είναι ότι έρχονται ευρωεκλογέ. και η αριστερή πτέρυγα, ε, οι φιλελεύθεροι θέλουν να τα βάλουν με την Ουγγαρία. Γιατί συμβαίνει αυτό όμως. Το γιατί συμβαίνει αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ουγγαρία. Ουσιαστικά οι περισσότεροι στην Ουγγαρία συμφωνούν, ανεξάρτητα από ποιο κόμμα προέρχονται, ότι δεν θέλουν τη μετανάστευση. Οι περισσότεροι όμως εδώ θέλετε να στηρίξετε τη μετανάστευση. Πιστεύετε ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα και θέλετε να νομιμοποιήσετε την παράνομη μετανάστευση. Θέλετε να σώσετε τα διάφορα προβλήματα και να τα λύσετε που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη μέσω από την παράνομη μετανάστευση θέλετε να αφαιρέσετε από τις χώρες μέλη το δικαίωμα που έχουν να προστατεύουν τα σύνορά τους ή για τις αποφάσεις τους σε σχέση με τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις. Ε, θέλετε, όπως και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, να εγκατασταθούν οι μετανάστες. Θέλετε εσείς να μας υπαγορεύετε πού θα εγκατασταθούν οι μετανάστες αυτοί. Θέλετε να μας τιμωρήσετε. Και ο κόσμος στην Ουγγαρία λέει όχι στη μετανάστευση. Εμείς όμως θα προστατεύσουμε τα σύνορά μας απέναντι στη μετανάστευση και με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ε, δεν θέλουμε να εισαχθεί το πρόβλημα στην Ευρώπη. Θέλουμε να εξαχθεί βοήθεια έξω από την Ευρώπη προς τις χώρες αυτές. Αυτό ζητούν οι Ουγγροί πολίτες. Γι' αυτό το λόγο εσεί έχετε πρόβλημα μαζί μα. Τέσσερι ε, μήνε πριν από τι εκλογέ δεν εξυπηρετεί κανέναν απολύτως να επιτίθεστε κατά της Ουγγαρίας. Οι Ούγγροι θα ψηφίσουν ώστε η Ευρώπη να αντιληφθεί επιτέλους το αυτό που πρέπει. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ. Κύριε Πρόεδρε, με την εισαγωγή της διαδικασία κατά της Ουγγαρία έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σημαντική ιστορική απόφαση την οποία λάβαμε δύσκολα, όμως μας επέκριναν πολύ διότι χρειαστήκαμε τόσο πολύ χρόνο. Ήταν αναγκαίο όμω αυτό διότι χρειάστηκε να συγκεντρώσουμε προσεκτικά όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και βεβαίω να τι ζυγίσουμε υπεύθυνα. Το Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο ψήφισε την έκθεση με σημαντική πλειοψηφία θα έπρεπε να περιμένει κανείς ότι μετά από αυτό θα ακολουθούσε μια κατάλληλη αντίδραση από πλευρά του Συμβουλίου Υπουργών και από πλευρά Ουγγαρία. Τίποτε τέτοιο δεν συνέβη. Η Ουγγρική κυβέρνηση, η οποία πριν δεν άφηνε καμία ευκαιρία που να μην εκμεταλλευτεί για να εμπλακεί στη διαδικασία, τώρα απεφάσισε να γνωρίσει το Κοινοβούλιο. Και η απουσία της σήμερα δείχνει την περιφρόνησή της προς το Κοινοβούλιο θεώρησε ότι δεν είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη τις αμφιβολίες, τις, ε, την, τις επιφυλάξεις των Ευρωπαίων φίλων της. Γιατί είμαστε φίλοι της. Η Ουγγαρία γίνεται όλο και περισσότερο μια δημοκρατία βιτρίνας. Δεσμεύει τα δικαστήρια, δεν επιτρέπει στις μη κρατικέ οργανώσεις να λειτουργούν. Η πανεπιστημιακή ελευθερία βρίσκεται σε κίνδυνο και την πολιτική ανάλυση αντικαθιστούν πλέον θεωρίες συνωμοσία. Είναι εκπληκτικό το ότι το Συμβούλιο Υπουργών εξακολουθεί να μην λαμβάνει μέτρα για να ακολουθήσει αυτά που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εξελίξεις, τις εξελίξεις τις λαμβάνει υπόψη σιωπηρά. Αυτό σημαίνει όμως ότι εγκαταλείπει την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ελπίζω η Προεδρία του Συμβουλίου να μην καθυστερήσει περισσότερο για να λάβει τις τα αναγκαία μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Βάιντεν Χόλτσερ. Θα δώσω τον λόγο τώρα στον κύριο Βίστισεν, εξ ονόματος της ομάδας συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Πάλι το Κοινοβούλιο ξεσπάει κατά της Ουγγαρίας για θέματα κράτους δικαίου και δημοκρατίας το ίδιο σώμα το οποίο πρότεινε να στερηθούν το δικαίωμα ταξιδιού άνθρωποι με του οποίου διαφωνεί. Το ίδιο σώμα το οποίο εδώ στην Ολομέλεια πρόκειται να υπερψηφίσει τροπολογίες για τα άρθρα του κανονισμού τα οποία στρέφονται κατά των απόψεων της μειοψηφίας στο ίδιο το Κοινοβούλιο. Αν δεν βλέπει κανείς αυτήν την υποκρισία, τότε σημαίνει ότι έχει μείνει υπερβολικά πολύ μεγάλο διάστημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν γνωρίζω το ακριβέ περιεχόμενο των κατηγοριών κατά πίεση των Αυτό που γνωρίζω ωστόσο είναι ότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση των κρατών μελών. Βλέπουμε καταπίεση των διαδηλωτών στην Καταλωνία, βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, αλλά δεν βλέπουμε καμιά αντίδραση εδώ. Όταν υπάρχει καταστολή διαδηλώσεων στη Βουδαπέστη, προφανώ για το Κοινοβούλιο αυτό είναι παράβαση του κράτου δικαίου. Βρίσκω ότι είναι θεμελιωδώς προβληματικό. Ξεκινώντα από τον Γιώργ Χάιντερ στην Αυστρία πριν από 10 χρόνια μέχρι τι επιθέσει σήμερα κατά Ουγγαρία και Πολωνία που ξεκινούν πάντοτε από το ευρωπαϊκό κατεστημένο. Και είναι βαθύτατα ενοχλητικό το γεγονό ότι εσεί εδώ δεν βλέπετε ότι το μόνο που κάνετε είναι να προκαλείτε ακόμα περισσότερη υποστήριξη για αυτούς που θέλετε να εξαφανίστε, όπως τους Κατσίνσκι, Όρμπαν και λοιπούς. Και τους οποίους έχουν εκλέξει δημοκρατικά οι ευρωπαϊκοί λαοί. Τροπή για την Ευρώπη και τροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και τώρα η Judith της Αργεντίνη τους Πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να καταλήξουμε ότι από την ε, ψηφοφορία της έκθεσής μου ε, το Σεπτέμβριο τα, τα πράγματα στην Ουγγαρία επιδεινώθηκαν. Οι Ούγγροι πολίτες έχουν κάθε λόγο να κατεβαίνουν στους δρόμους και πρέπει να τους δείξουμε αλληλεγγύη. Θα ήθελα να σας απαριθμίσω μερικές από τις εξελίξεις του φθινοπόρου. Ο κύριος Τίμερμανς επίσης αναφέρθηκε σε αυτά. Το Κεντρικό Πανεπιστήμιο αναγκάστηκε να πάει στη Βιέννη γιατί η συμφωνία με... που, έχει υπογραφεί, που είχε συμφωνηθεί δεν θα υπογραφεί. Ε, ένα διοικητικό δικαστήριο δημιουργείται και το Υπουργείο Δικαιοσύνη είναι το αρμόδιο γι' αυτό. Ο πρώην Υπουργό τη Μακεδονία ε, που έχει καταδικαστεί για διαφθορά ε, προστατεύεται. 450 ΜΜΕ δημιούργησαν έναν όμιλο, ένα ενιαίο όμιλο με βάση νόμο. Επίσης, κάποια πράγματα που όλοι ξέρουμε, ότι οι Ούγγροι ε, χρονοτριβούν. Υποτίθεται ότι συνεργάζονται, μας κατακλείζουν με χαρτούρα, αλλά θέλουν να κερδίσουν χρόνο. Αυτό δεν μας εκπλήξει. Το γεγονός όμως ότι η, τα αιτήματα της Ρουμανικής ε, Προεδρίας να υπάρξει μόρφωση με το χρονοδιάγραμμα είναι σαφές. Οι Ούγγροι πολίτε έχουν το δικαίωμα προστασία και πρέπει να ξέρουν ε, τι σκοπεύετε να κάνετε. Οι Ευρωπαίοι πολίτε πρέπει να ξέρουν τι θα κάνετε ε, και τι θα κάνουν οι πολιτικοί ηγέτε. Σα ρωτάω λοιπόν να λάβετε ευθύνη, να, καλ... με καλέσετε στο Συμβούλιο και να αρχίσετε μια σοβαρή διαδικασία. Προς τους συναδέλφους ε, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ορισμένοι από εσάς είσαστε εδώ και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά οι περισσότεροι δεν είστε. Συνεχίζω να σα εκτιμώ εσά που υπερψηφίσατε την έκθεσή μου. Αλλά έκτοτε τι κάνατε. Πού βρίσκονται οι ευθύνε σα, τι έχετε αναλάβει. Κυρία Σαρτζεντίνη, τέλειωσε ο χρόνος σας. Μάλιστα και τώρα η κυρία Βεργιά έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η Ουγγαρία είναι θαυμάσια χώρα, ε, ένα αμάλγαμα πολιτισμών. Ε, το σύμβολό της είναι η Βουλγαρία. Κανείς δεν θέλει να επιτεθεί στους Ουγγρούς πολίτες. Αλλά ο δικτάτορας Ορμπάν θέλει να γίνει πρωταθλητής ενός ε, νέου μοντέλου εθνικιστικού και κατά των μεταναστών. Είναι κρίμα για την ιστορία αυτής της όμορφης χώρας και της υπήρου μας. Από το Σεπτέμβριο ε, έχουμε τεράστιες διολυστήσεις. Ε, διοικητικά δικαστήρια, ΜΜΕ που υπο... Ε, και δικαστήρια που υποτίθεται κρίνουν δημόσια πράγματα είναι υπό έλεγχο. μεγάλη διαφθορά. Η Ουγγαρία δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. μία νέα αυταρχική δι... ε, εισαγγελική διοίκηση δημιουργείται υπό τον Ορμπάν. Ε, υπάρχει ο νόμος για τα εργατικά, νόμος της σκλαβιάς όπως λέγεται, ο κύριος Τίμερμα, κύριε Τίμερμα, μάλλον τα ιδιολεστήσει ε, ξεκίνησε το 2010, παρακολουθείτε υποτίθεται τα πράγματα, εξετάζετε ποια είναι τα δικαιώματα. Δεν υπάρχει πόλεμος, λέω, στους Ούγγρους. Το θέμα των ε, μεταναστών είναι ε, ένα υποπροϊόν. Το βασικό είναι να σεβαστούμε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, όντως, χρονοτριβεί η Ουγγαρία πίσω από διαδικαστικά ε, έτσι, διαδικασίες, αλλά είναι προβληματική κατάσταση. Όλαφ Στούγκερ τώρα από, την, ε, από το ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στην Ολλανδία το 2014 37% ήταν η συμμετοχή στις εκλογές. Στην Ουγγαρία ήταν 70% για τις ε, εθνικές εκλογές και βγήκε ο Ορμπάν. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διαφορά στα ποσοστά με τα οποία ήρθαν εδώ οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ούτε καν στον ύπνο τους δεν βλέπουν τα ποσοστά της Ουγγαρίας. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Καθόμαστε και κάνουμε ψηφίσματα και ασχολιόμαστε με το Περού, τις εγκυμοσύνες, εκείνο και τα λοιπά. Μα δεν είναι σοβαρό αυτό. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να ενδιαφέρουν. Και αυτό ακριβώς κάνει και ο Ορμπάν. Ασχολείται με την ασφάλεια στη χώρα του και φροντίζει για τους ανθρώπους του. Και αυτή είναι η διαφορά. Ένας Πρωθυπουργό ο οποίος ασχολείται με τον λαό του. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται σε τέτοιες ε, διαδικασίες δικαστικές εις βάρος του. Άγαλμα θα έπρεπε να του είχαμε κάνει. Ας φροντίσουμε λοιπόν να υπάρξει πρόβλεψη για τέτοιο κονδύλι στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Παλτζότορ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Γίνεται αγώνας στη χώρα μου κατά της, δια, της διαφθοράς και γι' αυτό ξεκινούν αυτά τα κηρύγματα μίσους. Είμαι πεπισμένος ότι αυτός ο πολιτικός αγώνας δεν μπορεί να συνεχιστεί εδώ στις Βρυξέλλες. Ο πολιτικός αγώνας πρέπει να γίνει στην Ουγγαρία μαζί με τους Ούγγρους πολίτες και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε συνταγματικό μέσο για να ανατρέψουμε το καθεστώς Όρμπαν. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Τώρα η κυρία Κούντριτσκα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ο νόμος είναι το μόνο μέσο που επιτρέπει σε ένα τόσο ποικιλόμορφο περιβάλλον όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί. Όπως έλεγε η κυρία Στούσερ, είναι ακριβώς αυτό ο σεβιβασμός δηλαδή η ψυχή της δημοκρατίας. Αν όμως εμείς υπονομεύουμε τον νόμο και τις ευρωπαϊκές αξίες και αν δημιουργούμε έναν εναλλακτικό κόσμο προκειμένου να φέρουμε σε πέρα τους στόχους του δικού μας κόμματος, τότε έχουμε φτάσει στο τέλος της δημοκρατίας. Στην αρχή του τέλους. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι Ουγγαροί συνάδελφοι δεν μπορούν να πείσουν τον ηγέτη τους ότι θα έπρεπε να προσπαθήσει να καταλήξει σε έναν συμβιβασμό και να υπάρξουν και πάλι οι βασικές αξίες της δημοκρατίας στην Ουγγαρία. Και έχω και μια ερώτηση. Δεν βλέπετε ότι δεν υπάρχει συμβιβασμός αντίθετα, υπάρχει κλιμάκωση της κατάστασης στην Ουγγαρία. Για παράδειγμα με την νομοθεσία για τα εργασιακά, το λεγόμενο νόμο της δουλείας ή ε, υποχρεώνοντας το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης να φύγει από τη χώρα. Είναι κοινικά αυτά, μα κάποιοι συνάδελφοι θα έπρεπε να έχουν δισταγμούς για όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Σάνι τώρα εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ε, ε, ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Προ τριακονταετίας έγινε μια σημαντική αλλαγή στην Ουγγαρία. Άνθρωποι που τότε είχαν συμβάλει στην αλλαγή αυτή είναι σήμερα ηλικιωμένοι, εύποροι και στην ουσία θεοδάρχες είχαν εκμεταλλευτεί το σοβιετικό σύστημα και τώρα, σήμερα δηλαδή, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχει, μιλούμε για μια χώρα φτωχοποιημένη. Οι άνθρωποι στερούνται τα δικαιώματά τους, η γνώση έχει απαξιωθεί, η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς. Οι εκπρόσωποι της εξουσίας και γενικότερα όλοι αυτοί που κυκλοφορούν με σωματοφύλακες εκπροσωπούν το έθνος. Μιλούν για πράκτορες, για πράκτορες του όρου, προσπαθούν να τους ανατρέψουν. Αυτά είναι τα νέα από την χώρα μου, τη νέα χώρα της δουλείας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Ο Βίκτορ Όρμπαν δεν θέλησε να έλθει στην ε, συζήτηση, να προσέλθει στη συζήτηση. Έχει τα δικά του αυτός. Θα πρέπει ωστόσο, γιατί θα χρειαζόταν τότε να προβάλλει επιχειρήματα αν ερχόταν δηλαδή. Εγώ τον ρωτώ τον Όρμπαν λοιπόν από εδώ. Τι είναι σημαντικότερο από του να συζητήσει με ποιον τρόπο μεταχειρίζεται και αντιμετωπίζει τις ευρωπαϊκές αξίες. Τι είναι πιο σημαντικό από το να συζητήσει ότι εδώ και εννέα χρόνια υπονομεύει τα δικαιώματα των Ούγγρων πολιτών στην Ουγγαρία. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα χρόνια αυτά. Έχει επιδεινωθεί σημαντικά στην Ουγγαρία. Συμβαίνουν πράγματα απαράδεκτα. Πρόκειται για ένα αυταρχικό σύστημα το οποίο έχει χαρακτηριστικά συστήματος Πούτιν. Τι πρέπει να γίνει επιτέλους ώστε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την κατάσταση αυτή και να αντιληφθούν ποιο είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αυτήν. Η κυρία Μπιόρκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση δεν βελτιώνεται στην Ουγγαρία, αλλά βλέπουμε ότι ο Ορμπάν πιέζει περισσότερο όσους σκέφτονται διαφορετικά, είτε είναι ακαδημαϊκοί, είτε είναι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, είτε άνθρωποι που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των μεταναστών. Αλλά βλέπουμε ότι η αντίσταση στην κυβέρνηση επίσης ενισχύεται. Πολλοί στις χώρες μας, αλλά και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το βλέπουμε αυτό και προσπαθούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Το Φιντές λέει ότι εγώ και άλλοι συνάδελφοι εδώ είμαστε εχθροί. Είμαστε αντίπαλοι, όπω και όσοι πιστεύουν σαν και εμάς στην Ουγγαρία. Αλλά κύριε Ορμπάν, όχι, δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε. Θέλουμε σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου, δεν θέλουμε τα δικά σα σχέδια εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίσουμε να υψώνουμε τη φωνή μα και να μιλάμε για τι ελευθερίε, για τα δικαιώματα των γυναικών, των μεταναστών και πράγματι θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τι ευρωεκλογέ τι επερχόμενε. Βεβαίω, και εδώ θα στηρίζουμε πάντα τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Ναι, θα είναι ένα θεμελιώδε ζήτημα, βασικότατο για τι ευρωεκλογέ, γιατί τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Μορβάη τώρα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την κυρία Σαρζεντίνη. Αλλά κυρία Σαρζεντίνη, για κοιτάξτε στην αίθουσα τι συμβαίνει, στην αίθουσα του Εμικυκλίου. Γνωρίζετε ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι 751. Ε, πάνω από μία δωδεκάδα δεν είναι παρόντα σήμερα και οι περισσότεροι είναι Ούγγροι. Βεβαίω τα πρόσωπα αυτά είναι εδώ, διότι η συζήτηση στρέφεται γύρω από την Ουγγαρία. Κατανοήστε επιτέλου ότι κανεί δεν ενδιαφέρεται για τον αγώνα που διεξάγεται κατά τη Ουγγαρία. Κοιτάξτε, κυρία μου, τελείωσε ο αγώνα. Χάσατε. Ψάξτε να βρείτε κάποιο άλλο πράγμα να ασχοληθείτε. Και επειδή σα ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, και εγώ άλλωστε ασχολούμαι με ανθρώπινα δικαιώματα, σα συνιστώ να κοιτάξετε με πιο βάρβαρο τρόπο καταστέλει η αστυνομία στην Γαλλία τις διαδηλώσεις. Δηλαδή γίνονται τα ίδια πράγματα όπως τότε παρημείνει στην Ουγγαρία πριν από το 2010. Άνθρωποι που έχουν χάσει την όρασή τους, έχουν υποστεί βαρύς τραυματισμούς στο κεφάλι και αυτά από τον αγαπημένο σας πολιτικό. Για ανθρώπους οι οποίοι ζητούν απλώς τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Να ασχοληθείτε και με αυτόν, κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι περισσότερα τα πρόσωπα που είναι παρόντα από αυτό που είπε η συνάδελφος. Κύριε Πρόεδρε, η κυρία Γκρέσλε, βρίσκομαι εδώ διότι ανησυχώ για λογαριασμό τη ε, επιτροπή Ελέγχου προπολογισμού με το τι συμβαίνει με τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ουγγαρία. Εμεί θεωρούσαμε ότι θα αυξηθεί το εισόδημα στη χώρα αυτή και θα μειωθούν οι άνεργοι. Δεν μπορούμε ωστόσο, το βλέπουμε αυτό, να προστατεύσουμε τα ε, ευρωπαϊκά κονδύλια όπως θα θέλαμε. Υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς και υπάρχει πρόβλημα με δικαστικές αρχές οι οποίες δεν διώκουν ή δεν τους επιτρέπεται να διώκουν σχετικά εγκλήματα, ίσως διότι προστατεύουν κάποιους. Οι δημοσιονομικοί ελεγκτές έχουν άλλωστε πρόβλημα, διότι η Ουγγρική κυβέρνηση δεν λαμβάνει απολύτω κανένα μέτρο για την καταστολή των περιπτώσεων αυτών. Κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, σα παρακαλώ φροντίστε ώστε να αρχίσει σύντομα τριμερή διάλογο όταν θα έχουμε τον σχετικό κανονισμό, διότι ο μετρητής διαφθοράς δείχνει την Ουγγαρία στον αριθμό 64, αμέσως μετά την Ελλάδα. Όμως στην Ελλάδα ο δείκτης ε, κοιτάζει προς τα πάνω, δηλαδή τα πράγματα βελτιώνονται, ενώ στην Ουγγαρία όχι. Είμαι βεβαία ότι η Ουγγαρία μπορεί να τα καταφέρει και καλύτερα και θα ήταν πραγματικά ένα σημαντικό βήμα αποκατάσταση εμπιστοσύνη εάν αποφάσιζε η Ουγγαρία να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αγαπητέ Αντιπρόεδρε, κύριε Τίμερμαν, παρακαλώ να τα λάβετε σοβαρά υπόψη σα τα πράγματα αυτά. Σα ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ. Κύριε Γκρέσλε. Ο κύριος Νίντερ Ευχαριστώ. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός δήλωσε ότι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται μια συνεδρίαση σώρος και ότι πρόκειται για πολιτική φάρσα. Αυτά λέει η Ουγγρική κυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο βλέπει η Ουγγρική κυβέρνηση την δημοκρατία. Ο Ούγγρο Πρωθυπουργό βεβαίω δεν είναι παρόν σήμερα εδώ, δεν θέλει να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι φοβάται τη δημοκρατία και φοβάται το δημοκρατικό διάλογο. Γι' αυτό και κατήργησε την ελευθερία του τύπου, υπονομεύει την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη, δεν λαμβάνει μέτρα κατά τη διαφθορά, η οποία έχει φτάσει και μέχρι τη δική του οικογένεια. Δυσχεραίνει το έργο των οργανώσεων των δικαστών και προσπαθεί να στρέψει την χώρα προς δικτατορικέ κατευθύνσει. Δεν έρχεται στη Βραζιλία, πάει όμω. Δεν, δεν έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έρχεται εδώ στι Βρυξέλλε, πηγαίνει όμω στη Βραζιλία ή στη Ρωσία. Και προδίδει έτσι τα συμφέροντα τη ίδια του τη χώρα. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την πολιτική αυτή. Οφείλουμε να πούμε ευθαρσώ ότι αυτού του είδου η πολιτική δεν μπορεί να γίνει ανεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος Χάντσεν τώρα. Ευχαριστώ. Αν ε, σήμερα ήταν να μπει η Ευρωπαϊκή, η Ουγγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πληρώσει τα κριτήρια ένταξης. Ε, ποινικοποιεί ε, δεν δέχεται πρόσφυγες και ποινικοποιεί αυτούς που δέχονται ε, ε, τούντες άσυλο. Ε, εν τω μεταξύ κάποιοι άλλοι ε, λαμβάνουν την ε, ηθαγένεια όπως ο Ε, κυρίες και κύριοι, στον κατάλογο των ανθρωπίνων αξιών, ξέρετε πολύ καλά ότι οι Ούγγροι βρίσκονται πολύ χαμηλά γιατί υπάρχει τεράστια διαφθορά, όπως είπε η κυρία Σαρτζεντίνη και άλλοι. Ε, ζητήσαμε να σεβαστεί το κράτος δικαίου, αλλά εις μάτιν. Ε, η μείωση των πληρωμών προς τα κράτη τα οποία δεν σέβονται το κράτος δικαίου είναι σωστό ε, θέλω να πω στο Συμβούλιο πόσο πρέπει να περιμένουμε για να δράσετε, για να ενεργοποιηθεί το άρθρο 7. Θα πρέπει ε, να μην δείξουμε στενοχή ε, στην προσπάθεια ανατροπής του κράτους δικαίου. Ο Κάρλος Κοέγιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς και αγορά έχει κοινέ αξίες, αξίες που υπάρχουν και στην Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στις συνθήκες. Όταν μιλήσαμε για τελευταία φορά για την Ουγγαρία, από τότε μέχρι σήμερα, εθνικοποίησε διάφορα ε, περιοδικά εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις ε, και αντιμετωπίζει με απάνθρωπο τρόπο τους πρόσφυγες. Η κυβέρνηση, ο πρόεδρος διακόπτη γιατί υπάρχει πρόβλημα διερμηνίας ε, στα αγγλικά και στα πολωνικά. Και τώρα συνεχίζει ο κ. Σκουέγιο. Αποκαταστάθηκε το θέμα της διερμηνίας. Μήπως να ξαναρχίσω την παρέμβασή μου. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Να συνεχίσετε από εκεί που είχατε σταματήσει. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ξαναρχίσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο κοινή αγορά. Έχει κοινέ αξίε, οι οποίε ε, σφραγίζονται και στην ε, χάρτα και στι συνθήκε. Από το Σεπτέμβριο, που μιλήσαμε τελευταία φορά, για τελευταία φορά για την Ουγγαρία, εθνικοποίησε η Ουγγρική κυβέρνηση τι περισσότερε ε, εφημερίδε, περιοδικά, ραδιόφωνα. Έκλεισε ένα πανεπιστήμιο ε, φημώνει την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζει απάνθρωπα τους πρόσφυγες. Η κυβέρνηση ε, δημιουργεί κίνδυνο για το κράτος δικαίου ε, εις βάρος των Ούγγρων πολιτών και όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι μια κακή περίπτωση ο Ορμπάν και υπάρχουν και άλλες χώρες, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Μάλτα που πρέπει να μας ανησυχήσουν και απασχολήσουν. Πρέπει να αντιδράσουμε, Πρόεδρε, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο ελέγχου που θα αντιμετωπίζει ε, θέματα τέτοιες ε, χώρες που δεν σέβονται τις, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να σεβόμαστε τις θεμελιώδεις αξίες και θα πρέπει να πετύσουμε από το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 όπως προβλέπει η συνθήκη. Ελευθερία, δημοκρατία, κράτος δικαίου. Αυτές δεν είναι ηχηρές λέξεις για να ξεκινάμε δεκάρικους λόγους. Είναι κομμάτια της ταυτότητάς μας η οποία απειλείται Γι' αυτό ας έχουμε την, το κουράγιο να την υπερασπιστούμε. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για το πρόβλημα που υπήρχε και σας διέκοψα. Η κυρία Κίνγκα Γκάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, η κυρία Γκάλ. Όταν άκουσα τα όσα δήλωσε ο κύριος Νίντερ Μιούλερ, σκέφτηκα ότι είναι μάλλον αδιάφορο το τι κάνουμε αφού δεν είναι παρόν ο Όγκρος Πρωθυπουργό. Είναι όμως αυτό το πρόβλημα. Εγώ το βρίσκω γελίο. Όλοι και όλες γνωρίζουμε εδώ ότι η δράση αυτή είναι υποκειμενική και όχι αντικειμενική. Διότι αν αναλύσουμε τα πράγματα λεπτομερώς θα έπρεπε να στραφούμε κατά όλων των χωρών μελών Γνωρίζουμε ότι στην Ουγγαρία δεν έχουν κρατικοποιηθεί μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν κλείσει πανεπιστήμια. Τα πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών στο Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο εξακολουθούν να λειτουργούν. Πρόκειται για φάρσα δηλαδή αυτή η συζήτηση εδώ. Όλοι στρέφονται κατά της Ουγγαρίας, ενώ όλη αυτή η συζήτηση είναι μια αστεία παραγωγή τα νήματα της οποίας κινούν κοινή αριστερά. Και όσοι είναι υπέρ της μετανάστευσης στρέφονται κατά της Ουγγαρίας η οποία είναι αντίθετη με την υποδοχή μεταναστών. Η η κυρία Σαρτζεντίνη είπε ότι οι Ούγγροι πολίτες πρέπει να έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι και οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Ούγγροι πολίτες έχουν το δικαίωμα να τους αφήσει στη ησυχία τους η κυρία Σαρτζεντίνη. Προχωρούμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για άλλο ένα παράδειγμα τη χρήση διπλών μέτρων και σταθμών απέναντι σε ορισμένε χώρε μέλη. Το βλέπουμε αυτό διαρκώ. επικρίνουν την Ουγγαρία για πράγματα τα οποία συμβαίνουν και σε άλλες χώρες μέλη και με τον ίδιο τρόπο. Όπως ο νόμος για τις υπερορίες ή η δικαιοδοσία των δικαστηρίων. Συχνά όμως ενημερώνουν με σφαλμένο τρόπο την κοινή γνώμη ή με υπερβολές ή κυκλοφορούν τα λεγόμενα fake news, οι ψευδείς ειδήσει. Δεν βοηθεί κανένα να διεξάγουμε τέτοιες απεραντοεπείς συζητήσεις γιατί δεν πάμε να δούμε τι γίνεται με τους Ούγγρους φοιτητέ, οι οποίοι δεν μπορούν τώρα να δώσουν εξετάσεις. Εδώ όμως διακυβεύεται η αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και δεν είναι δυνατόν να επικρίνεται διαρκώς η ίδια χώρα. Χουάν Λόπε Αγγιλάρη είναι ο επόμενο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμαντ. Για πρώτη φορά στην ιστορία, μετά τη Λισαβόνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε με τα δύο τρίτα πλειοψηφία στην πρωτοβουλία να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφο 1 σε σχέση με την Ουγγαρία. Και αυτό γιατί αυτά τα οποία περιγράφονται που κάνει ο Ορμπάν είναι μια κατάχρηση εξουσίας εντελώς ασύμβατη με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του, του κατά των μειονοτήτων, περιορισμός της ελευθερίας ε, ενημέρωσης αλλά και της ακαδημαϊκής ε, ελευθερίας. Και τα πράγματα χειροτερεύουν. Οπότε κύριε Τίμερμαντς, εγώ αυτό που θέλω είναι όταν αποφασίζει το Συμβούλιο παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συζητάει για τις συνέπειες μετά από την ψηφοφορία που με πλειοψηφία που σας είπα στα δύο τρίτα εγκρίθηκε ενεργοποίηση του άρθρου 7 θα έπρεπε τα τρία θεσμικά όργανα να ενώσουν τη φωνή τους και να πούνε φτάνει πια η κατάχρηση αυτή από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση διαφορετικών χωρών με διαφορετικές παραδόσεις. Αυτό που μας συνδέει είναι κοινέ αξίες που δεν μπορούν βέβαια να παλύψουν τις διαφορές μας, ούτε τις διαφορές στην οτροπία μας, Ακριβώς επειδή έχουμε πολλές και διαφορετικές ε, λύσεις μπορούμε και προχωράμε. Ο συμβασμός είναι το βασικό, αλλιώς κάθε φορά η κάθε χώρα νιώθει ότι πλήττεται. Έχει μεγάλη παράδοση η Ουγγαρία και σίγουρα σκέφτεται διαφορετικά από ό,τι άλλες χώρες. Η Ουγγαρία αποφάσισαν για μια κυβέρνηση και η κυβέρνηση αυτή είναι απόλυτα νόμιμη και μπορεί κάλλιστα να επιλέγει το δικό της πρόγραμμα. Μπορούν να γίνουν ε, διαμαρτυρίες ειρηνικά για να εκφράσει ο κόσμος και αντιπολίτευση ε, την απόψή του και αυτό το επιτρέπει η κυβέρνηση και έτσι μπορούμε και εμείς και έχουμε διάλογο με την Ουγγρική κυβέρνηση. Οτιδήποτε άλλο είναι θέμα του Ουγγρικού λαού και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υπονομεύει τη δημοκρατία σε ένα κυρίαρχο κράτος. Ευχαριστούμε. Γιώργος Επιτίδιος τώρα, παρακαλώ. panie przewodniczący! η ευρωπαϊκή ένωση κατηγορεί την ουγγρική κυβέρνηση ότι παραβιάζει τις αρχές του κράτους δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ για άλλες χώρες ανέχεται να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. ο πραγματικός λόγος για τον οποίο συμπεριφέρεται έτσι η ευρωπαϊκή ένωση είναι το ότι η ουγγαρία αρνείται να χορηγήσει πολιτικό άσυλο σε μετανάστες οι οποίοι διώκονται για ποινικά αδικήματα και σε άλλους οι οποίοι ελέγχονται και καθοδηγούνται από διεφθαρμένες μκο. αντί λοιπόν να συνεργαστεί με την ε, κυβέρνηση της ουγγαρίας τόσο ώστε αυτή να χορηγήσει πολιτικό άσυλο στο ποσοστό και των μεταναστών που οφείλει να χορηγήσει επιλέγει την οδό της συγκρούσεως. όμως η κυβέρνηση της ουγγαρίας προστατεύει τα συμφέροντα του κρικού λαού. δεν είναι σαν την ελληνική κυβέρνηση η οποία είναι ενδοτική ε, δέχεται και υποκύπτει στις πιέσεις και έχει μετατρέψει την ελλάδα σε ένα απέραντο καταβλισμό δυστυχισμένων μεταναστών στους οποίους ούτε χορηγείται πολιτικό άσυλο ούτε τους δέχεται κάποια χώρα αλλά και ούτε απελάβνονται. τελειώνω θέλοντας να πω ότι η συμπεριφορά αυτή προς την ουγγαρία αποτελεί ε, το χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποκρισίας της ευρωπαϊκής ενώσεως διότι ενώ στην ουγγαρία συμπεριφέρεται έτσι η τουρκία αρνείται να ακολουθήσει την ίδια συμπεριφορά πρέπει να ολοκληρώσουμε πριν τα μεσάνυχτα την ε, Ολομέλεια σήμερα. Λέσλο Τόκας τώρα είναι επόμενος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Η απόψινή συζήτηση οφείλεται στους πράσινους και στους συνοδοιπόρους τους. Ήδη την τελευταία φορά που συζητήθηκε το θέμα εδώ, είχε καταδικαστεί η Ουγγρική κυβέρνηση. Πάλι καταδικάζεται η Ουγγαρία σήμερα, διότι οι αριστεροί και φιλελεύθεροι κάνουν στην ουσία ευρωπαϊκό προοικοϊκό αγώνα εδώ. Και υφιστάμεθα εμείς το στίγμα στην Ουγγαρία οι χειρότεροι όμως είναι οι Ούγγροι βουλευτέ τη αντιπολίτευσης, οι οποίοι όπως και επί εποχής κομμουνιστικού καθεστώτος απεργάζονται την κατάρρευση της ένομης τάξη στην Ουγγαρία. Σας παρακαλώ να μην του ακούτε. Ζήτω η Ουγγαρία, ζήτω η Ευρώπη. Ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμαντς, όταν γίνεται μια συζήτηση για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Ευρώπη, εκείνος λέει «Α, συζητάτε μονίμως για την Πολωνία και την Ουγγαρία». Εγώ συμφωνώ λοιπόν με την ιδέα σας και ας ε, μιλήσουμε για την ενεργοποίηση του άρθρου 7. Το κράτος δικαίου απειλείται αυτές τις μέρες από αυταρχικά καθεστώτα. Στην συνθήκη αναφέρεται ότι το άρθρο 7 μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά από μία ψηφοφορία η οποία θα περάσει με τα δύο τρίτα των ψήφων των ψηφισάντων. Αυτό, δεν, αυτό το νούμερο δεν το φτάσαμε ποτέ το 2 τρίτα των ψηφισάντων. Στα αυταρχικά καθεστώτα, για να ξεκινήσει μια αντίστοιχη διαδικασία, ε, γίνεται νοθεία στις εκλογές. Πρέπει να σας πω το εξής. Ο Όρμπαν έκανε μία διάγνωση για το τι συμβαίνει σε αυτή την αίθουσα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να αντιδράσω σε κάποια από αυτά που άκουσα. Καταρχάς, αυτοί που λένε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, είναι πολιτικό παιχνίδι εδώ, να σας παραπέμψω σε αυτά που είπα στην αρχική μου παρέμβαση. Ε, εμείς εξετάζουμε συγκεκριμένα πράγματα και θέτουμε ερωτήματα. Πιστεύουμε όταν πιστεύουμε ότι οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δεν συνάδουν με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εμείς προχωρούμε. Έχουμε τον νόμο Stop Soros, να σταματήσουμε το σώρο. Η επανεγκατάσταση ε, εκτός της Ουγγαρίας ε, για το, το πρόγραμμα του, Ευρωπαϊκού, του Κεντρικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Κάτι έχει αλλάξει λοιπόν δραστικά και έχουμε ερωτήματα η συγχώνευση πάνω από 400 ΜΜΕ, χωρίς να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να ελέγχουν αν αυτό συνάδει με την νομοθεσία. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα. Η υιοθέτηση δύο νέων νόμων ε, για τα νέα ε, διοικητικά δικαστήρια. Συγκεκριμένο πράγμα. Ο νέος νόμος για τις υπερορίες. Έχουν συζητηθεί πολλά πράγματα σχετικά. Ερωτήματα γύρονται για το αν ε, συνάδει αυτό με το ευρωπαϊκό δίκαιο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και τώρα, ας πάμε στο θέμα αρχής που μπαίνει εδώ. Η δημοκρατία πάντα χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να μην συμμορφωθεί κανείς με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι η δημοκρατία, δεν λειτουργεί έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουγγαρία, ευτυχώς, Ε, επέλεξε, ευτυχώς επέλεξε, με κυρίαρχη απόφαση να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ε, ενέκρινε το Κοινοβούλιο, επιβεβαιώθηκε από δημοψήφισμα του Ουγγρικού λαού. Αν αποφασίσει να γίνει μέλος μια οργάνωση που βασίζεται σε συνθήκε όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω τη επιλογή σου λε ότι θα ακολουθήσει του κανόνε τη συνθήκη. Και η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, έχει το καθήκον να εξετάσει εάν τα κράτη-μέλη ακολουθούν του κανόνε τη συνθήκη. Οι οποίοι κανόνε είναι ξεκάθαροι για πολλά θέματα και ειδικά για το θέμα του κράτου δικαίου. 2 και 19 της συνθήκης που λένε ξεκάθαρα για το διαχωρισμό των ε, εξουσιών, την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης κτλ. κτλ. Αυτά ψάχνουμε, αυτά κοιτάμε. Δεν θέλουμε να στυλιτεύσουμε χώρες που δεν θέλουν τους μετανάστες. Δεν θέλουμε να επιτεθούμε στην δημοκρατική λειτουργία ενός κράτους μέλους ή στην ε, πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε οι χώρες να λογοδοτούν για κάτι που επέλεξαν να κάνουν χωρίς να τις πιέσει κανένας. Ε, ελεύθερα έκαναν μια κυρίαρχη επιλογή. Επέλεξαν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η μορφιά τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κάθε κράτο κυρίαρχα αποφασίζει. Ακριβώ γι' αυτό η Ουγγαρία επωφελήθηκε πάρα πολύ από αυτή την ένταξη και όλα τα άλλα κράτη-μέλη έδειξαν τεράστια αλληλεγγύη με την Ουγγαρία για να κλείσει το χάσμα και να εφημερούν οι πολίτες οι Ούγγροι όπως το αξίζουν. Αλλά δεν έχετε μόνο δικαιώματα, έχετε και υποχρεώσει. Έχει υποχρεώσει η Ουγγαρία. Ε, υποχρεώσει αναφέρονται στη συνθήκη και είναι καθήκον των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, του Συμβουλίου, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Κοινοβουλίου να φέρνουν να ελέγχουν το πώς συμπεριφέρεται ο κανένας και να λογοδοτούν όλοι ενώπιόν τους. Αυτό κάνουμε εμείς ενώπιον της Ουγγαρίας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμανς και τώρα η κυρία Τσότεκ μέρος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας διαβεβαιώ για άλλη μια φορά ότι η Προεδρία και το Συμβούλιο συνολικά δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην τήρηση του κράτους δικαίου και στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι πράγματα τα οποία βρίσκονται στην καρδιά των όσων πιστεύουμε. Σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις απόψεις που εκφράσατε σήμερα κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Ακούσαμε τι ζητάτε και παραμένουμε ανοιχτοί υπέρ μιας πραγματιστικής προσέγγισης. Σας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Πρόεδρος, κυρία Χοτάλα στο Προεδρείο, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Συμβούλιο. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Και το επόμενο μας θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της ΥΠΑ εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση στην Βενεζουέλα. Δεν θα έχουμε μπλε κάρτες ή catch the κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής. Ενημερώθηκα ότι ο Επίτροπος Τελιανίδης θα αντικαταστήσει την κυρία Μογκερίνη στη συζήτηση αυτή. No niin, siirrymme sitten keskusteluun. Παρακαλώ. Τώρα θα περάσουμε στη συζήτηση, όπως έλεγα, για την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Ο Επίτροπος Τηλιανίδης θα πάρει το λόγο εκ μέρους της κυρίας Μογκερίνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι. Οι στιγμές που ζει η Βενεζουέλα είναι πολύ σημαντικές. Η κρίση επιδεινώνεται από ό,τι φαίνεται καθημερινά και κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα και πολύ παραπάνω φεύγουν από τη χώρα, την εγκαταλείπουν κάθε στιγμή προκειμένου να γλιτώσουν. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για να μπορέσει ο κόσμος της Βενεζουέλας ελεύθερα με δίκαιες εκλογές να αποφασίσει για το μέλλον του. Αυτή είναι η μόνη λύση για να βγούμε από την κρίση. Στις 23 Ιανουαρίου μαζικά ο κόσμος στην Βενεζουέλα ζήτησε δημοκρατία. Οι διαδηλώσεις αυτές αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη βία από τις αρχές, κάτι το οποίο οδήγησε σε πολλούς θανάτους και ακόμα πιο πολλούς τραυματισμούς και συλλήψεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φρόντισε να ακούγεται τη φωνή της με δύο δηλώσεις. Είπα το εκπρόσωπος, η συναδερφός μου έκανε τις δηλώσεις αυτές εκ μέρους και των 28 χωρών μελών και σε συνεργασία με τους εταίρους μας διεθνώς. Και ζητήσαμε να οργανωθούν ελεύθερες δίκες και αξιόπιστες εκλογές προκειμένου να επανέλθει η δημοκρατική και συνταγματική τάξη στη χώρα. Με ελεύθερε, δίκες και αξιόπιστες εκλογές πιστεύουμε ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα έπρεπε να μπορούν να συμμετέχουν χωρίς εμπόδια θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα εθνικό συμβούλιο με ισορροπημένη σύνθεση. Εννοούμε επίσης ότι διεθνείς παρατηρητές θα έπρεπε να παρακολουθήσουν ολόκληρη τη διαδικασία, κάθε πτυχή της εκλογικής διαδικασίας. Οι προεδρικές εκλογές του ΜΕΜ που μας πέρασε δεν ήταν ούτε ελεύθερες, ούτε δίκες, δεν είχαν ούτε και αξιοπιστία. Δεν είχαν λοιπόν καθόλου δημοκρατική νομιμότητα η χώρα χρειάζεται μια χώρα που να εκπροσωπεί πραγματικά τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας. Αν δεν ανακοινωθούν νέες προεδρικές εκλογές σύντομα, οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν και άλλη δράση και μπορεί μέχρι και να αναγνωρίσουν νέα ηγεσία για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει απόλυτα την Εθνική Βουλή και προς το παρόν είναι το μόνο ε, νομιμοποιημένο όργανο και το μόνο που έχει εκλεγεί ελεύθερα από τους κατοίκους της Βενεζουέλας. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουν οι εξουσίες στο σώμα αυτό. Και πρέπει επίσης να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κάθε μέλους, πρώτα απ' όλα του Προέδρου της, του Χουάν Αγκοίντο, και πρέπει να υπάρξει εγγύηση για τις πολιτικές του ελευθερίες. Τώρα, θα πρέπει να αποφύγουμε στρατιωτική κλιμάκωση και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια ειρηνική και δημοκρατική λύση στην κρίση αυτή. Με αυτό το στόχο λοιπόν, είπα εκπρόσωπο, εκπρόσωπος, είναι συνεχώς σε επαφή με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσε, αλλά και με άλλους μας εταίρους διεθνώς και στη Λατινική Αμερική. Χτες, είπα εκπρόσωπος, συναντήθηκε με τους Υπουργούς Εξωτερικών ε, του Ισημερινού και της ε, Βολιβίας και με τον Αντώνιο Κοτιέρης και με τον ε, Γενικό Γραμματέα ο πλευράς του Βατικανού με τον Αργεντινό Πρόεδρο Μάρση με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Πομπέο και με τους Υπουργού Εξωτερικών του Καναδά, της Χιλής, της Κωνσταντίνα, της Κούβας, του Μεξικού, και της Με όλους αυτούς συζήτησε την πρότασή μας να δημιουργήσουμε μια διεθνή ομάδα επαφής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό οι περιφερειακοί παράγοντες να συνεργαστούν για να επιτραπεί αυτή η δημοκρατική διαδικασία. Πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι η στρατιωτική παρέμβαση μόνο χειρότερα θα έκανε τα πράγματα. Η λύση σε αυτή την κρίση πρέπει να έρθει από τον ίδιο τον κόσμο της Βενεζουέλας. Βέβαια, οι προποθέσει οι συνθήκε δεν είναι καλές σήμερα για να υπάρξει διάλογος μεταξύ των διαφόρων πλευρών στη χώρα. Συνεπώς, η ομάδα αυτή επαφής δεν θα έχει απευθεία διάλογο με τι δύο πλευρέ στη Βενεζουέλα, αλλά μια διεθνή πρωτοβουλία θα μπορούσε να βοηθήσει να δημιουργηθούν οι προποθέσει οι οποίε θα οδηγήσουν τελικά σε μια πολιτική διαδικασία μέσα στη Βενεζουέλα και σε ελεύθερε και δίκαιε εκλογέ με όλε τι απαραίτητε εγγυήσει. Θέλουμε να αρχίσουν και πάλι συνομιλίες σε διεθνές επίπεδο που θα είναι ένα διάμεσο βήμα για να αρχίσουν οι συνομιλίες στη Βενεζουέλα. Οι προετοιμασίε για την ομάδα αυτή επαφή έχουν ήδη ξεκινήσει και είπα το εκπρόσωπο θα τα συζητήσει όλα αυτά αύριο με τους 28 Υπουργούς Εξωτερικών. Συγχρόνως η Ευρωπαϊκή Ένωση εμένει στη θέση της που αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου που μας πέρασε. για περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το καθεστώς του Μαντούρο. Και θέλω να τελειώσω με δύο λόγια για το ανθρωπιστικό μας έργο, γιατί η κατάσταση στην Βενεζουέλα, η ανθρωπιστική, δυστυχώς επιδεινώνεται. Από στιγμή σε κάθε στιγμή επιδεινώνεται. Εμείς έχουμε αναλάβει την υποχρέωση και συνεχίζουμε να θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο στην Βενεζουέλα αλλά και όλους αυτούς που έφυγαν από τη Βενεζουέλα και να στηρίξουμε τις χώρες που τους υποδέχτηκαν. Θα θυμόσαστε ότι στο Στρασβούργο είχα υποσχεθεί 20 εκατομμύρια παραπάνω σε ανθρωπιστική βοήθεια. Οπότε η συνολική στήριξη μόνο για πέρυσι έφτασε στα 55 εκατομμύρια για τους ε, ανθρώπους από τη Βενεζουέλα, είτε μέσα στη Βενεζουέλα είτε εκτός. Οι εταίροι μας στην ανθρωπιστική βοήθεια ε, πολλές φορές προσφέρουν και βοήθεια παρασκηνιακά με πολύ αποτελεσματικούς τρόπους και απτούς. Η Φρεντερίκα Μαγκερίνη συναντήθηκε με τον Εντουάρτο Στέν που είναι ο ειδικό αποστελμένος του ΟΗΕ και εμείς εκφράσαμε την επιθυμία μας να συνεργαστούμε μαζί του για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι προκλήσεις και στηρίζουμε μία απάντηση από την περιφέρεια, από την περιοχή για αυτό το πρόβλημα της Βενεζουέλας. Υπάρχουν και Ευρωπαίοι πολίτες εκεί, υπάρχουν και ε, Ευρωπαίοι που έχουν οικογένειες εκεί πέρα και εννοείται ότι θέλουμε να αποφύγουμε πάση θυσία ένα πόλεμο στην περιοχή Βενεζουέλα πρέπει να βοηθηθεί να βρει διέξοδο από αυτή την τραγική κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επίτροπε Στυλιανίδη. Από το ΕΛΚ, ο κύριος Κονσάλες Πόνς. Στις 3 ε, ε, Ιανουαρίου, ο πρόεδρος της Βουλής, ε, Χουάν Γουαϊδό, ανέλαβε προσωρινά την προεδρία της χώρας. Η εντολή του έχει ένα και μόνο σκοπό, να οδηγήσει την Βενεζουέλα σε ελεύθερες εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Πολλά κράτη από τότε, μεταξύ των οποίων και μεγάλα ε, λατινοαμερικανικά κράτη, Αυστραλία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Καναδάς, αναγνώρισαν την ε, ενδιάμεση προεδρία του Γκαϊδό. Το θέμα είναι γιατί περιμένει η Ευρώπη. Όλοι μας κοιτάνε. Η Βενεζουέλα μας κοιτάει. Εμείς τι κάνουμε. Μέχρι πότε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα περιμένουμε. Αυτό που βλέπετε στους δρόμους της Βενεζουέλας, ε, αυτοί που κατεβαίνουν στους δρόμους δεν είναι Ευρωπαίοι, αλλά πολεμούν για τις ίδιες αξίες με εμά. Δεν είναι Ευρωπαίοι, αλήθεια είναι, αλλά πολεμούν για μια αξιοπρεπή ζωή όπως και εμείς. Δεν είναι Ευρωπαίοι, αλήθεια είναι, αλλά πολεμούν για την ειρήνη και την ελευθερία όπως πολεμούμε και εμείς. Δεν είναι Ευρωπαίοι, αλλά πολεμούν για τα παιδιά τους να μην παραμείνουν στις φυλακές του Μαδούρου, αλλά, του Μαδούρου, αλλά στις, ε, στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Πολεμούν ούτω ώστε πάνω από 2,5 εκατομμύρια Βενεζουελιάνοι που είναι πρόσφυγες και εξόριστοι να επιστρέψουν στη χώρα ψηλά το κεφάλι, όπως και εμείς μετά τον πόλεμο. Δεν είναι Ευρωπαίοι, αλλά πολεμούν ούτω ώστε ο θάνατος τόσων πολλών αθώων ανθρώπων πάνω σε, κατά τη διάρκεια 19 ετών και πλέον τυραννίας να μην πάει σμάτιν. Δεν είναι Ευρωπαίοι, αλλά είναι Ευρωπαίοι, γιατί και εμείς είμαστε Βενεζουλελιάνοι όταν πρόκειται για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια. Όταν πρόκειται για αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν έχουμε δικαίωμα να λεγόμαστε Ευρωπαίοι αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα και δεν λειτουργήσουμε σαν να ήμασταν οι Βενεζουελιάνοι. Πρέπει να υπερασπιστούμε την ε, δημοκρατία, την ελευθερία. Δεν μπορούμε να είμαστε ουδέτεροι και να πάρουμε ίσες αποστάσεις. Η Ευρώπη είναι μια φιλοδοξία, ένα όνειρο, ένα ιδεώδες. Όταν γίνονται τόσοι βίαιοι θάνατοι, όταν πεθαίνουν άνθρωποι γιατί δεν υπάρχουν φάρμακα, όταν πεθαίνουν έγκυες γυναίκες γιατί δεν έχουν να φάνε, όταν πεθαίνουν παιδιά γιατί δεν έχουν να φάνε, τι άλλο πρέπει να συμβεί στη Βενεζουέλα, ούτω ώστε να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει εκεί. Γι' αυτό ζητούμε και από το Κοινοβούλιο και από όλου εδώ τρία πράγματα. Να αναγνωρίσουμε την Εθνική Συνέλευση και τον ενδιάμεσο πρόεδρο, ως, τον Χουάνο Γουαϊδό, ως ε, το μόνο νόμιμο πρόεδρο ε, στη Βενεζουέλα. Επίσης, να ζητήσουμε από το, στρατό ε, ειρηνική μετάβαση με σεβασμό του συντάγματος. Επίσης, για τι νέε αρχέ να δώσουμε ένα πακέτο βοήθειας για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση που ζει η Βενεζουέλα. Ο Μαδούρο είναι τύρανο. Αν ναι, δεν μπορούμε να του δώσουμε περιθώριο για να καλέσει εκλογές. Αν είναι τύρανο, δεν μπορούμε να του ζητήσουμε διάλογο. Εάν είναι τύρανο, δεν μπορούμε να περιμένουμε να διορθωθεί και να διορθώσει τα πράγματα. Αν περιμένουμε τον τύρανο, του δίνουμε ευκαιρίε. Οι τύρανοι δεν συγκαλούν ε, εκλογέ, δεν συνομιλούν, δεν διορθώνουν τα πράγματα. Είναι τύρανοι, δεν είναι λουλουδάκια του αγρού, είναι επικίνδυνοι. Και με τους τύρανου πρέπει να υψώσεις το κεφάλι και με αρχές στο πλάι σου, με σοβαρότητα, ούτω ώστε να αλλάξουν. Ας αναγνωρίσουμε την νόμιμη εξουσία στην Βενεζουέλα. Εμείς είμαστε το Κοινοβούλιο και ας είμαστε το πρώτο θεσμικό όργανο που αναγνωρίζουμε την νέα εξουσία στη Βενεζουέλα. Και ας βοηθήσουμε την Βενεζουέλα να αλλάξει. Οι τύρανοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν σε καμία περίπτωση τη δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ κύριε Γκονθάλεθ Πόνς. Τώρα, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Ατόντο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε ότι η Βενεζουέλα εδώ και πολλά χρόνια υποφέρει από μια πολιτική δημοκρατική κρίση πάρα πολύ σοβαρή και οικονομική και κοινωνική όμως τεράστια συνεπώς υποφέρει από ανθρωπιστική κρίση. Αυτό τα λέει όλα. Η διεθνής κοινότητα δεν αναγνώρισε τις εκλογές του Μαΐου που μας πέρασε, οπότε δεν αναγνώρισε ούτε και τον κύριο Μαντούρο ως πρόεδρο από τις 10 Ιανουαρίου που ορκίστηκε. Ο κύριος Γκουάιντο αυτό προκηρύχθηκε πρόεδρος της χώρας και αυτό έφερε τη χώρα σε μεγάλη αστάθεια. Οπότε, κύριε Κονσάλες ε, Πόντς, η Ευρώπη έχει βάλει ένα σωστό κριτήριο και το κριτήριο είναι ότι προτιμάει συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, την κυβέρνηση που διαθέτει τον μηχανισμό, τον εκλογικό κτλ. Και έτσι κι έχει 30 μέρες στη διάθεσή του για να συγκαλέσει εκλογές και μπορεί να φροντίσει να υπάρχουν εγγύσεις. Υπάρχει μια προθεσμία και είπαμε στον κύριο Μαντουρό, αν δεν προκηρύξετε εκλογές, τότε εμεί θα αναγνωρίσουμε τον κύριο Κουαϊντό. Λοιπόν, αύριο, βάσει τη συμφωνία που πετύχαμε οι πολιτικέ ομάδε, αυτό ακριβώ θα κάνουμε. Και αυτό θα κάνουν και χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση τι επόμενε ημέρε. Και αυτό είναι η συνέπεια του ότι δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει μια λογική εξέλιξη στην κατάσταση αυτή. Η συμφωνία λοιπόν, την οποία αύριο θα ψηφίσουμε όλες οι πολιτικές ομάδες κυρίες και κύριοι, συμπεριλαμβάνει και την απόρριψη οποιασδήποτε παρέμβασης που μπορεί να υπάρξει με βία ή μέσω του στρατού. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε γιατί πρέπει να καταδικάζουμε και να απορρίπτουμε οποιαδήποτε πρόταση, οποιαδήποτε πρωτοβουλία που να περιλαμβάνει τη βία. Αναφέρθηκε στρατιωτική κλιμάκωση ο Επίτροπο. Όντω δεν είναι έτσι που θα λυθεί η κρίση στη Βενεζουέλα. Ε, από την άλλη, η ομάδα μα λέει ότι πρέπει να υπάρξει στήριξη στην ομάδα επαφής που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί κυρίες και κύριοι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να παίξει ένα ρόλο, όχι σαν και αυτό που παίζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Το δι... κάνει ό,τι θέλει ο καθένα. Αλλά ο δικό μα ο ρόλο είναι ρόλο κάποιου που διευκολύνει, διαμεσολαβητή, που ελέγχει, που φροντίζει να εξασφαλίσει, να εγγυηθεί τη δημοκρατική διαδικασία. Και μόνο έτσι μπορούμε να τα καταφέρουμε να βγούμε από την κρίση στη Βενεζουέλα. Οποιοδήποτε από τα άλλα σενάρια που ακούγονται, να γίνουν εκλογές από τον Μαντούρο, να γίνουν εκλογές από τον Γουαϊντό ή από κανέναν, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δικιά της ομάδα επαφή και με τις χώρες τη περιοχή πρέπει να συνεχίσουν να προσπαθούν να βρουν μια ειρηνική και δημοκρατική διέξοδο για τη Βενεζουέλα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται, εντάξει, να πούμε ότι είναι, α πούμε ότι αναγνωρίζουμε τον Γκουάιντο, ότι λέμε ότι ναι, αυτό είναι πρόεδρο και η αντιπολίτευση. Πολύ ωραία. Αλλά πρέπει πολιτικά να είμαστε διατεθειμένοι να δράσουμε επίσης. Εμείς εδώ και χρόνια, οι σοσιαλιστές κυρίως, λέμε ότι ο σοσιαλισμός είναι ελευθερία και ότι δεν μπορεί να υπάρχει αριστερά κατά της δημοκρατίας. Και αυτό το επαναλαμβάνω ξανά εδώ και το λέω και μπορώ να το πω και τότε κατάματα τον κύριο Μαντούρο. Οπότε ναι, έχουμε μια συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων ακριβώς για να επανέλθει η ισορροπία και για να μπορούμε να δράσουμε πολιτικά από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσουμε μια διέξοδο ειρηνική και δημοκρατική στη Βενεζουέλα μέσω τη πολιτική δράση που μπορούμε εμείς οι Ευρωπαίοι να ασκήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Πρώτα πρώτα καλησπέρα σε όλες και όλους. Έχουμε και την μεγάλη χαρά να έχουμε στα θεωρία επισκέπτες που είμαι βέβαιος ότι εκτιμούν τις ομιλίες. Όμως υπενθυμίζω στους επισκέπτες ότι δεν επιτρέπεται να χειροκροτούν ούτε να κάνουν ιονδήποτε θόρυβο, όσο και αν επιθυμείτε να ενθαρρύνετε τους ε, αγορητές. Παρακαλώ λοιπόν να σεβαστείτε τους κανόνες που ισχύουν στις ορομέλειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Τάνοκ, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, με τον πληθωρισμό τη Βενεζουέλα να φτάνει στα 10 εκατομμύρια της εκατό, με 3 εκατομμύρια Βενεζουελάνου να έχουν φύγει από τη χώρα. Δυνάμεις ασφαλεία υπό τι εντολέ του Μαδούρο χρησιμοποιούν όλο και πιο α, βάρβαρες τακτικές. Δεν είναι λοιπόν να απορεί κανεί με τις πρόσφατες εξελίξεις. Εγώ συμφωνώ με τον Γοηδό που να κηρύχθηκε πρόεδρος χρειάζεται να αναγνωριστεί από τις δημοκρατικές κυβερνήσεις όλου του κόσμου και έχει έρθει και η σειρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει πολυφωνία, δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Αυτά τα κατέδειξε και είπατε εκπρόσωπος ήδη από εδώ και 1,5 χρόνο. Ο ίδιος, η ίδια μάλλον, η Γενική Γραμματέας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών κατηγορεί ανοιχτά τον Μαδούρο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σημειώνοντας ότι ναι μεν η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι διπλωματική δράση, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλειστεί κανένα άλλου είδου δράση. Ωστόσο, οι διπλωματικέ δράσει ω τώρα απέτυχαν. Η απομάκρυνση του Μαδούρο είναι και η πρώτη, το πρώτο βήμα που θα πρέπει να γίνει. Χαίρο για την απόφαση της ε, Τράπεζας της Αγγλίας που δεν επιτρέπει στην Βενεζουέλα να έχει πρόσβαση σε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποθεματικά που διαθέτει στην τράπεζα αυτή. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθήσει και να κάνει το ίδιο όπως οι Αμερικανοί, δηλαδή να επιβάλλει κυρώσεις στις ε, εταιρείες που συνεργάζονται με το καθεστώς Μαδούρο. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ ολοκληρώστε για να αποφευθεί η αδίποτε βία κατά πολιτών. Ζητώ συγγνώμη αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά θα πρέπει να τηρήσουμε απολύτω τα χρονικά όρια. Διότι πληροφορούμε ότι έχουμε ήδη υπερβεί ε, τον χρόνο μας και έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Ναρτ, δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Βενεζουέλα οικονομικά, κοινωνικά, θεσμικά είναι μια καταστροφή με εκατομμύρια θύματα είτε που βρίσκονται στην εξορία. Αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι που είπε ο Λένιν, που είπε ότι η εξορία είναι ένα δημοψήφισμα στο οποίο ψηφίζει κανείς με τα πόδια. Ε, ναι, τρία εκατομμύρια ψήφισαν και φύγανε. Συνεχίζω λοιπόν. Ο Ματούρο είναι μια εξουσία που βασίζεται σε ψεύτικες εκλογές, στη βία, στην καταστολή, που στηρίζεται από τους κουβανούς. Βρίσκεται στον αντίποδα της ελευθερίας, της επανάστασης και μια ιδέα που για μένα παραμένει ευγενή και ονομάζεται σοσιαλισμός. Ο νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλα, ο συνταγματικός, είναι ο Χουάν Καϊντό, βάσει του άρθρου 233 του συντάγματος. Γιατί έπαψε να είναι ο πρόεδρος Μαδούρου όταν προκήρυξε εκλογές πριν λήξει η θητεία του, οι οποίες όμως δεν ήταν σωστές, ήταν επιξενοθεία. Έτσι λοιπόν, τώρα είναι δυνατόν αυτός ο πρόεδρος να προκηρύξει εκλογές. Αυτό είναι σουρεαλιστικό, θυμίζει Σαλβαντόρο Γαλή. Είναι δυνατόν, Νταλή. Όλη αυτή η περίοδος οδήγησε σε λίγες μέρες σε παραπάνω χίλιους κρατούμενους. Πώς λοιπόν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να προκηρύξει εκλογές απέτυχαν όλες οι διαμεσολαβήσεις. Οπότε πρέπει να είναι αποφασιστικό το Κοινοβούλιο. Αύριο θα ψηφίσουμε και θα ψηφίσουμε την αναγνώριση του νόμιμου Προέδρου της Βενεζουέλα που είναι ο Χουάν Κουαϊτό. Θα ψηφίσουμε τη διατήρηση της αναγνώρισης του μόνης νόμιμης βουλής της Βενεζουέλας που είναι η μόνη που έχει εκλεγεί δημοκρατικά. Θα Ζητήσουμε επίσης να καταδικαστεί το καθεστώς του Μαντούρο και θα απαιτήσουμε πλήρη διερεύνηση των εγκλημάτων του τυράννου. Οπότε, συμπερασματικά, υπάρχει κάτι που λέγεται ε, αξιοπρέπεια, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, ελευθερία. Οπότε πραγματικά από το βάθος της ψυχής μου για τον κόσμο της Βενεζουέλας λέω ζήτω η ελεύθερη Βενεζουέλα. Πρόεδρος. Παρακαλώ πολύ ε, τους επισκέπτες ε, στα θεωρία. Αντιλαμβάνομαι ότι ε, παρακολουθεί το θέμα με κάποια συναισθηματική φόρτιση, ωστόσο οι κανόνες, οι κανόνες του Κοινοβουλίου δεν επιτρέπουν χειροκροτήματα ή άλλες ενθαρρύνσεις των αγοριτών. Ορίστε, η κυρία αγορητών. οριστε η κάτω καταδικάζουμε τις δράσεις ε, του καθεστώτος της Βενεζουέλας που έχει οδηγήσει στα όρια την Βενεζουέλα και έχει οδηγήσει στην έξοδο 3 εκατομμύρια Βενεζουελινού πολίτε. Ωστόσο, στην απάντηση που θα δώσουμε δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τι βασικέ αξίε τη διπλωματία για να διατηρήσουν πρώτα-πρώτα οι άνθρωποι το δικαίωμα να επιλέγουν τι ηγεσίε του. Η Λατινική Αμερική, Αμερική έχει μακρά και τραγική ιστορία παρεμβάσεων από ξένου παράγοντε, οι οποίοι συχνά κινούνται από την ε, επιθυμία αρπαγής του φυσικού τη πλούτου. Για την ασφάλεια των πολιτών τη, δεν επιτρέπεται αυτοί να μπουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Η κρίση στην Βενεζουέλα πρέπει να λυθεί ειρηνικά και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω πολιτικού διαλόγου. Υποστηρίζουμε τι προσπάθειε τη υπάτη εκπροσώπου Μογκερίνη σε συνεργασία με Λατινοαμερικανούς ηγέτες για να δημιουργήσει ομάδα επαφών που να ανοίξει τον δρόμο για ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Για ένα λεπτό ο κύριος Πιμέντα Λόπες. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να νομιμοποιήσει το πραξικόπημα που συνέβη στην Βενεζουέλα που ανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ να βάλει στην εξουσία μια μαριονέτα του. Αυτά είναι απαράδεκτα. Και τώρα ζητούν προεδρικές εκλογές στην Βενεζουέλα και αυτό πρόκειται για συστηματική υπονόμευση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών αρχών στην χώρα αυτή. Πρόκειται για θέματα οικονομικών συμφερόντων και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τροφοδοτεί αυτά. Πρόκειται για μεγάλο κίνδυνο για την χώρα αυτή και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στρατιωτικής παρέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών που υποσκάπτει την ειρήνη. Πρόκειται για τον βενεζουελάνικο λαό και δεν μπορούν να παίζουν με τον λαό αυτό. Κάτω τα χέρια από την Βενεζουέλα. Για δύο λεπτά εξ ονόματος του ομάδας EFDD. Ορίστε. Έχω συναντηθεί με Βενεζουελανούς πρόσφυγες από το καθεστώς Μαδούρο. Μια χώρα που θα έπρεπε να είναι εύπορη, όπου όμως ο πληθωρισμός τι είναι, 100.000 ή 100, 10 ε, εκατομμύρια τη εκατό πώς να το μετρήσει κανείς αυτό; Οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα, διότι δεν υπάρχουν τρόφιμα και το, αυτό το έχει προκαλέσει το καθιστό Μαδούρο. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει από τη Βενεζουέλα, άλλοι χιλιάδε βρίσκονται σε φυλακέ και εκατοντάδε έχουν τραυματιστεί βαριά σε διαμαρτυρίε. Όταν ο ίδιος αρχηγός της αντιπολίτευσης δεν του επιτρέπεται να βγει από τη χώρα και του παγώνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Πώς θα λυθεί αυτή η ανθρωπιστική κρίση στην Λατινική Αμερική. Όλε οι κυβερνήσει μα πρέπει να συνεργαστούν. Είτε είναι τη αριστερά, τη δεξιά ή του κέντρου. Δεν με ενδιαφέρει. Είτε πιστεύει κανεί στη δημοκρατία, είτε δεν πιστεύει στη δημοκρατία. Και όταν ο Μαντούρο λέει σήμερα ότι θα κάνει προεδρικές εκλογές το 2025 όσοι συμπαρατάσσονται μαζί του συμπαρατάσσονται με την βία και τη δικτατορία. Και πρόκειται για έσχος, πρόκειται για ντροπή για το Ηνωμένο Βασίλειο όταν βλέπω τον ε, σκιώδη υπουργό εξωτερικών της, ε, της, ε, του, μεγάλου, του Ηνωμένου Βασιλείου να μην κάνει τίποτα και ο ίδιος ο Τζέρεμι Κόρμπιν δεν κάνει τίποτα και εξακολουθεί να υποστηρίζει το καθεστώς αυτό. Η διεθνή κοινότητα θα πρέπει πράγματι ενωμένη να απαντήσει. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε στα Ισπανικά. Ο Μαδούρο δεν είναι νόμιμος πρόεδρος. Είναι τύρανος. Πρέπει να αλλάξει το καθεστώς της Βενεζουέλας. Άγγλοι, Ισπανοί, Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι, Όλοι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αλήθεια. Η λύση είναι η δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Σοφχάουσερ, για ένα λεπτό. Oui. Ευχαριστώ. Δεν μ' αρέσει ο κύριος Μαντούρο το καθεστώ του, αλλά ή που θα είσαστε για το κράτος δικαίου και θα το κάνετε πράξη ή αλλιώς θα είσαστε πραξικοπηματίες ή που θέσαστε το ένα είτε το άλλο. Τώρα, ο πρόεδρος που έχει αυτοκηρυχθεί πρόεδρος δεν είναι νόμιμος. Υπάρχουν πέντε περιπτώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Ο θάνατος, η παρέτηση, η σωματική ανεκανότητα, η καθαίρεση, η εγκατάλειψη του αξιώματος και καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν καλύπτεται. Οπότε δεν είναι δυνατόν να καθαιρεθεί με έτσι από την Εθνική Βουλή ο πρόεδρο μόνο με δημοψήφισμα. Το ανώτατο δικαστήριο αποτελεί και την εγγύηση του συντάγματο και εκεί ακριβώ ορκίστηκε ο κύριο ο πρόεδρο Μαδούρο στι 10 ε, Ιανουαρίου. Άρα αυτό είναι ο νόμιμο πρόεδρο και σε περίπτωση τη κέρνωση θέση αυτό που αναλαμβάνει δεν είναι ο πρόεδρο τη Εθνική Συνέλευση, αλλά είναι ο αντιπρόεδρο, δηλαδή η κυρία Ροντρίγκε. Ο Χουάν Γκριντο δεν ήταν υποψήφιος ε, στις προεδρικέ εκλογές ε, του Μαΐου του 18. Είναι πολιτικά άγνωστος, οπότε στο όνομα ποιας υποτιθέμενης λαϊκή στήριξη. Ποιου κράτου δικαίου λοιπόν θα μπορούσε να είναι ο νόμιμος πρόεδρος της χώρας. Πρόεδρο διακόπτη. Εξαντλήθηκε ο χρόνο σα. Ένα λεπτό. Ο κύριο Παπαδάκη, μία γεγραμμένο. καταγγέλουμε την ομοίη επέμβαση των ηνωμένων πολιτειών της ευρωπαϊκής ένωσης του νατο κυβερνήσεων της λατινικής αμερικής στα εσωτερικά της βενεζουέλας και την απόπειρά τους να επιβάλλουν με πραξικόπημα έναν πρόεδρο μαριονέτα και εκεί απειλούν με στρατιωτική επέμβαση για την προώθηση των επικίνδυνων σχεδίων τους όπως κάνουν παντού διεθνώς. καταγγέλουμε τη στάση κυβερνήσεων σαν της γερμανίας της ισπανίας της πορτογαλίας Όσο για την ελληνική, δεν βγάζει άχνα για την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα και ισχυρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δήθεν αδυνατή να έχει δική της εξωτερική πολιτική. Ενώ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν αναγνωρίζει τον πρόεδρο Μαδούρο και προκλητικά απειλεί με τελεσίγραφα. Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας έχει την ευθύνη για την υπεράσπιση των συμφερόντων του και την εκλογή της ηγεσία της χώρας του. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με το βενεζουελάνικο λαό που βιώνει την καπιταλιστική κρίση και εκμετάλλευση εκμετάλλευση. Στηρίζουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλα στη μάχη του για τα δικαιώματα της εργατικής τάξης για να ζήσει ο λαός χωρίς εκμετάλλευση και υπερελιστή. Ευχαριστώ συναδελφοί. Τέτοιες στιγμές λυπάμαι που είμαι πρόεδρος και ως πρόεδρος δεν, δεν μπορώ να παρέμβω επί της αρχής. Αλλά δυστυχώς ως πρόεδρος δεν μπορώ να παρέμβω επί της ουσίας. Αλλά θα δώσω το λόγο παρόλα αυτά στον Επίτροπο για να κάνει τις καταληκτικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ για τις ε, χρήσιμες και τολμηρές παρεμβάσεις σας. Όπως είπα και στην πρώτη μου παρέμβαση, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξακολουθήσει να είναι πολυσχηδής και θα έχει δύο στοιχεία. Και πίεση, αλλά και πολιτικά κανάλια μέσω των οποίων μπορούμε να φτάσουμε σε ειρηνική και δημοκρατική λύση. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνοδεύσουμε τη χώρα προς μια ειρηνική και διαπραγματευμένη λύση. Είναι δύσκολο το μονοπάτι, αλλά είναι το μόνο που μπορεί να προωθήσει μια δημοκρατική και βιώσιμη λύση στα προβλήματα και δεινά της χώρας. Φυσικά, οι Βενεζουελιάνοι και εντός και εκτός της χώρας, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν εκατομμύρια εκτός της χώρας πρόσφυγες, θα είναι το βασικό μας μέλημα. Ε, θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις α, ανάγκες τους. Ε, η δημοκρατία είναι και αυτό, πάνω απ' όλα. Θέλω, κλείνοντας, να σας εκφράσω την εκτίμησή μου για την υποστήριξή σας, για το ρόλο που παίζετε για να μείνει αυτό το σημαντικό θέμα στη διεθνή ατζέντα και όπως πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται στις δικές σας προσπάθειες, στη δική σας στήριξη, ούτω ώστε να έρθει η δημοκρατία στη Βενεζουέλα. Ευχαριστώ Επίτροπε. Χαίρομαι να προεδρεύω σε μια τέτοια συζήτηση, γιατί υπάρχει πλατιά συνένεση και είναι πραγματικά ευχάριστο συνέστημα να βλέπει κανείς αυτή τη συνένεση. Ε, ένας πρόεδρος δεν βλέπει πάντα κάτι τέτοιο στις συζητήσεις που γίνονται. Ο Επίτροπος μίλησε για αυτή την ε, συμμαχία, έκλεισε συζήτηση και τώρα θα ακούσουμε τις δηλώσεις ε, της Αντιπροέδρου και είπαν σε εκπροσώπου της Κομισιόν για την εξωτερική πολιτική, για τις τελευταίες εξελίξεις, στις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν. Ο Επίτροπος έχει το λόγο πάλι. Thank you Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι αρχή του έτους και από την αρχή του έτους οι εντάσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν έχουν οξυνθεί. Αφότου και τα δύο καθεστώτα επαναδιατύπωσαν τη θέση τους ε, ο ένας για τον άλλον. Εμείς είπαμε ακριβώς που βρισκόμαστε. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε το διάλογο ανάμεσα στην Κίνα και την Ταϊβάν και λυπόμαστε που οι σχέσεις ε, μεταξύ των στενών είναι παγωμένες τα τελευταία δύο έτη. Εμείς έχουμε την πολιτική μία Κίνα, για μία Κίνα. Δηλαδή αναγνωρίζουμε την ε, κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ως μοναδική νόμη κυβέρνηση της Κίνας, αλλά παράλληλα ε, θέλουμε να υπάρξουν στενότερες σχέσεις με την Ταϊβάν. Η, η συνεργασία και ο διάλογος με την ε, Ταϊβάν γίνεται όλο και πιο έντονος σε ανεπίσημο ε, επίπεδο. το σύστημα Ταϊβάν βασίζεται στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ταϊβάν μοιάζουν πάρα πολύ από πολλές απόψεις. Γι' αυτό πάντα ενθαρρύναμε την Ταϊβάν να είναι δραστήριο μέλος στην διεθνή κοινότητα. Και εμείς είμαστε σε επαφή με την Ταϊβάν. Ακόμα και όταν υπάρχει έλλειψη διπλωματικής αναγνώρισης. Ε, εμείς θέλουμε ειρήνη στην Ασία και δημοκρατία. Είμαστε μακριά γεωγραφικά, αλλά οι εντάσει στην Άπο Ανατολή μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη δική μας ασφάλεια, καθώ και το εμπόριό μας και τις οικονομίες μας. Ακριβώς για αυτού τους λόγους παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ όλες τις ε, εξελίξεις στα στενά της Ταϊβάν τα πρόσφατα χρόνια και οι δύο πλευρέ ε, σκλήριναν τη στάση του. Ε, γύρω από το θέμα μίας ε, προσέγγισης. Το Πεκίνο έκλεισε τα υψηλά κανάλια ε, επικοινωνίας από το 2016 και από τότε έχει αυξήσει μεγαλύτερη διπλωματική πίεση στην Ταϊβάν για να περιορίσει την Ταϊβάν και να αναγνωρίσει, να αναγκάσει μάλλον τους συμμάχους της Ταϊπέη να την εγκαταλείψουν. Οι ηγέτες της Ταϊπέη αρνήθηκαν την φόρμουλα «μία χώρα, δύο συστήματα». Οι οικονομικές και οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές ανθούν παράλληλα και η Κίνα είναι ο βασικός προορισμός των επενδύσεων του, εμπορικού, του Υπουργείου Εμπορίου της Ταϊβάν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς οι Ευρωπαίοι ζητάμε και από τις δύο πλευρές να αποφύγουν δράσεις και λόγια τα οποία μπορεί να κλιμακώσουν την ένταση ανάμεσα στα στενά της Ταϊβάν. Ενθαρρύνουμε και την Κίνα και την Ταϊβάν να συζητήσουν συνομιλ... Ε, επικοδομητικά μεταξύ τους και να αρχίσουν εκ νέου το διάλογο. Είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε όλες τις πρωτοβουλίες, να προστηρίξουμε το διάλογο, την συνεργασία, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είμαι ικανοποιημένος που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάει αυτό το θέμα θα πρέπει με κάθε ευκαιρία να προωθούμε μια πιο δυναμική και θετική σχέση ανάμεσα στην Κίνα και στην Ταϊβάν. Παράλληλα, να συνεργαζόμαστε πιο στενά με την Ταϊβάν όταν συγκλίνουν τα συμφέροντα και οι αξίες μας. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, Επίτροπε. Εκ μέρους του ΕΛΚ. Η κυρία για 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι σχέσει μεταξύ Ταϊβάν και Κίνα ποτέ δεν ήταν εύκολε. Και η ειρήνη ήταν εγγυημένη μόνο χάρη στις μεγάλες διπλωματικέ προσπάθειες τη Ταϊβάν για να διατηρήσει την αυτοδιάθεση και τον τρόπο ζωής της. Στι 2 Ιανουαρίου ο, πρόεδρο Κινέζος πρόεδρος Xi δήλωσε ότι η Κίνα επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει την βία για να ελέγξει την Ταϊβάν ακόμη και εάν είπε ότι θα επιδιώξει πρώτα την ειρηνική επανένωση με την Νήσο, με την Ταϊβάν δηλαδή, πάντως αυτή η τάση είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Η δήλωση ότι η Ταϊβάν αποτελεί μέρος της Κίνας και ότι οι λαοί και των δύο πλευρών θα πρέπει να επιδιώξουν την επανένωση υπό την ισχύ της συνένεσης του 1992 είναι σαφώς ξεπερασμένη. Όσο γνωρίζουμε, η πρόεδρος της Ταϊβάν Τσάι αμέσως απέριψε την αρχή μία χώρα με δύο συστήματα ως βάση για διαπραγματεύσεις. Η κυρία Πρόεδρος έχει ένα ισχυρό επιχείρημα. 75% των ε, ε, πολιτών της Ταϊβάν απορρίπτουν την συνέλευση του 1992. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η καθαρή πρόθεση και το δικαίωμα των ε, πολιτών της Ταϊβάν να ζήσουν σε ελευθερία και δημοκρατία πρέπει να γίνουν σεβαστά. Πρέπει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα η Κίνα της ύπαρξης της Δημοκρατίας της Κίνας, δηλαδή της Ταϊβάν, στην βάση ισότητας και χωρίς επιβολή όρων. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να δηλώσει την ισχυρή αντίθεσή της απέναντι στη χρήση βίας για την επίλυση διαφορών μεταξύ των δύο μερών και να τονίσει την ανάγκη σταθερότητας. Διακόπτη. Η κυρία νομίζω ότι το μήνυμά σας ωστόσο ήταν πάρα πολύ ε, καθαρό και μου επιτρέπετε να δώσω τον λόγο στον επόμενο που είναι ο κύριος Λάινεν εκ, εκ μέρους των ε, Δημοκρατιών και Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η Σοσιαλδημοκρατική Ομάδα αναγνωρίζει την πολιτική τη μιας Κίνας. Αυτό είναι και το light motif το οποίο έχουμε εφαρμόσει από πολλά χρόνια και εξακολουθούμε να το εφαρμόζουμε. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν μεγάλες συμπάθειε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και παροιμήν στην ομάδα μου δηλαδή για την Ταϊβάν, υπέρ της Ταϊβάν λόγω της λειτουργούση δημοκρατία στην περιοχή αυτή του κόσμου αλλά και λόγω της ένταξης της χώρας αυτής στα παγκόσμια οικονομικά και εμπορικά ρεύματα λόγω του ότι εκεί επικρατεί η οικονομία της αγοράς. Το Κοινοβούλιο κατ' επανάληψη έχει ταχθεί υπέρ της ιδέας οι διαφορές, η σύγκρουση μεταξύ των δύο μερών Κίνας δηλαδή και Ταϊβάν να επιληθεί μέσω μέτρων αποκατάστασης εμπιστοσύνης και διαλόγου. Ισχύει αυτή η αρχή ακόμη. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Η μόνη λύση που μπορεί να υπάρξει είναι πολιτική με τις διάφορες μορφές διαλόγου που θα επιτρέψουν μια προσέγγιση και στενότερη συνεργασία. Πολλοί έχουν ανησυχήσει μετά από την ομιλία του Προέδρου Xi Jinping που δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη η Κίνα να χρησιμοποιήσει ακόμη και βία. Ωστόσο θα πρέπει να διαβάσει κανείς προσεκτικά την ομιλία αυτή. Στην αρχή λέει ότι οι Κινέζοι δεν πολεμούν κατά άλλων Κινέζων. θεωρεί μάλλον ότι πρέπει να αντιταχθούν σε παρεμβάσεις έξωθεν και εννοεί πιθανότατα το ότι στην αντίθεση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας οι ΗΠΑ ίσως να χρησιμοποιήσουν μέσον πίεση στην Ταϊβάν. Ο Ξι Τζινπίνγκ είπε μια χώρα με δύο συστήματα. Αυτό μπορεί να το πει κανείς, αλλά υπάρχουν όντω διαφορετικά πολιτικά συστήματα τα οποία δεν προσεγγίζουν, αλλά μάλλον αποκλίνουν διακόπτει ο πρόεδρος το μικρόφωνο του ομιλητού. Λοιπόν, πολύ κύριε συνάδελφε, ούτε, ούτε θα θέλατε να γνωρίζετε πότε προβλέπετε να τελειώσουμε και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα μειώσω τον χρόνο του Catch the Eye και δεν θα κάνω Catch the Eye για οποιοδήποτε άλλο θέμα που πρόκειται να συζητηθεί διότι πρέπει να καλύψουμε τον χρόνο που έχουμε χάσει. Για 1,5 λεπτό λοιπόν Μπέντερ της ομάδας ECR. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Την χρονιά ο πρόεδρος της ε, Κίνας παρακολούθησε τα πυροτεχνήματα και επανέλαβε το status quo ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ταπέι. Για την ε, κινέζικη ελίτ έπρεπε να ξεχαστεί το τραύμα της Ταϊβάν. Υπάρχει όμως κλιμάκωση της κατάστασης εξαιτίας της ε, πίεσης του κινέζικου στρατού. Ο πρόεδρος τι εννοούσε με την ομιλία του εννοούσε ότι είναι εσωτερικό ζήτημα το ζήτημα της Ταϊουάν, ότι δεν αφορά μόνο τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ταϊβάν. Εδώ όμως πρόκειται για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις δικές μας τις αξίες. Και γι' αυτό πρέπει να στραφούμε προς το Πεκίνο για να καταλάβει, αλλά και προς την ΤΑΠΕΙ για να την στηρίξουμε απέναντι στην Κίνα. Ευχαριστούμε για δύο λεπτά εκ μέρους του Άλντε, Φαν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι η δημοκρατία της ε, Κίνας και συγκεκριμένα το κομμάτι της Ταϊουάν δεν ήταν ποτέ εξ ολοκλήρου τμήμα της. Αυτό σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί για το ότι η Κίνα έχει την κυριαρχία στην Ταϊβάν δεν θα στέκανε. Όμως και οι δύο πλευρές έχουν κρατήσει το status quo, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους και ασφάλεια στην περιοχή. Οπότε είμαι υπέρ του status quo, το οποίο όμως έσπασε από την ηγεσία της Κίνας και από τον πρόεδρο Xi Jinping που είπε ότι ακόμα και η βία μπορεί να είναι τρόπος για να ενωθεί η χώρα. Η Άλντε δεν δέχεται τη χρήση στρατιωτικής βίας, ούτε καν την απειλή της, ούτε οποιοδήποτε άλλο εκβιασμό. Ο κόσμος της Ταϊβάν πρέπει να μπορεί να καθορίσει το μέλλον του. Με τις Ηνωμένε Πολιτείε πρέπει να προστατεύσουμε την Ταϊβάν και τη δημοκρατία της. Η Κίνα θα πρέπει να γνωρίζει ότι η χρήση βίας και οποιαδήποτε άλλη πίεση θα έχουν σοβαρές συνέπειες για την ίδια την Κίνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φανμπάλεν. Τώρα για ένα λεπτό εκ μέρου των Πρασίνων ο κύριος Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν αλλάζει και γίνεται επιθετικότερη. Αυτό το δήλωσε άλλος ο ίδιος ο πρόεδρος Σι Πίνκ η απειλή του για χρήση στρατιωτικής βίας είναι εσφαλμένη. Όμως είναι ένα θέμα και το γεγονός ότι ασκεί πιέσεις οικονομική, διπλωματική η Κίνα στην Ταϊβάν. Οικονομική πίεση με το να παίρνει τους ε, οικονομικούς και εμπορικούς εταίρους της Ταϊβάν. Και βεβαίως αυξάνει και την ένταση στα στενά. Η δική μας πολιτική της μιας Κίνας είναι αποδεκτή μόνο εάν προβλέπει ειρήνη και από τα δύο πλευρά των κινέζικων στενών. Γι' αυτό και είμαστε αλληλέγγυοι με τη δημοκρατική Ταϊβάν. Ευχαριστώ κύριε Σόλτς, Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην εξωτερική πολιτική απέναντι στην Κίνα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφή κοινή θέση πολιτική της μιας Κίνας. Άρθρο 2 της συνθήκης της Λισαβόνας που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην διεθνή ειρήνη, στον αλληλοσεβασμό των εθνών και ούτω καθεξής. Δεν λέει τίποτε για έλλειψη ομόνιας. Κανές, σε κανένα δεν αρέσει η κλαγή των όπλων. Ούτε στην Καραϊβική, ούτε στα στενά της Ταϊβάν. Είναι περίπλοκη είναι περίπλοκε οι διαφορές. Δεν είναι δυνατόν να απλοποιηθούν τα πράγματα για αυτά γιατί αυτό είναι τακτική Τραμπ. Χρειάζεται διάλογος και αναζήτηση λύσεων. Με τη σωστή σειρά οφείλουν τα δύο μέρη να συνδιαλέγονται, να προωθηθεί ο διάλογος, τα περίπλοκα θέματα ε, του διεθνούς δικαίου πρέπει να συζητηθούν. Ορισμένοι μιλούν και για συμφωνίες Διακόπτει ο Πρόεδρος τον κύριο Σόλτς. Σας ευχαριστώ. Και πάλι για όσους ήλθατε με κάποια καθυστέρηση έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα χρόνου. Λόγω καθυστερήσεων έχουμε τροποποιήσει το πρόγραμμα. Θα κάνω λοιπόν το Catch the Eye το πολύ τρεις βουλευτές από κάθε πολιτική ομάδα και δεν θα κάνω catch the eye για, τις τα υπόλοιπα θέματα. Από τους, ε, μη, ε, ε, ο κύριος Επιτίδιος. Κύριε Πρόεδρε, από το 1949 όποτε έληξε ο εμφύλιος ε, πόλεμος ε, στην Κίνα ε, η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν ως κινέζικο έδαφος το οποίο πρέπει να επιστρέψει στην χώρα όπως επέστρεψε το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο. Επειδή όμως η Ταϊβάν θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί υπάρχουν συνεχώς τριβές μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Και με τις δύο χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχέσεις καλές τόσο εμπορικές κυρίως όσο και άλλης φύσεως. Γι' αυτό λοιπόν στη διαμάχη αυτή θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κοιτάξει να εξυπηρετήσει τα πολιτικά και οικονομικά της συμφέροντα. Όταν θεωρεί ότι πρέπει να συμπλέει με την Κίνα θα πρέπει να υποστηρίζει το δόγμα της ενιαίας Κίνας όταν όμω θεωρεί ότι τα συμφέροντά τη εξυπηρετούνται από τη συνεργασία με την Ταϊβάν, πρέπει να συνεργάζεται με την Ταϊβάν. Ευχαριστώ. Κύριο Πρέντα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις, στις, δηλώσεις του Xi Jinping υπάρχει κάτι φοβερό. Γιατί ένα κομμουνιστικό καθεστώς που θέλει να εκφοβήσει τους δημοκράτες γειτονέ του με προσφυγή στη βία οι αρχές του Πεκίνου έχουν ερμηνεύσει λάθος το αποτέλεσμα των εκλογών της Ταϊβάν που έγιναν τον Νοέμβριο του 2018. Γιατί σε καμία περίπτωση στην προεκλογική εκστρατεία το θέμα της επανένωσης με την Κίνα δεν τέθηκε. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Οι Ταϊβανέζοι δεν έστειλαν ένα μήνυμα στον Xi Jinping. Μίλησαν για τα εσωτερικά τους θέματα. Και οι περισσότεροι από αυτούς, η συντριπτική πλειοψηφία, είναι κάθετα αντίθετη στην ιδέα μία χώρα, δύο συστήματα. Αυτό που επιθυμούν πάνω απ' όλα οι Ταϊβανέζοι είναι να προστατεύσουν τη δημοκρατία τους, το κράτος δικαίου και τις ελευθερίες τους. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι άγνωστα για ένα κομμουνιστικό καθεστώς που αντίθετα εκείνο τι κάνει συλλαμβάνει όσους ε, υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσους ε, ζητούν ε, και με φήμωση της ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας έκφρασης. Υπάρχουν όλο και μεγαλύτερε εντάσει στα στενά τη Ταϊβάν. Προτείνω λοιπόν μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πάει στην Ταϊβάν ε, το συντομότερο δυνατόν, ούτω ώστε να δούμε ποια είναι η κατάσταση και να υποστηρίξουμε τη δημοκρατία τη ε, Ταϊβάν. Ευχαριστώ. Ο κύριο Καπούτο, συγγνώμη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε οι ε, τεταμένες ε, σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν περαιτέρω. Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Jinping επανέλαβε ότι θα πρέπει να ενωθεί το νησί με την Κίνα με βάση το, ε, τη φόρμουλα μία, ένα κράτος, δύο συστήματα. Και δεν αποκλεί σε κάποια φάση να υπάρξει και στρατιωτική χρήση και ενδεχομένω μάχες. Αυτό που περιέπλεξε τα πράγματα είναι η παρεμβολή του Τραμπ στα, και η χρήση της, η σύνταξη της Αμερικής με την Ταϊπέη και, και το γεγονός ότι έδωσε στρατιωτικό υλικό παρά την απόσταση. Εμεί θέλουμε παρόλα αυτά μια ειρηνική Κίνα. Είναι προς το συμφέρον όλων μας. Δεν θέλουμε ένταση. Και αυτή η ανάγκη γίνεται όλο και πιο προφανή σε ένα όλο και πιο συγκρουσιακό κόσμο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις σχέσεις που έχουμε με την Κίνα και με την Ταϊβάν για να διαπραγματευτούμε μία σχέση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούκαν για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Με ανησυχεί κάτι που όλους πρέπει να μας ανησυχεί. Είναι η ένταση, η κλιμακούμενη στα στενά και πρέπει να ζητήσουμε αποκλιμάκωση και όχι να ρίχνει λάδι στη φωτιά με την ομιλία του ο πρόεδρος Xi Jinping. Είναι προς το συμφέρον όλων η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή. Πρέπει να στηρίξουμε οποιαδήποτε επίλυση διαφορών ειρηνικά, με επικοδομητικό διάλογο, με συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Πρέπει να είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πιστεύει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε επιθετικά μέτρα για να λυθεί αυτή η κατάσταση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την ασφαλεία, ε, για την ασφάλεια, συγγνώμη, για το κοινωνικό και οικονομικό σύστημα της Ταϊουάν. Το θέμα της επανένωσης είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να συζητιέται. Είναι προς το συμφέρον μας να ζητήσουμε και από τις δύο πλευρές να βρουν τρόπο να ε, εντατικοποιήσουν το διάλογό τους για να βρεθεί μια ειρηνική λύση. Και πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε τις αξίες, τις κοινέ που έχουμε με την Ταϊουάν και να τη στηρίξουμε στην περιοχή. Θέλω επίσης να ζητήσω από την είπα το εκπρόσωπο την κυρία Μογκερίνη να, να χρησιμοποιήσει όλα τα διπλωματικά μέσα που διαθέτουμε για μια βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκόμες έχει τώρα το λόγο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήλια κατά της Ταϊβάν στην περιοχή από πολλές περιοχές εκεί γύρω. ήθελε να υποστηρίξει ένα κράτος δικαίου η Ταϊβάν, γι' αυτό και ζήτησε την ανεξαρτησία της, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην Κίνα. Δυστυχώ ό,τι θέλει να κάνει τα Ιβάν το απαγορεύει η Κίνα και την πιέζει. Αν θέλουν αυτό που θέλουν οι κάτοικοι της Ταϊβάν και το ζητούν ειρηνικά, θα πετύχουν το στόχο τους. Γιατί η βία, πρέπει να πούμε, είναι πάντα σε βάρος και θα είναι και σε βάρος της Κίνας αν την ασκήσει. Έχει μεγάλη σημασία η παγκόσμια ειρήνη. Πρέπει να δρούμε βάσει του διεθνούς δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ακολουθήσει οποιοδήποτε άλλο δρόμο από τον ειρηνικό, γιατί αλλιώς θα προσβληθεί στα Ηνωμένα Έθνη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Στις 2 ε, Ιανουαρίου του 2019 έκανε μια ομιλία ο Xi Jinping και δημιούργησε μια πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση σε όλους τους εταίρους στην περιοχή. Οικονομικά και στρατηγικά είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμβαθύνει στις σχέσεις της με την αναπτυσσόμενη αυτή περιοχή. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε είχαμε την συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ίντα ήταν με τη Σιγκαπούρα και με το Σιγκαπούρ και το Βιετνάμ. Διαπραγματεύσεις γίνονται με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Όμως, με την ε, Νότια Ασία δεν έχουμε κάνει τίποτα με την Ταϊβάν, γιατί την εμποδίζει η Κίνα. 30 χρόνια διμερών σχέσεων γιορτάσαμε όμως το 2018 οι επενδύσεις είναι μόνο 1,9% από πλευρά τη Ταϊβάν, ενώ βέβαια τη Κίνα πολύ μεγαλύτερε. Πρέπει να στηρίξουμε την δημοκρατία και την ελευθερία. Πρέπει, διακόπτει ο πρόεδρο, συγγνώμη, αλλά έληξε ο χρόνο σα. Λάγκεν, για ένα λεπτό παρακαλώ, ο κύριος Λάγκεν. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε ως πρόεδρος της ομάδας φίλων ευχαριστώ τις και τους συναδέλφους που είναι υπέρ και αγωνίζονται υπέρ της δημοκρατικής Ταϊβάν. Συμφωνώ με τον Πιούτι Κόφερ. Από το 1992 είναι η πολιτική τη μιας Κίνας. Αλλά αυτό μόνο εφόσον υπάρχει ειρήνη. Και εντυπωσιάζομαι που ο κύριος Λάινεν, πρόεδρος της αντιπροσωπείας για σχέσει με το Κινέζικο Κοινοβούλιο, που τώρα έχει αποχωρήσει από την αίθουσα, το θεωρεί μια απλή δήλωση. Όχι, ήταν μια δήλωση η ε, ε, πολιτικής αξίας που ήταν μάλιστα, δηλαδή αυτή η δήλωση του Xi Jinping που την έκανε ενώπιον υψηλών αξιωματούχων της κυβέρνησής του. Αν συνεχίσει με την πολιτική αυτή η Ευρώπη δεν έχει παρά μια μόνο λύση. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την Ταϊβάν. Άλλη γλώσσα δεν αντιλαμβάνεται η Κίνα. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ε, Ταϊβανέζους ώστε να μην μπορούν οι Κινέζοι να τους πετάνε έξω από διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Ευχαριστώ. Και έλα ένα λεπτό. Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Είναι μια δημοκρατία η Ταϊβάν δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ούτε για το Πεκίνο, ούτε για τον υπόλοιπο κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι η Κίνα θέλει να απορροφήσει την Ταϊβάν και ότι είναι μια κομμουνιστική δικτατορία που είναι ε, υπεύθυνη για τη φυλάκιση και θανάτωση δεκάδων χιλιάδων πολιτών της που καταπιέζει τις μειονότητες, τα πολιτικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Η προειδοποίηση του Προέδρου ότι δεν θα διστάσει ακόμα και να καταφύγει σε βία είναι δυσίωνη. 23 εκατομμύρια τα Ιβανέζοι έχουν κάνει μια δημοκρατική επιλογή. Θέλουν ελεύθερη κοινωνία. Αυτό ψήφισαν. Πριν επιμείνουμε για επανένωση, η Κίνα θα πρέπει ίδια να μεταρρυθμιστεί, να γίνει δημοκρατική κοινωνία η οποία θα σέβεται τις ελεύθερες επιλογές όλων των πολιτών της. Ο κύριος Δίας Τεμέρα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κάτω από την ηγεσία του Xi ε, Jinping ε, αυξήθηκε η πίεση απέναντι στην Ταϊβάν ε, για να αλλάξει το καθεστώς στα στενά της Φορμόζας και να ε, ανατραπεί η ευαίσθητη ισορροπία της περιοχής σε επιχρόνια ε, είχε το καθεστώς του παρατηρητή η Ταϊβάν και Παρόλα αυτά η Κίνα έστειλε στρατεύματα, φρεγάτες, ε, αεροπλανοφόρα στα στενά της Ταϊβάν ε, ή την απομόνωνε στα διεθνή φόρουμ. Δεν ε, αποκλείει να χρησιμοποιήσει την βία η Κίνα για την επανένωση. Η Ταϊβάν όμως είναι μία ε, δημοκρατία. Δέστε τι λέει η πρόεδρος Σάι. Μία δημοκρατία μπορεί να επιβιώσει εάν όλοι με διαφορετικές ιδέες δουλέψουν μαζί για το κοινό καλό. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δεσμευτεί περισσότερο και να στηρίξει την δημοκρατία στην Ταϊβάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κλείνουμε τη συζήτηση. Πάμε στο Catch the Eye. Έχουμε καθυστερήσει, το ξαναλέω. Δεν μπορώ να δεχτώ όλα τα αιτήματα για το Catch the Eye. Ο κύριος Φαρία για ένα λεπτό. E Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Πεκίνο προσπαθεί να προσαρτήσει τη Φορμόσα και εδώ και χρόνια το έχει δείξει ότι θα το κάνει και αν όχι αλλιώς με τη βία. Η ε, εισβολή, έλεγχη, αεροπλάνη είναι πολύ συνδυσμένα πράγματα στα στενά της Ταϊουάν. Πιέζουν και οι εκστρατείες τους έχουν σαν στόχο η Ταϊουάν σιγά σιγά να αρχίζει να βλέπει με πιο καλό μάτι την ένωση με την Κίνα και αυτή την πολιτική μια ε, μιας χώρας δύο συστημάτων που πιστεύω ότι είναι λάθος. Λοιπόν εμείς θέλουμε να στηρίξουμε την Ταϊβάν που είναι μια πιο ανοιχτή δημοκρατία και οικονομικά πολύ σημαντικό εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρξει αυτοσυγκράτηση και από τις δύο πλευρές. Να μην δεχτούμε τις απειλές για τη χρήση βίας. Η Κίνα θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε κίνηση πρωτοβουλία που θα θέσει σε κίνδυνο το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα και το λαό τη Ταϊβάν. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, λέει ο κύριος Τροκεύσκη. Άκουσα αυτά που είπαν οι κύριοι Κούκαν, Λάγκεν, Πρέντα Συμφωνώ με αυτά που είπανε. Δύο πράγματα όμως έχω να προσθέσω. Ότι τα Ιωάννη έχει κάνει τεράστιο δρόμο για να βελτιώσει τις σχέσεις της με τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Και η Κίνα θα έπρεπε να το εκτιμήσει αυτό και να σταματήσει να θεωρεί την Ταϊουάν δικιά της επικράτεια. Έπειτα μην ξεχνάμε την κληρονομιά και την επιτυχία της Ταϊουάν, πολιτιστικά, τεχνολογικά, υπάρχει σεβασμό απέναντι στην Ταϊβάν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε. Σέντροβα, ένα λεπτό τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Κίνα θέλει την Ταϊβάν κομμάτι της επικράτειάς της. Εγώ βλέπω ότι το θέλει αυτό η Κίνα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλά κοινά ανάμεσα στην Ταϊουάν και την Κίνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να προσαρτιστεί στην Κίνα η Ταϊουάν. Η Ταϊουάν έχει ελεύθερη οικονομία, έχει δημοκρατία και φέτο ο πρόεδρο τη Κίνα, η Τζιπίνγκ, μίλησε πολύ επιθετικά για το δεχόμενο προσχώρηση τη Ταϊουάν στη λαϊκή δημοκρατία τη Κίνα, ακόμα και με στρατιωτική βία. Αυτό είναι εκφοβισμό από πλευρά ισχύω και δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Η Ταϊβάν αποτελεί ένα παράδειγμα μια λειτουργούσα δημοκρατία με τι ίδιε αξίε όπω και η Ευρωπαϊκή Ένωση και αξίζει την πλήρη στήριξή μα και αναγνώρισή μα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζω να στηρίξει τα Ταϊβάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βασίζεται συνέχεια στι ΗΠΑ. Πρέπει να καθίσουμε, σταθούμε και εμεί στα πόδια μα και να παίξουμε το διεθνή μα ρόλο. Ευχαριστούμε. Άλλο ένα. Σακβάρη, παρακαλώ. για να καταλάβουμε το μήνυμα την πρωτοχρονιά που έστειλε ο πρόεδρος της ε, Κίνας, θα πρέπει να δούμε και το πλαίσιο και το περιεχόμενο και τι σημαίνει μια νέα πολιτική για την Ταϊβάν και τι σημαίνει για τη σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο, υπάρχει απόκληση από τον τότε πρόεδρο του 2009. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, ο Xi Jinping δεν μιλάει με αμφισημία για το, τη συνένεση του 1999. Ε, χρησιμοποιεί την ίδια λογική με αυτή που χρησιμοποιεί για το Χονγκ Κόνγκ. Ένα κράτος, δύο συστήματα. όμως ε, η Ταϊβάν ποτέ δεν δέχτηκε τη συνένεση του, του 1992. Η Κίνα θα πρέπει να δεχτεί την πραγματικότητα της ύπαρξης της ε, Ταϊβάν των 23 εκατομμυρίων πολιτών που θέλουν ένα ελεύθερο καθεστώς. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαφορές αυτές η ειρηνικά η Κίνα. Θα πρέπει να κάνουν συζητήσεις οι δύο κυβερνήσεις. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, ο κ. Σόλα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, όταν ε, εξέφρασε την ομιλία του μίλησε για τη χρήση όλων των απαραίτητων μέτρων για να προωθήσει την πολιτική της μίας Κίνας θα πρέπει να μας ανησυχεί όλους μας. Παίζονται πάρα πολλά. Για να ρυθμιστούν οι πολιτικές διαφορές και οι πλευρές πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Δεν θα πρέπει καταρχάς να φυστούμε κόπο για να γίνουν πραγματικά επίσημοι διάλογοι. Όλα Όλε οι διαφορές θα πρέπει να λυθούν ε, με ειρηνικό τρόπο, με βάση το διεθνές δίκαιο και με την αρχή της ισότητας. Πιστεύω ότι η δέσμευση των, του λαού τη ε, Ταϊβάν στην ελευθερία και στην δημοκρατία και προ ένα δημοκρατικό σύστημα που έχουν χτίσει στη χώρα τους θα πρέπει να γίνει σεβαστό και να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ ο Επίτροπος, για τα τελευταία του λόγια. Πρόεδρε, ήταν μια πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Καταλήγω και κρατάω από αυτή τη συζήτηση ότι όλοι θεωρούμε ότι η πολιτική για τη μία και ενιαία Κίνα μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Παρ' αυτά θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας με την Ταϊβάν όπως ε, καθορίζεται η στρατηγική όπως καθορίζεται από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016 για την ε, σχέση με την Ταϊβάν. Θα πρέπει να δεσμευτούμε περαιτέρω, ούτως ώστε το status quo να παραμείνει ο κανόνας στα στενά της Ταϊβάν. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που δίνω στο ρόλο του Κοινοβουλίου γιατί βάζει αυτό το θέμα ε, μεταξύ άλλων στην ατζέντα για τα διεθνή θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχει ολοκληρωθεί εδώ η συζήτηση. Θα δώσω μισό λεπτό για να μπορέσει να καθίσει η Επίτροπος κ. Μάλμστρομ. Με την ευκαιρία όμως θα επαναλάβω ότι για λόγους χρόνου δεν θα διεξαχθεί η διαδικασία Catch the ούτε μετά από την επόμενη συζήτηση και καμία άλλη. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν είναι κάτι που επιθυμώ. Δυστυχώς αναγκάζομαι να υποκριθώ στην πραγματικότητα. Δήλωση τώρα της Επιτρόπου. Έχετε το λόγο κύριε Επιτροπέ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάντοτε στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακόμη και εάν ο χρονισμό της παρούση συζητήσεω πράγματι υπήρξε πρόκληση για μας. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την έγκριση της κοινή δηλώσεω των Προέδρων Γιούνκερ και Τραμπ μπήκαμε σε μια νέα φάση των σχέσεων μα με τι Ηνωμένε Πολιτείε που είναι και ο πρώτος επενδυτικός και οικονομικός εταίρος μας και δώσαμε μια θετική ατζέντα. Έχω συναντηθεί με τους Αμερικανούς ομολόγους μέχρι τότε πολλές φορές για να εφαρμόσουμε το κοινό πρόγραμμα το οποίο καταστρώσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι. Έχουμε εντοπίσει μελλοντικέ οδούς για εθελοντική συνεργασία με τις ΗΠΑ... και για ε, τομείς όπως φαρμακευτικά, ιατρικές συσκευές και κυβέρνο ασφάλεια... Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί ως τώρα απηχείται και σε έκθεση που δημοσίευσαμε σήμερα το πρωί και είναι διαθέσιμη να την αναγνώσετε. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων όπως η μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου καθώς και άλλες προκλήσεις κρατικού καπιταλισμού. Για παράδειγμα εμπόριο ε, σόγιας, υγροποιημένου φυσικού αερίου και άλλα που έχουμε περιλάβει στην κοινή δήλωση του Ιουλίου. Επίσης, ασφάλεια παροχής ενέργειας και ασφάλεια για τους γεωργούς μας. Πριν από δύο εβδομάδες εξέδωσε δύο συστάσεις αφενός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφενός για, τις, ε, ε, για τους δασμούς που είναι και προφανείς και δεν περιλαμβάνει τα γεωργικά προϊόντα όπως και συμφωνηθεί άλλωστε τον Ιούλιο η προτινόμενη εντολή για την ε, αξιολόγηση της συμμόρφωσης χρειάζεται κάποια εξήγηση. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καθιερωμένες πρακτικές για την ε, αξιολόγηση της συμμόρφωσης. παραγωγοί μπορούν να διαθέτουν προϊόντα στις αγορές μόνο εφόσον αυτά συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις προϊόντα μη ασφαλή ή που δεν συμμορφώνονται δεν θα πρέπει να φτάνουν μέχρι τα χέρια ανύποπτων καταναλωτών. Αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται υποχρεωτική αξιολόγηση και επιστοποίηση από τρίτους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό έξτρα κόστος, χωρίς και την βελτίωση του προϊόντος, τη βελτίωση της ασφάλειας του προϊόντος. Έχουμε λοιπόν συστάσεις για conformity assessment για να μειωθεί το περιττό κόστο, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουμε ότι διατηρείται το επίπεδο προστασίας. Οι δύο συστάσεις εκπληρούν τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε τον Ιούλιο. Αναγνωρίζουμε ότι η πρόοδο στι διαπραγματεύσει με την κυβέρνηση Τραμπ είναι δυνατόν να γίνει μόνο σε επιμέρου project τα οποία συμφωνούν και οι δύο πλευρέ. Έχουμε αρχίσει λοιπόν τι προσπάθειε αυτέ ήδη από τον Ιούλιο θα οδηγήσουν σε σημαντική ατζέντα με ε, και για τις δύο πλευρές. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την ατζέντα για με τις ΗΠΑ και είναι σημαντικό να μην επανέλθουμε σε έναν καταστροφικό κύκλο ε, μέτρων περιοριστικών του εμπορίου. Ταυτόχρονα πρέπει να δηλώσουμε σαφώς, σαφώς ότι κάθε προσπάθεια υπέρβασης της κοινή δήλωσης και μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν είναι για την ώρα σκόπιμη. Οι ΗΠΑ Πολιτείες δεν είναι διατεθειμένες να ε, συμφωνήσουν για ευαίσθητα θέματα όπως δημόσιες ε, προσφορές ή γεωγραφικές ενδείξεις. Ένα από τα πιο σημαντικά διδάγματα λοιπόν από τις ε, διαπραγματεύσεις για την συνθήκη TTIP είναι ότι Μία ατζέντα μαζί με τις ΗΠΑ είναι καλύτερα να διεξάγεται με απόλυτη διαφάνεια και εκτός πλαισίων FTA. Υπάρχουν τομείς όπου θα είναι δύσκολο να γίνουν βήματα. Οι προσπάθειές μας λοιπόν θα αποδώσουν καρπού αν προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για την μεταρρύθμιση ορισμένων κανόνων του παγκόσμιου εμπόριου. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και θα είμαστε πανέτοιμε για να αντιπαντήσουμε εάν οι ΗΠΑ δεν σεβαστούν τι δεσμεύσεις που ανέλαβαν τον Ιούλιο και αν λάβουν και άλλα περιοριστικά μέτρα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το σενάριο όμω δεν θα είναι κάτι που θα επιλέξουμε εμεί. Αναμένω με ενδιαφέρον την συζήτηση και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε καθώς και εσάς κυρίες και κύριοι που με παρακολουθήσατε. Επαναλαμβάνω, λέει ο Πρόεδρο, ότι για λόγου χρόνου δεν θα διεξαχθεί η διαδικασία CatchDI ούτε για την παρούσα συζήτηση ούτε και για οποιαδήποτε θα ακολουθήσει. Εξ ονόματο τη ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, για τρία λεπτά ο κύριο Χάνσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε με ανθρώπου, οι οποίοι λένε τα δικά μου δικά μου αλλά τα δικά σα δικά μα. Δεν μπορούμε λοιπόν να βασιστούμε σε κάτι τέτοιο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να μειώσουν το δικό τους έλλειμμα. Πιέζουν για τα γεωργικά προϊόντα και για τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις. Η δική τους στόχη είναι εντελώ διαμετρικά αντίθετη από αυτούς που τον Ιούλιο που μας πέρασε συνονοήθηκε ο πρόεδρος Γιούγκερ. Μην ξεχνάμε ότι όταν εμείς συζητάμε δεν οδηγούμαστε σε εμπορικό πόλεμο. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι φιλόδοξες. Η Γεωργία δεν είναι δυνατόν ποτέ να μπει σε συζήτηση. Πρόκειται για 15 εκατομμύρια ε, θέσεις η συμφωνία αυτή, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να φοβούμαστε να συζητάμε με θετικούς στόχους. Αυτή τη σύγκρουση Α τη σταματήσουμε και α δείξουμε ότι η συνεργασία είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε σε εμπόριο βασισμένο σε κανόνες. Ποτέ δεν πρέπει να διαπραγματευόμαστε με το φόβο, αλλά να μην φοβόμαστε ποτέ να διαπραγματευτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρενά τώρα για δύο λεπτά εκ μέρου των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πράγματι ποτέ δεν θα καταλάβω ε, γιατί επιμένετε σε διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο Τραμπ. Το 2018, ενώ αποφάσισε ο Τραμπ για δασμούς παράνομους για το χάλιβα και το αλουμίνιο της Ευρώπης, λέγατε ποτέ δεν θα διαπραγματευτώ υπό την απειλή. Και όμως, οι δασμοί αυτοί πάντα απειλούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ξακολουθεί να υπάρχει απειλή και εσείς μπαίνετε σε διαπραγματεύσεις. Αυτό προτείνεται στο Συμβούλιο. Ενώ αμφισβητεί το πολυμερές σύστημα ο Τραμπ, το οποίο τόσο πολύ θέλουμε εμείς στην Ευρώπη, εσείς αποφασίζετε εκ νέου διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ. Μα δεν δέχεστε έτσι την διμερή λογική, τη λογική των διμερών διαπραγματεύσεων. Εμείς δεν θέλουμε να αρνηθούμε τις δεσμεύσεις μας ε, για ε, τις συμφωνίες ε, των Παρισίων. Εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Και έπειτα, όταν βλέπουμε την ελάχιστη προσφορά που κάνετε στις διαπραγματεύσεις και τις ευρείες προσφορές που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, τελικά τι κοινό σημείο θα βρείτε με την Αμερικανική κυβέρνηση σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το να αρχίζουν διαπραγματεύσεις για μας είναι τακτικό λάθος, πολιτικό λάθος και ελπίζουμε το Σεβούλιο να μην δεχτεί την εντολή που προτείνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εκ μέρου του ECR, κυρία Μακλάρκιν, δεν είναι εδώ από ό,τι βλέπω, οπότε επόμενος ομιλητή είναι η κυρία Σχάκε. 1,5 λεπτό παρακαλώ, εκ μέρου τη ομάδα ALDE. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Ορισμένοι περιμέναμε αυτή την συζήτηση να την κάνουμε το ψήφισμα του Μαρτίου. Αλλά την κάνουμε τώρα. Δυστυχώ, κάνουμε μια συζήτηση για τι εμπορικέ σχέσει με του Αμερικανού ε, σε καθημερινή, σε εβδομαδιαία βάση. Δυστυχώ. Φτάσαμε σε μια ανακοχή πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά οι παράνομοι δασμοί για, τα, για το χάλιβα και το αλουμίνιο στην Αμερική παραμένουν και ε, υπάρχει το, το πάνελ αυτό στον ΠΟΕ. Ε, αυτή τη βδομάδα ο Τραμπ απείλησε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν ακολουθήσει τους Αμερικανούς για την απαγόρευση του εμπορίου με το Ιράν θα έχει επιπτώσεις. Νομίζω ότι το εμπόριο θα πρέπει να γίνεται με βάση κάποιου κανόνε, με κάποια ατζέντα. Με κάποιου εταίρου όπω ο Καναδά, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία που έχουν την ίδια άποψη για να αυξάνουμε τον πύχη, να προστατεύουμε τα δικαιώματα, το περιβάλλον, ε, τα υψηλά πρότυπα, τι αρχέ και μία νέα δέσμη κανόνων για, εμπο... για το εμπόριο στην ψηφιακή εποχή. κατοσορίζω την ε, πρωτοβουλία τη περασμένη εβδομάδα για το ηλεκτρονικό εμπόριο στον ΠΟΕ. Ζητάω όλου αυτού του συμμάχου τη ΗΠΑ να ε, συμπαραταχθούν μαζί μα για τη δουλειά να ενισχύσουμε το πολυμερέ ε, σύστημα εμπορίου. Και υπάρχουν πολλοί αυτοί. Στο μεταξύ, ε, συνομιλώντα με την Αμερικανική κυβέρνηση, υποστηρίζω την προσπάθειά σα, Επίτροπη, να κάνετε στοχευμένε συζητήσει ε, για του δασμού, ε, για τα βιομηχανικά αγαθά, αλλά όχι για τα γεωργικά προϊόντα και για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Δεν είναι ιδανικό, αλλά είναι η καλύτερη επιλογή προς το παρόν και είναι σημαντικό να κρατήσουμε το διάλογο ανοιχτό. Ευχαριστώ από τους πράσινους για 1,5 λεπτό ο, Ζαντό, ο κύριος Ζαντό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, σήμερα το βράδυ ε, δείξατε μια φοβερή ικανότητα μας ε, διηγήστε παραμύθια. Μετά από ένα μήνα για την επανεκκίνηση αυτών των συζητήσεων, τελικά μιλάμε για μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που θα έχουμε τις ΗΠΑ Πολιτείες. Αλλά ευτυχώς επί μήνες οι Ευρωπαίοι ηγέτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσεί ακόμα μα είχατε πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διαπραγματευτούμε με το πιστόλι στον κρόταφο. Πού είδατε ότι ο Ντόναλτ Τραμπ κατέβασε το όπλο αυτό και δεν μας ε, ε στοχεύει. Για τα αυτοκίνητα, για τον ε, Χάλιβα, μας απειλεί. Απειλεί την παγκόσμια πολυμερή τάξη. Εμείς είμαστε οι καλοί μαθητές ε, της δήλωσης του Ιουλίου, λέτε. Τι κάνουμε, εισάγουμε περισσότερο πετρέλαιο και σχιστολιθικό αέριο. Είμαστε οι καλοί μαθητές. Ε, βάλετε, να βάλετε και διπλασιάστε τις εισαγωγές ε, μεταλλαγμένης σόγιας από τις ΗΠΑ. Και με το μαγικό ραβδάκι τροποποιείτε την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων ε, με τον Καναδά ήταν από την, τα κάψιμα από, ε, από άσφαλτο ενώ με τους Αμερικανούς είναι με τη, με σόγια. Έτσι διαπραγματεύεστε κατά τον, του κλίματος ε, αυτά τα πράγματα που κάνετε είναι ό,τι να είναι και θα πρέπει να σταματήσετε. Θα δώσω το, το λόγο την εκπρόσωπο του ECR για 1,5 λεπτό. Uh- Δεν ήσασταν πριν εδώ. Πάρτε τώρα το λόγο. Είσαστε αντιπρόεδρος της, του ομίλου Rugby. Ε, σας ευχαριστώ που μας στηρίζετε. Ε, σήμερα όμως συζητάμε κάτι πολύ σημαντικό. Ε, η ECR θέλει ελεύθερο εμπόριο με όλους τους εμπορικούς εταίρους και κυρίω με το μεγαλύτερο, τι ΗΠΑ εμπορικό εταίρο. Υποστηρίξαμε τι διαπραγματεύσει TTIP και, τις προτιμήσεις, και η προτίμησή μα είναι να διαπραγματευόμαστε ευρείε ε, συμφωνίε ε, ελευθέρου εμπορίου, απελευθέρωση τη υπηρεσία ε, στι κρατικέ προμήθειε. Δεδομένου του σημερινού κρατικού εμπορίου και των κυρώσεων, καλωσόρισα την συμφωνία με τι ΗΠΑ του Ιουλίου να μην επιβληθούν περαιτέρω δασμοί στα πράγματα τα οποία είναι εκτό διαπραγμάτευση, στα προϊόντα που είναι εκτό διαπραγμάτευση και εμεί υποστηρίζουμε την Κομισιόν για να συνεχίσει τι διαπραγματεύσει με τι ΗΠΑ. Το να έχουμε δύο χωριστέ συμφωνίε, μία για του δασμού και μία για τα βιομηχανικά αγαθά και μία άλλη για την αξιολόγηση ε, την αξιολόγηση συμμόρφωσης. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια διαρθρωμένη διαπραγμάτευση. Για τη διαπραγμάτευση για του ε, βιομηχανικού δασμού. Ευτυχώ, η εντολή τη Κομισιόν για τι έχει και προϊόντα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους εξαγωγείς και στις δύο μεριές του Ατλαντικού. Και θα εξασφαλίσει ε, την ε, συμμόρφωση οποιασδήποτε συμφωνίας με τον ΚΑΤ. Ε, οι διπλές δια, διαδικασίες για να αποδείξουμε τη συμμόρφωση είναι τρομερό εμπόριο, εμπόδιο στις εξαγωγές και για μας και για τους Αμερικανούς. Να προσθέσω και κάτι άλλο, μια προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις. Δεν μπορεί να είναι επιτυχής χωρίς τους δασμούς για το χάλιβα και το αλουμίνιο, οι οποίες οι οποίοι δασμοί πρέπει να μηδενιστούν. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό εξ ονόματο Ενωτική Αριστερά, ο κύριο Σόλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εσεί κύριε Επίτροπε, είμαστε υπέρ του νόμου και ηθικού εμπορίου. Είπατε ότι δεν θέλετε ε, περίστροφο στον κρόταφο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση του παγκόσμιου εμπορίου παραμένει κάπου χαμένη στην ομίχλη. Υποβάλατε σχέδιο εντολή στο Συμβούλιο που είναι είτε ανηλικρινέ είτε μη ρεαλιστικό. Δεν θα μπορέσετε ποτέ να ανταποκριθείτε. Ο Τραμπ δεν πρόκειται να αναλάβει δεσμεύσει να μην επιβάλλει ποτέ δασμού στο μέλλον. Θα προσπαθήσει να περιλάβει στις συμφωνίες και τα αγροτικά προϊόντα, γιατί αυτή είναι η εντολή που του έχει δώσει το Κογκρέσο ως fast track. Το να αντιταχθείτε σε αυτό θα έχετε καθυστερήσει ήδη 8 μήνες. 77% μερίδιο αγοράς ενώ πριν από τη συμφωνία ε, Τραμπ-Γιούνκερ ήταν 9% και μιλούμε για την ε, χρήση αμερικανικής σόγιας για το ευρωπαϊκό βιολογικό δίζελ. Αυτό που χρειάζεται είναι έντιμη όρη προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Η FTD, δύο λεπτά, η κυρία Μπέκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν πέντε χρόνια άρχισα να... τη θητεία μου στο Κοινοβούλιο με μία ερώτηση. Γιατί τα έγγραφα της TTIP είναι μυστικά. Έχουμε νέο TTIP ε, πια, αλλά τα έγγραφα δεν είναι μυστικά. Ε, έχουμε μια πιο λεπτή στρατηγική. Τα έγγραφα δεν είναι πάντα δημόσια, αλλά ό,τι δημοσιεύεται είναι λευκό. Έχετε μία ε, σελίδα και καμία λεπτομέρεια για τι διαπραγματεύσει δύο μεγαλύτερε οικονομίε του κόσμου. Ε, δεν θα αγγίξει η συμφωνία, όπω είπατε, ε, τι γεωργίε, δεν, θα δεν θα εισάγουμε κρέα με ορμόνε ή γαματαφόμικρον. Αλλά ποιε είναι οι αποδείξει, στα λόγια σα. Έχουμε, εν πάση περιπτώσει, δύο εντολέ με τόσο γενικόλογια, ε, γενικόλογη περιγραφή που δεν αισθάνομαι ήρεμη και καθησυχασμένη. Πριν από λίγους μήνες, μάλιστα, είχατε δηλώσει ότι δεν θέλετε να διαπραγματευτείτε υπό την απειλή αμερικανικών δασμών, αλλά τώρα τι κάνετε, διαπραγματευόσαστε. Υποτίθεται ότι μας πουλάτε την επικοδομητική σας ε, στάση, αλλά οι Αμερικάνοι μας τσακίζουν με τους δασμούς ε, στο χάλιβα και στον αλουμίνιο. Επίσης, μας υποχρεώνουν να αγοράσουμε τη σόγια τους και τώρα ε, μας απειλούν με περαιτέρω δασμούς στα αυτοκίνητα. Επομένως, το περιβόητο ε, πιστόλι στον κρόταφο είναι πάντα ε, στον κρόταφό μας. Εγώ διάβασα όλα τα σχετικά έγγραφα είναι ε, όλα όσα λέγονται. Οι Αμερικανοί θέλουν ελεύθερη πρόσβαση, θέλουν να μπουν στις κρατικές μας προμήθειες, χωρίς εμείς να μπορούμε να επενδύσουμε στις δικές τους. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεν θα συμφωνήσουμε μέχρι η Αμερική να δείξει καλή θέληση και να σταματάει την, τις απειλές. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό, κύριο Ζαμέκ, μέρους του ΙΕΝΕΦ. Ή κύριε Ζαμέκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ή που μας λέτε ότι δεν ξέρετε, ή δεν ξέρετε τι μας λέτε. Λέτε ότι θα συμπεριληφθούν και τα προϊόντα τη θάλασσα στι διαπραγματεύσει. Ναι, αλλά οι ειδικέ σχέσει που έχουν οι με το Μεξικό και τον ε, Καναδά ε, θα ανοίξουν τι πόρτε στην είσοδο των Αμερικανικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά με το εφέ κοκτέιλ e που γνωρίζουμε. Μπορούμε λοιπόν να αναρωτηθούμε. Μήπω θα έπρεπε να εμποδίσουμε το κύριο Γιούνκερ να πηγαίνει και χωρίς εντολή να διαπραγματεύεται την εισαγωγή τόσων τόνων σόγιας Όπω το έκανε. Όχι, τελικά εμεί δεν αποφασίζουμε για τίποτα, ούτε για την υγεία, ούτε για την προστασία, ούτε για την διατροφική κυριαρχία. Η κυρία Χουμπινέρ, τώρα για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι διατλαντικές σχέσεις δεν είναι μόνο με μία κυβέρνηση, δεν αρχίζουν και τελειώνουν σε, σε αυτήν και μόνο την κυβέρνηση. Η εμπορική στόχοι, θετική εμπορική στόχη είναι κάτι πολύ σημαντικό για να ενισχυθούν οι δεσμοί μας. Λέτε κύριε Επίτροπε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την περιορισμένη εμπορική συμφωνία με, ε, τον, ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείες ακόμα και αν έχουμε μια πολύ περιορισμένη ημερήσια διάταξη αλλά έτσι θα αποφύγουμε εμπορικούς πολέμους. Οι διατλαντικές σχέσεις είναι κάτι παραπάνω από εμπορικές σχέσεις, οπότε αν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο για να εξασφαλίσουμε τα μηδέα μας συμφέροντα εμπορικά, έτσι θα μπορέσουμε να διασώσουμε και τις γενικότερες σχέσεις μας διατλαντικά. Εδώ στο σώμα αυτό προσβλέπουμε στη συνεργασία με το νέο Κογκρέσο σε ε, ισόρροπη βάση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πετροπέ, είναι πολύ σημαντικές οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εμπορικές και τώρα βρισκόμαστε σε εξαιρετικές καταστάσεις έχουμε να χάσουμε και δύο πλευρέ αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και από αυτό έχουν να χάσουν πολλοί. Γι' αυτό και είμαι θετικό για τι διαπραγματεύσει με τι ΗΠΑ και σα ευχαριστώ για τι προσπάθειε που κάνετε να το πετύχετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σαφή όσον αφορά τους δασμούς του Χάλιβα. Δεν δεχόμαστε όμως δασμούς στα αυτοκίνητα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τον Πρόεδρο Τραμπ. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα για τους δασμούς στο χάλιβα και για τους δασμούς στα αυτοκίνητα. Θέλουμε να μας ενημερώνει συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξελίξεις σε αυτή την τόσο σημαντική υπόθεση. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις μας με τις ΗΠΑ, ακόμη και αν είναι περιορισμένες οι διαπραγματεύσεις, γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ανησυχίες χωρίς λόγο. Ευχαριστούμε κύριο Μπατικόφερ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίρομαι που συζητούμε σήμερα το θέμα αυτό, διότι χρειάζεται προσοχή να μην λάβουμε εσφαλμένες κατευθύνσεις. Κανείς δεν έχει αντίρρηση να μειωθούν οι δασμοί. Νομίζω όμως ότι κυρία Μάλμστρομ η εντολή που προτείνεται δεν είναι ρεαλιστική. Οι Αμερικανοί δεν θέλουν να τηρήσουν τη συμφωνία που επέτυχε μαζί τους ο πρόεδρος Γιούνκερ και βλέπε Γεωργία. Τι γίνεται και με την συμβολή του εμπορίου για την βιώσιμη οικονομία και την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Τι γίνεται με την υπόσχεση Τραμπ ότι θα καταργήσει όλους τους εμπορικούς φραγμούς όταν βλέπουμε ότι αρνείται εξ αρχής να συζητήσει καν για τους κανόνες των δημόσιων ε, προμηθειών. Τι γίνεται με θέματα αμοιβαία αναγνώρισης προδιαγραφών και προτύπων. Φοβούμε κυρία Μάλμστρομ ότι αυτό που κάνετε περισσότερο παίζεται καθυστερήσεις σαν να κλωτσάτε το τενεκεδάκι όπως λένε στα αγγλικά. Ο κύριος Πρέτσελ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι ενδιαφέρον να ειδεί κανεί το γεγονός ότι ένας πρόεδρος Τραμπ που είναι συνομιλητής μας στις ΗΠΑ επηρεάζει την συζήτηση που γίνεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Εάν θυμηθώ με πιο ενθουσιασμό είχατε αντιμετωπίσει την TTIP παρόλο που προέβλεπε ε, τρομερά περιοριστικούς όρους, τότε εκπλήσωμε για τις επιφυλάξεις που ακούω τώρα πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Κυρίε και κύριοι, ο Ντόναλτ Τραμπ έκανε μια πρόταση απλή και ξεκάθαρη. Και επειδή όλοι εδώ είστε υπέρ της μείωσης των δασμών, είπε όλοι οι δασμοί να καταργηθούν. Αυτό είπε ο Τραμπ, να τους καταργήσουμε όλους. Εγώ βρίσκω ότι είναι μια επικοδομητική πρόταση, κυρία Μάλμστρεμ, που θα μπορούσατε έτσι να τη χρησιμοποιήσετε και να γίνει πάρα πολύ απλή διαπραγμάτευση με τον Τραμπ. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι χαόδηση η διακυβέρνηση η Τραμπ έχει αρχίσει εμπορικούς πολέμους, έχει αποσύρει τις ΗΠΑ Πολιτείες από τις συμφωνίες για το κλίμα και έχει πολύ στενές σχέση με τον Πούτιν. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσουμε την διατλαντική σχέση, διότι έχουμε και το Κογκρέσο και πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αυτό το καταστροφικό ρεύμα Τραμπ. Ελπίζω να μπορέσουμε να δούμε τι θα επιτύχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις Καταλήξαμε στο συμπέρασμα την τελευταία φορά ότι με τον Τραμπ να προσπαθεί κανείς να, να βγάλει άκρη είναι δύσκολο. Και για τη συμφωνία TTIP υπήρχαν σκανδαλώδεις ρήτρε. Και υπάρχουν και τα θέματα της ε, απορροής κεφαλαίων σε φορολογικούς παραδείσους. Πρέπει να κάνουμε ωστόσο προσπάθεια για να προχωρήσουμε. Διακόπτει ο πρόεδρο. Ε, ε, αντιμετωπίζουμε μεγάλη πίεση χρόνου, κυρία συνάδελφε. Σας παρακαλώ να σέβεστε πάντοτε τον χρόνο σας. Η Επίτροπος, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ναι, πράγματι έχουμε διαφορές με τους ε, Αμερικανού, με την Αμερικανική κυβέρνηση σε πολλού τομεί και βεβαίω και στον τομέα του εμπορίου. Αυτό που κάνουμε και αυτό που ήταν ο στόχος της συναντήσεως του Ιουλίου ήταν παρά τις διαφορές αυτές να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε μια κοινή ατζέντα, μια θετική πλατφόρμα στον χώρο του εμπορίου για να μπορέσουμε να αποφύγουμε περαιτέρω κλιμάκωση που θα ήταν κακή και για μας και για αυτούς αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό συμφωνήθηκε τον Ιούλιο και δημοσιεύθηκαν αμέσως τα όσα συμφωνήσαμε. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να δείξουμε σεβασμό στην ατζέντα ε, που συμφωνήθηκε τότε, τότε. και ακολουθούμε αυτό που ομόφωνα συνεπέρανε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνάντηση στη Σόφια πριν από ορισμένους μήνες και πρότεινε αυτά τα πράγματα ομόφωνα στους Αμερικανούς. Έξι μήνες διαπραγματευόμαστε με τους Αμερικανού Εγώ στα πολλές φορές σε απόλυτη διαφάνεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή ΙΝΤΑ. Η δε έκθεση για το τι συζητείτε σε όλου του τομεί βρίσκεται στην ιστοσελίδα μα από το πρωί και μπορείτε να την αναγνώσετε. Αυτό που ζητούμε από το Συμβούλιο είναι δύο εντολέ. Αφενό για conformity assessment, αξιολόγηση συμμόρφωση, και το άλλο για βιομηχανικά αγαθά. Βιομηχανικά αγαθά, όλα τα βιομηχανικά αγαθά μεταξύ αυτών και τα αυτοκίνητα και προϊόντα αλίας το ίδιο γίνεται και στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Μπαίνουν εκεί τα αγαθά αυτά, στο πλαίσιο αυτό. Αυτό είναι όλο και τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει τίποτε το κρυφό. Αυτό προτείνουμε. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Δεν πρόκειται για διαπραγματεύσεις ελεύθερου εμπορίου. Μια πλήρης FTA, Free Trade Agreement, θα, θα και όλα αυτά που λέτε. Δηλαδή δημόσιες προσφορές, γεωγραφικές ενδείξεις, άλλα θέματα δικά μας όπως η γεωργία. Αυτά τα πράγματα δεν περιλαμβάνονται. Και βεβαίως θα είχαμε ζητήσει τότε από ε, τον εταίρον μας να υπογράψει τη Συμφωνία των Παρισιών. Αλλά δεν πρόκειται για free trade agreement. Είναι περιορισμένη, ωστόσο αποφέρει ωφέλειες και σε εμά και σε αυτούς. Και μιλούμε για δισεκατομμύρια ευρώ εκατέρωθεν, εάν μειωθούν ή καταργηθούν οι δασμοί. Γι' αυτό και είναι σύντομη εντολή, γιατί περί αυτού και μόνο πρόκειται. Μόνο για τα θέματα αυτά. Είναι προφανές ότι η συμφωνία δεν θα μπορέσει να συναυθεί εάν δεν υπάρξει ε, λύση για αλουμίνιο και χάλιβα. Δηλαδή πρέπει να φύγουν οι δασμοί. Και δεν θα προχωρήσει επίσης εάν οι Αμερικανοί επιβάλλουν και, άλλες, και άλλους δασμούς όπως συζητείτε. Είναι και αυτό σαφές και απηχείται και στην, και στην ε, διαπραγματευτική εντολή. Και μιλώ πολύ σοβαρά. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο ε, θα είναι καλό, επικοδομητικό και για τις βιομηχανίες και για τους καταναλωτές και για τα δύο μέρη και υπόσχομαι ότι θα σας τηρώ ενήμερους και, ενήμερους, και ενήμερες συγγνώμη, για το που βαδίζουμε. Πάντως, ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν υπάρχει καμία κρυμμένη ατζέντα. Thank you, thank you for being... Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για αυτό το θέμα εδώ. Και περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση του κ. Φέντερλεϊ σχετικά με την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα νοτά του επίπεδου. Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά ως εισηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ δεν νομίζω να χρησιμοποιήσω όλο μου το χρόνο. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφου που συνεργάστηκαν μαζί μου προκειμένου να προχωρήσει αυτός ο κανονισμός που θέτει νέες προδιαγραφές και απλοποιεί τι διοικητικέ διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την χρήση του ονόματος τομέα του επίπεδου EU. Έχουμε μία στρατηγική και πιστεύουμε ότι θα ενισχυθεί με ε, το όνομα αυτό και έτσι θα υπάρχει μια πλατφόρμα EU που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και επιχειρήσεις αλλά και πολίτες ανεξάρτητα από το σε ποια χώρα κατοικούν να επιλέξουν ένα τομέα ανωτά του επίπεδου για το όνομα EU. Οι αγορές και η δυναμική του ψηφιακού τοπίου σίγουρα θα ενισχύσουν τη θέση μας. Η χρήση του ονόματος αυτού είναι πολύ σημαντικό για την ψηφιακή ταυτότητα το όνομα αυτό, το ψηφιακό, προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, σε πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση έτσι στο όνομα αυτό EU. Δεδομένου ότι μοιραζόμαστε και έχουμε κοινέ αξίες μεταξύ μας. Δέχτηκε την πρόταση της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο, αλλά θέλησε να προσθέσει κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, το σεβασμό του ιδιωτικού βίου ε, των χρηστών, την ασφάλεια, την προστασία των ε, δικαιωμάτων. Χαίρομαι που ενισχύσαμε το κείμενο όσον αφορά το κράτο δικαίου και τα δικαιώματα. Το Κοινοβούλιο επίση ήθελε καλύτερο έλεγχο στην, ε, στον καθορισμό των κριτηρίων και τα κριτήρια του Μητρώου και πώς θα λειτουργεί αυτό. Ελπίζουμε τις διαπραγματεύσει να διασφαλιστεί αυτό. Η Επιτροπή θέλει να καταργήσει τον περιορισμό ότι δηλαδή αυτά είναι μόνο για μη κυβερνητικέ οργανώσει και το έχει εγκρίνει αυτό το Κοινοβούλιο. Αυτό που μπορούμε να διασφαλίσουμε είναι η Επιτροπή να κάνει ενδεχομένως προτάσεις για αλλαγέ αν αποδειχτεί ότι χρειάζεται. Μπορούμε να ζητήσουμε, από, να ζητήσουμε δράσεις προκειμένου να αποφευθεί η καταχρηστική καταχώρηση με το όνομα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν προτείνει αλλαγές που κάνουν τη διαφορά και που αλλιώς δεν θα ήταν δυνατόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το προσωπικό, τους συνεργάτες μας που βοήθησαν πολύ στην επιτυχία αυτή. Είμαστε ενωμένοι μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων. Είχαμε έναν μόνο τριμερή διάλογο με τρία σημεία και το Κοινοβούλιο πέτυχε πάρα πολλές νίκες αυτών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Ε, Καλώ ήρθατε, κύριε Επίτροπε Γιούροβα. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτέ, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον Φρέντερικ ε, Φέντερλεϊ, καθώ και του ε, σκιώδει εισηγητέ για την πολιτική συμφωνία που έφτασαν στι 5 Δεκεμβρίου οι συνομοθέτε και ενέκριναν ενεκρίθηκε στις 14 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή Βιομηχανίας. στηρίζουμε τη συμφωνία και ολοκληρώνεται έτσι μία πολύ ταχεία διαδικασία από την υιοθέτηση της πρότασης της Κομισιόν για ένα κανονισμό ε, τον Απρίλιο του 2018 για το όνομα .eu. Η Συμφωνία των Συνομοθετών ενισχύει τον κανονισμό σε διάφορα σημαντικά θέματα. Κυρίως διευκρινίζει ότι το νομικό πλαίσιο για το, το όνομα .eu ε, σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές ε, που υπάρχουν στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και κυρίως την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης και την προστασία των καταναλωτών. Προβλέπει επιπλέον ασφαλιστικές δικλείδες κατά της καταχρηστικής ε, καταχώρησης του τομέα ονόματος e με μια αξιολόγηση για το πόσο για το πώς λειτουργεί το Μητρό ε, ως γραφείο ε, πνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Εφαρμόζεται γρήγορα έξι μήνες ε, μετά τη θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού με νέα κριτήρια επιλεξιμότητας που θα επιτρέπουν σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να καταχωρούνται στον τομέα .eu ανεξάρτητα με το που ζουν είτε εντός εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα ο τομέας .eu ε, ε, υπάρχει για 500 εκατομμύρια ανθρώπους και επιχειρήσεις στις 28 χώρες στην Ισλανδία, Λίχτενστάιν και Νορβηγία επιπλέον. Ο κοινό μας στόχος είναι να έχουμε ένα καλό μελλοντικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στο όνομα.eu να αναπτύσσεται, να δίνει τις καλύτερες δυνατές ε, υπηρεσίες στους πολίτες και στις ε, επιχειρήσεις. Ο συμβασμός που πέτυχαν οι συνομοθέτες ακριβώς βοηθάει στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Ευχαριστώ την Επίτροπο και τώρα οι ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες. Για δύο λεπτά ο κύριος Χακμάρκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία διαπραγμάτευσης και την τελική απόφαση. Είναι μικρό νομοθέτημα, αλλά σημαντικό για να αναπτύξουμε την ενιαία ψηφιακή αγορά. Ο νέος τομέας .eu ε, θα ενισχύσει την ε, ενωσιακή διαδικτυακή ταυτότητα, θα αυξήσει και θα πλουστεύσει το διασυνοριακό εμπόριο. Όμως, η αξιοπιστία του τομέα ε, Υγιού μπορεί να, τύχει, να πέσει θύμα εκείνων όσους, όσων θέλουν να ε, υποσκάψουν το δημοκρατικό μας σύστημα με κυβερνοεπιθέσεις που γίνονται σε όλα τα επίπεδα συνέχεια. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δούμε το, την ψηφιακή μας υποδομή, να τη θεωρήσουμε κρίσιμη υποδομή, που πρέπει να είναι ανθεκτική σε εξωτερικές πίεσεις και επιθέσεις. Οι νέοι κανόνες ε, λένε ότι όσοι καταχωρούν αυτόν τον τομέα καλή την πίστη, θα πρέπει μαζί με αυτούς που καταχωρούν τους ενδιαφερόμενους ε, να το κάνουν γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι ένα μικρό βήμα για την ενιαία ψηφιακή αγορά και σημαντικό όμως για την κυβερνοασφάλεια της Ευρώπης. Είναι βήμα προς σωστή κατεύθυνση ε, και είναι ένα βήμα μεταξύ πολλών άλλων. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών για δύο λεπτά ο κύριος Ζωρίνιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για να μπορέσουμε να παγιώσουμε τις αξίες μας που είναι κοινέ μεταξύ μας στην ψηφιακή αγορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει αυτή την ταυτότητα και να τη βασίσει σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους. Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε την ίση πρόσβαση στον εξοπλισμό και τρίτον, να σεβόμαστε τον ε, προσωπικό βίο, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Με αυτή την ονομασία .eu μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτό. Και λέω συγχαρητήρια σε όσους δούλεψαν προς αυτή την κατεύθυνση στον κύριο Φέντερλη, τον εισηγητή, τους σκιώδης ε, ε, εισηγητές, τον Μόναρ για παράδειγμα από τους σοσιαλιστές που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια αλλά και ευελιξία στην ονομασία αυτή. Συγχρόνως όμως πρέπει να πάμε και πιο μακριά. Με ένα δίκτυο πρόσβασης και κοινέ υπηρεσίες με μια συγκεκριμένη και μοναδική ταυτότητα, ταυτότητα όπως γίνεται με το Wi-Fi for You, μπορούμε να βοηθήσουμε με το στίγμα της Ευρώπης στον ψηφιακό χώρο οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι πιο κοντά ε, στο κόσμο και όσοι είναι περισσότερο δικτυωμένοι πρέπει να μπορέσουν να υποφεληθούν. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω κάποιες σημαντικές πτυχές του κανονισμού αυτού. Πρώτα απ' όλα διατηρείται η διαχείριση του ονόματος αυτού από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμό. Επιτρέπεται να καταγραφούν οι πολίτες ανεξάρτητα από το που κατοικούν επιτρέπεται ένα μητρό επιχειρήσεων που βρίσκονται είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μπορεί να γίνει καταγραφή και σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις αλφαβήτους. Οι χρήστες λοιπόν έχουν αυτήν την ευελιξία και επίσης υπάρχει και προστασία κατά της καταχρηστικής καταχώρησης. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνοψίζοντας, η ονομασία αυτή τομέα τελεία η αποτελεί μέρο της κληρονομιάς μας και είναι η δικιά μας η ψηφιακή κληρονομιά. Είναι αναγκαίο να υποστηρίζουμε την ονομασία αυτή και να φροντίσουμε για την επιτυχία της. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτό, κύριος Πακέτ. Η ονομασία αυτή έχει ένα στόχο, τον οποίο στηρίζω 100%. Την ενίσχυση της ψηφιακής μας ταυτότητας. Όμως η ονομασία αυτή πρέπει να έχει επιτυχία που τώρα δεν έχει. Ενώ από την άλλη μεριά είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι γνωστή σε ολόκληρο το κόσμο. Υπάρχουν περιθώρια πολλά βελτίωση λοιπόν. Ίσως να έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε υπερβολική γραφειοκρατία και διοικητικό άχθος για την ονομασία αυτή τελεία EU. Γιατί θέλουμε υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Ναι, συμφωνώ, αλλά μήπως πηγαίνουμε υπερβολικά μακριά με την ρύθμιση της ονομασίας αυτής. Και αυτό που με απασχολεί είναι και οι επιχειρήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Τι θα γίνει με τους Βρετανούς που θα έχουν αυτή την ονομασία. Δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να την έχουν. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να προσφέρουμε περισσότερη ευελιξία στο σύστημα της ονομασίας αυτής. Πρόεδρος, ένα λεπτό κύριο Ζάβορα. σημαντικό είναι το όνομα αυτό υψηλού επίπεδου για την ε, ελευθερία του λόγου και για τις επιχειρήσεις και γι' αυτό και πρέπει να ρυθμίζεται με στόχο ε, να υπάρχουν κοινέ ευρωπαϊκές αξίες και αυτές να υποστηρίζονται. Μέσω του κανονισμού δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ισορροπημένο σύνολο κανόνων για το πώς θα γίνεται η καταχώρηση των ε, EU domains στο μέλλον. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα δύσκολοι κύριοι μπροστά μας. Σε μια εποχή όπου πολλοί πιστεύουν σε εναλλακτικέ αλήθειε και αυτό συμβαίνει μάλιστα σε βιομηχανική κλίμακα, οι ιστοσελίδε που θα διατηρούν τις ευρωπαϊκές αξίες πρέπει να βρουν ασφαλέ λιμάνι στο ίδιο e domain και να συνεχίσουν να διαδίδουν τη γνώση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά η οποιαδήποτε προσπάθεια να υπονομευθεί, αυτή, να αυτός ε, ο τομέας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος, για ένα λεπτό η κυρία Λόπε Μπερμέζο. Θέλω να συγχαρώ τη δουλειά που έκανε ο εισηγητή για να φτάσει σε πλατιά συνένεση. Στις διαπραγματεύσεις ε, υπερασπιστήκαμε την ανάγκη να θεωρήσουμε αυτό το εργαλείο πέρα από την οικονομική του διάσταση, να δούμε και άλλα στοιχεία και να το δούμε μέσα σε ένα ε, πλαίσιο όπου και τα συμβολικά του χαρακτηριστικά έχουν μεγάλη σημασία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε σωστή χρήση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με βάση τις κοινέ αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα πρέπει να επωφεληθούν από αυτό το τομέα, πέρα από τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, και οι πολίτε, λοιπόν. Σημαίνει επίση ότι οι δημόσιε ρυθμιστικέ αρχέ θα εξασφαλίζουν ισορροπημένη και σωστή χρήση του τομέα στι διάφορε διαστάσει. Επίση, η ιδιωτική παρέμβαση και η διαχείριση του τομέα θα υπόκειται στου σωστού ελέγχου, κρατώντα την δημόσια διάσταση του τομέα αυτού. Υπάρχουν ε, και άλλε πτυχέ που θα πρέπει να συμπεριλάβει η συζήτηση αυτή, σαφώ πιο πολιτικέ. Για 1,5 λεπτό, η κυρία Λεσεβαλιέ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι καλές οι προθέσεις με την ονομασία αυτή για να αντιμετωπιστούν και οι καταχρήσεις και τα λοιπά. Υπάρχει μια ιδεολογική διάσταση. Θέλετε να ενισχύσετε στο πνεύμα των χρηστών μια ευρωπαϊκή διάσταση. Να προωθηθούν online οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολυγλωσία, ε, ασφάλεια, ε, εμπιστευτικότητα, αλλά και η δικιά σας άποψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι τελικά δικαιώματα κάθε μειονότητα. Και όσοι δεν συμφωνούν με τα δικά σας κριτήρια, θα τιμωρούνται, θα χάνουν την ε, διεύθυνση αυτή. Για να προστατευτεί, λέτε, το κράτος δικαίου. Οι χώρες που για σας δεν σέβονται το κράτος δικαίου θα υποβάλλονται σε κυρώσεις. Ουγγαρία, Πολωνία, Ιταλία, των οποίων η μεταναστευτική πολιτική επικρίνεται πολύ συχνά σε αυτό εδώ το σώμα. Υπάρχουν ελευθερίες μεταξύ άλλων και ελευθερία έκφρασης. Αδιαπραγμάτευτη. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα τέτοιο σχέδιο. Ευχαριστούμε. Επίτροπος Γιούροβα τώρα για να απαντήσει παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις θετικές σας παρατηρήσεις. Αυτό το τελικό κείμενο όχι μόνο εξυγχρονίζει το νομικό πλαίσιο του τελεία EU, αλλά προωθεί ε, σε επιγραμμικό επίπεδο το κράτος δικαίου και ενισχύει την προσέγγιση ε, του κατόχου με βάση τις απόψεις ε, και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε όλο και περισσότεροι άνθρωποι και επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τον τομέα .eu γιατί είναι σημαντικός τρόπος για να συμμετάσχουν στην ενιαία ψηφιακή αγορά και να διατρανώνουν την ευρωπαϊκή διαδικτυακή ταυτότητα. Περιμένω με υπομονησία την, το αποτέλεσμα της αυριανής συζη... Ε, ψηφοφορίας. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Και τώρα ο εισηγητής μας ξανά, ο κ. Φέντερλε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι τόσο συχνά, τόσο ενωμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Και όχι το λέω αυτό μόνο επειδή είμαι εγώ εισηγητή, αλλά και ο κύριο Όκμαρ και άλλοι σκιώδει ε, συμφωνούν. Οπότε όλοι προσβλέπουμε στην αυριανή ψηφοφορία που νομίζω ότι θα πάει καλά. Όπω και ο τριμερή διάλογο που κράτησε μία ώρα και 17 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν κυρία Επίτροπε και ευχαριστώ όλου του συναδέρφου σκιώδης κλπ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τι ωραία που είναι να ακούει κανεί ότι τα πράγματα πάνε ομαλά και εύκολα, που και που. Καλό είναι να το ακούμε. Ωραία, ολοκληρώθηκε η συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο. Και τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, που είναι η έκθεση Ρέιμον, ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού. Το λόγο έχει ο συγητής μας, ο κύριος Ρέμον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι εισηγητής για τον ανταγωνισμό. Και θα πρέπει να σας πω ότι το Κοινοβούλιο συνεργάστηκε με επικοδομητικό τρόπο και κινηθήκαμε προς την ίδια κατεύθυνση όλοι. Και εμείς με σας. Και αυτό μας ικανοποιεί η Κομισιόν ε, τεκμηρίωσε πολύ σωστά τις αποφάσεις της και χάρη σε αυτό το Κοινοβούλιο έφτασε σε πλατιά συνένεση μεταξύ των διαφορών πολιτικών ομάδων. Αυτό είναι ενδιαφέρον και παρατηρήθηκε σε τέσσερις τομείς. Την ενεργοποίηση του δικαιώματος ανταγωνισμού, την ε, ψηφιακή ανάπτυξη και το περιβάλλον και την τραπεζική οικονομία. το δίκαιο του ανταγωνισμού είναι ένα βασικό εργαλείο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουμε να προβληματιζόμαστε, ειδικά και το πώς εφαρμόζεται σε ψηφιακό επίπεδο. Ε, υπήρξε μεγάλη συνένεση εδώ μεταξύ των σκιωδών εισηγητών ότι θα πρέπει αυτός ο τομέας να αναπτυχθεί περαιτέρω. Ο ψηφιακός δηλαδή, ο ανταγωνισμός στο ψηφιακό τομέα. Οι επιχειρήσεις, οι ψηφιακές, συχνά προσφέρουν υπηρεσίες δωρεάν στους ε, χρήστες. Και συχνά όμως προσπαθούν να μονοπολίσουν την αγορά. Αυτό δεν σέβεται το δίκαιο ανταγωνισμού. Δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στα κέρδη και στο τζίρο θα πρέπει να αναπτύξουμε μια νέα λογική για τον ψηφιακό τομέα. Θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να τροποποιήσουμε το δίκαιο ανταγωνισμό, να το προσαρμόσουμε μάλλον στην ψηφιακή, στο ψηφιακό πλαίσιο. Ή αν θα πρέπει να έχουμε ένα χωριστό εργαλείο για να υπρασπιστούμε την αγορά από επιχειρήσεις που είναι υπερβολικά μεγάλες και μονοπωλιακές. Ορισμένοι ε, βουλευτές είναι πεπισμένοι για τη σημασία του κλίματος και έθεσαν την έμφαση στο περιβάλλον. Πράγματα τα οποία ασφαλώς και πρέπει να σκεφτούμε, αν δηλαδή θα αναπτύξουμε περαιτέρω τους μηχανισμούς αυτούς. Όπως είπα, ακόμη στην έκθεση αυτή, μάλλον έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει διάθεση των πολιτικών ομάδων να δραστηριοποιηθούν για το μέλλον. Η κυρία Επίτροπος έχει δραστηριοποιηθεί σημαντικά. Δυστυχώς είναι απούσα σήμερα. Γνωρίζω ότι ασθενεί. Όμως η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λειτουργεί μέχρι τώρα πραγματικά άριστα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Επίτροπο κυρία Γιούροβα. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι εξ ονόματος της συναδέλφου μου, θέλω να πω στον κύριο Ρεϊμόν και να ευχαριστήσω μάλλον τον εισηγητή κύριο Ρήμον... και τους ε, συνεισηγητές του. Ευχαρίστως θα μεταφέρω το θετικό σας μήνυμα στην συνάδελφό μου κυρία Βεστάγκερ για την θετική αξιολόγηση της συνεργασίας ε, μαζί της που κάνετε. Η έκθεση δείχνει για ποιο λόγο ο ανταγωνισμό βρίσκεται στο επίκεντρο τη πολιτική και θα αποτελέσει τμήμα των συζητήσεων και για τις επικείμενες ευρωεκλογέ. Όλοι συμμετέχουμε στην αγορά καθημερινά. Καταναλώνουμε. Θέλουμε να είμαστε πεπισμένες και πεπισμένοι ότι είναι έντιμες οι επιχειρήσεις απέναντί μας και θέλουμε να μεγαλώσουν, να μεγαλώνουν οι επιχειρήσεις μας, τα εργοστάσια μας και όχι να τα πετάμε έξω από την αγορά άλλοι με αθέμητες πρακτικές. Κρατώντας ανοιχτά στις αγορές μας, δίνουμε σε όλους την ευκαιρία να επιτύχουν. Και αυτό είναι άλλωστε και στην καρδιά της δημοκρατίας μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παίζει τον ρόλο της για να διασφαλίζει ώστε κάθε επιχείρηση να καταβάλει το ποσό φόρων που της αρμόζει. Οι ευρωπαϊκές ε, χώρες μέλη δεν μπορούν να δίνουν επιλεκτικά σε επιχειρήσεις φορολογικά πλεονεκτήματα που άλλε άλλες δεν λαμβάνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει 8 αποφάσεις για επιλεκτικά ε, φορολογικά πλεονεκτήματα πολυεθνικών και μιλούμε για πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ και πάνω από 40 επιχειρήσεις οι πολλές από τις οποίες είναι ευρωπαϊκές. Τούτο το μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασίες για τις φορολογικές ρυθμίσεις της εταιρείας Nike στις ε, κάτω χώρες. Θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή για να μεταρρυθμιστεί το πλαίσιο Φορολογία επιχειρήσεων ώστε να γίνει πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό. Μόνο η βελτιωμένη φορολογική νομοθεσία θα κλείσει τα παράθυρα που ανοίγονται για όλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλογίζεται και το ψηφιακό μας μέλλον. Τότε το μήνα η ε, Επίτροπος Βεστάγερ διεύθυνε συνεδρίαση για θέματα ανταγωνισμού. Μίλησαν για τον ψηφιακό κόσμο και τι σημαίνει αυτό για τον ανταγωνισμό. Στην διάσκεψη και στις πάνω από 100 ε, γραπτές ε, παρεμβάσεις είδε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ορισμένα θέματα επανέρχονται. Πρόσβαση στα δεδομένα, απειλέ κατά του ανταγωνισμού από μεγάλες επιχειρήσεις κατά νεοφιών επιχειρήσεων και μια αναστάτωση που προκαλεί κόστο σε άλλου. Και οι επιχειρήσει οι οποίε χρησιμοποιούν και τις πλατφόρμες τους και δεν επιτρέπουν σε ανταγωνιστές να ανταγωνίζεται στη βάση των ίδιων πλατφορμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβληματίζεται σοβαρά για όλα τα θέματα αυτά, διότι εάν αποτύχει ο ανταγωνισμός θα αυξηθούν οι τιμές, θα μειωθεί η ποιότητα και χάνουμε τότε αυτήν την θεμελιώδη υπόσχεση του ψηφιακού κόσμου ότι η τεχνολογία της αύριο θα είναι καλύτερη από αυτήν της σήμερον. Η έκθεσή σας σημειώνει ότι οι αγορές θα πρέπει και αυτές να λάβουν υπόψη τις ανάγκες του περιβάλλοντος. Συμφωνούμε. Η απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απορρίψει την συγχω... μάλλον ε, να δεχθεί την συγχώνευση Bayer Monsanto λήφθη μόνο όταν δεσμεύτηκαν οι δύο επιχειρήσεις να δώσουν ορισμένα τμήματα της παραγωγής τους όπως τα φυτοφάρμακα σε άλλο ανταγωνιστή. Ο ανταγωνισμός οδηγεί τις επιχειρήσεις να θέτουν στην αγορά νέα ασφαλέστερα προϊόντα. Μέσα στα πλαίσια των συνθήκων θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε υπέρ του κλίματος και του περιβάλλοντος. Όπως λέει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ανοιχτό πνεύμα και ο ελεύθερος ανταγωνισμός ωφελούν όλη την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Χρειαζόμαστε τους Ευρωπαίους πρωταθλητές, αλλά που να είναι οι σωστοί επιχειρήσεις οι οποίες να ανταγωνίζονται μεταξύ των και να στέφονται πρωταθλητές επειδή τους τις προτιμούν οι καταναλωτές. Αυτό θα ωφελήσει και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και τις άλλες επιχειρήσεις, δηλαδή μικρές και μεσές επιχειρήσεις που είναι και κουκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Βεβαίως και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Για κάθε μια επιχείρηση που θέλει να κάνει μια συγχώνευση υπάρχουν πολλές βιομηχανίες που αγοράζουν τα προϊόντα τους όπως χάλιβας και τσιμέντο. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές βασίζονται στον ανταγωνισμό ώστε να έχουν δίκαιους όρους στις αγορές που κάνουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Θα κάνουμε και HDI τώρα, εάν επιθυμούν οι συνάδελφοι να αγορεύσουν και δίνω το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Ζάινφελτ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι μια καλή έκθεση αυτή. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποιες σημαντικές της πτυχές. Πρώτον, οι επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών στον ψηφιακό κλάδο αντιμετωπίζουν συχνά αθέμητο ανταγωνισμό από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγοράζονται δηλαδή ευρωπαϊκές εταιρίες από μη ευρωπαϊκές εταιρίες. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τη δημόσια ασφάλεια. Ένα δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω εδώ είναι οι μεταφορές. Έχουμε δει δράσεις που περιορίζουν τον ε, ανταγωνισμό όχι μόνο μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ χωρών εξαιτία της μεταφοράς των επιχειρήσεων. Έπειτα, εμείς έχουμε γραφειοκρατία η οποία δυσκολεύει τον ανταγωνισμό από πλευρά των πιο μικρών επιχειρήσεων.